Εντάξει αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, άρχεται εκ νέου η συνεδρίασή μας και περνάμε στο σημείο της ημερήσια διάταξη υπαριθμών 10. Χαίρομαι που για αυτό το σημείο της ημερήσια διάταξη έχουμε τη νέα Επίτροπο για το Διεθνές Εμπόριο, την κυρία Σεσίλια Μάλμστρεμ ανάμεσά μας. Για πρώτη φορά μετά τον διορισμό ε, σε αυτό το αξίωμα έρχεται στην δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή, προσέρχεται. Χαίρομαι επίσης για το ότι αυτή η συνάντηση καταφέραμε να συντονιστεί σε αυτή τη χρονική στιγμή και μάλιστα για την πρωτοβουλία για την διαφάνεια όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις TTIP για τις επενδύσεις και το εμπόριο με τις ΗΠΑ και χαιρετίζουμε το ότι τεχνικά θα μπορέσουν ίσως αυτά γοργά να διευθετηθούν και από πλευρά Ευρωκοινοβουλίου να μπορέσει να επιτευχθεί και μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και στους πολίτες να καταδείξουμε ότι η συζήτηση έχει ορθολογικά θεμέλια πλέον περισσότερο από ό,τι κατά το παρελθόν. Αλλά οπωσδήποτε κύριε Επίτροπε θα μας πείτε και δύο λόγια για την περαιτέρω εξέλιξη των προτεραιοτήτων της πολιτικής εμπορίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν για τα όσα θα μας πείτε στην εισήγησή σας. Πρωτού ξεκινήσουμε όμως, δεν θέλω να αμελήσω να αναφερθώ και στον Υπουργό για το εμπόριο από τη χώρα του Ισημερινού, το Εκουαδόρ. Τον καλοχαιρετίζω ανάμεσά μας, που κάθεται εκεί ακριβώς απέναντί μου. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ του Ισημερινού και χαίρομαι που στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή τη θεωρείτε τόσο ενδιαφέρουσα ώστε να αξίζει την επίσκεψή σας. Και τώρα δίνω στην κυρία Μάνστρομ τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι η πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται να σας συναντήσω υπό την ιδιότητά μου μετά την ακρόαση και πραγματικά προσβλέπω στη μελλοντική μας συνεργασία. Η στιγμή αυτή είναι πολύ σημαντική, η πρώτη μας συνάντηση. Πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε την επόμενη πενταετία και πολλά θα προχωρήσουμε με επιτυχία ελπίζω στα κοινά θέματα που σας απασχολούν. Η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου και η Επιτροπή Εμπορίου είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίως έχουμε τη σχέση μας με το Συμβούλιο αλλά και με τους πολίτες. Από κοινού έχουμε την ευθύνη οι σχέσεις αυτές να φροντίσουμε να λειτουργήσουν γιατί έχουν σημασία. Το εμπόριο είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. 30 εκατομμύρια ε, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δουλεύουν για την, ε, στις υψηλό, υψηλόμιστες θέσεις που στηρίζουν τις εξαγωγές. Και αυτό είναι 10% του, του πληθυσμού μας και θέλουμε να αυξηθούν. Πολλά εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται σε επιχειρήσεις που, εργάζονται, που εξαρτώνται από το εμπόριο για τις ε, προμήθειές τους. Το εμπόριο, όπως γνωρίζετε επίσης, μας συνδέει με τον κόσμο. Ο Μάρκο Πόλο ταξίδεψε στην Ασία πάνω σε άλογα και μετέφερε ιδέες. Το ίδιο γίνεται σήμερα με τα εμπορικά πλοία αλλά και τις οπτικές ίνες. Λοιπόν, η σχέση αυτή δυναμώνεται από εμά και είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να μεταδοθούν αξίες και να προσεγγίσουν μεταξύ τους οι άνθρωποι. 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε χώρες όπου η, Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος. Και όλα αυτά έχουν σχέση με το εμπόριο. Έχουμε λοιπόν καθήκον να συνεργαστούμε και να εξασφαλίσουμε ότι θα υποφεληθούμε, θα δρέψουμε τα ωφέλη από αυτό. Βεβαίως δεν συμφωνούμε πάντοτε, αυτό είναι φυσιολογικό. Και γνωρίζω το σώμα σας για λίγο. Προσβλέπω όμως σε μια επικοδομητική συνεργασία και ελπίζω όπως είπε και ο Χάμφρι Γκόγκαρτ ότι τώρα είναι η αρχή μιας ωραίας σχέσης. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να πω μερικά πράγματα επί τριών θεμάτων. Η συνεργασία, δεύτερον για κάποια θέματα που είναι επιτάπητος και τρίτον για το πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Ξεκινώντας από τη συνεργασία. Η συνεργασία απαιτά, απαιτεί να ακούμε. Αυτό θα αποτελέσει την προτεραιότητά μου τον επόμενο μήνα και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Όλο και περισσότερο ασχολούμαι με το να ακούω τους πολιτικούς, τις μη κυβερνικές οργανώσεις, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τους διάφορους εμπλεκόμενους, ώστε να καταλάβω το πλήρες φάσμα των απόψεων για όλα τα θέματα. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι κατόπιν πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν σταθερότερο διάλογο. Διάλογο με εσά, πολύ σημαντικό, αλλά και με πολλούς άλλους εμπλεκόμενους. Ένας καλός διάλογος και συνεργασία απαιτεί διαφάνεια. Σας υπόσχέθηκα κατά την ακρόασή μου θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να αυξηθεί η διαφάνεια σε θέματα ε, διαπραγματεύσεων της TTIP. Και άρχισα αυτή τη δέσμευσή μου να την υλοποιώ. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε και σας υπέβαλε ε, κάποια νέα σημαντικά βήματα. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύει περισσότερες από τις προτάσεις που έχουμε προτείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη διαφόρων κεφαλαίων και όλοι θα μπορούν να τις μελετήσουν. Επιπλέον, και αυτό είναι σημαντικό για τη συνεργασία μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε, ε, ε, έχουμε σταματήσει να ε, ανταλλάσσουμε τα έγγραφα που αφορούν τη TTIP με λίγα μέλη. Όλα τα 750 μέλη θα έχουν τη δυνατότητα και θα είναι ε, ε, περιορισμένης διανομής πολύ λιγότερα. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο όταν βρίσκουμε τρόπο ότι να εξασφαλίσουμε ότι αυτά που πρέπει να μείνουν εμπιστευτικά θα μείνουν. Και οι υπηρεσίε μου είναι ήδη σε επαφή με τι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου για να εξασφαλιστεί κάτι τέτοιο. Βεβαίω θα υπάρξουν έγγραφα που δεν θα είναι δημόσια. Γνωρίζετε ότι μερικές φορές σε κάποια διαπραγμάτευση πρέπει κανείς να μένει σε ένα δωμάτιο χωρίς κάμερες οι διαπραγματεύσεις ε, για την ειρήνη, για θέματα εργασίας και για το εμπόριο. Χρειάζεται εμπιστευτικότητα μερικές φορές ώστε να επιτευχθούν σωστά αποτελέσματα. Ελπίζω ότι αυτό θα το κατανοήσετε. Ελπίζω όμως ότι τα πρώτα αυτά βήματα θα τα εκτιμήσετε και θα μας επιτρέψετε να δείξουμε στον κόσμο τι ακριβώς συζητείτε, τι ακριβώς προτείνετε και τι ακριβώς δεν προτείνετε, τι ακριβώς προτείνουμε και τι δεν προτείνουμε, έτσι ώστε να διαλυθούν οι παρεξηγήσει, οι μύθοι και να προχωρήσουμε από εκεί, ώστε οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι, οι πολίτες, οι μικρές επιχειρήσεις να ξέρουν τι ε, πρόκειται να ε, συμβεί. Οπότε έρχομαι στο δεύτερο σημείο. Τα θέματα που είναι επιτάπητος. Η που είναι φυσικά το πιο σημαντικό και το μεγαλύτερο θέμα που μας απασχολεί τώρα. Όπως είπα και κατά την ακροασή μου, θέλουμε να κάνουμε μια νέα αρχή στις διαπραγματεύσεις αυτές. Η πρωτοβουλία διαφάνειας είναι ένα σημαντικό κομμάτι της νέας αυτής αρχής. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι να εμπλακούμε περισσότερο στη συζήτηση, όχι μόνο δημοσιεύοντας άρθρα στην εφημερίδα, αλλά μιλώντας με την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις της. Με τη συμμετοχή σε πολλές συναντήσεις και εδώ και εκτός Ευρώπης αυτό θα συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο. Και επίσης πρέπει να αυξηθεί η δέσμευσή μας, ε, η ενασχόλησή μας με ε, συζητήσεις στο διαδίκτυο. Χρειάζεται ε, βεβαίως όλα αυτά, χρειάζεται ισορροπία, αλλά χρειάζεται και ρεαλισμό. Στην, την Κυριακή θα πάω στη Ουάσιγκτον για να συζητήσω τα θέματα με τον, ε, με τον πρέσβη κύριο Φλόμαν. Και βεβαίως θα δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Και θα ήθελα να σας ε, ε, παρουσιάσω κάποιες σκέψεις για μια φιλόδοξη και ρεαλιστική TTIP φιλόδοξο αποτέλεσμα όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά για τα προϊόντα, τις ε, υπηρεσίες και τις ε, κρατικές προμήθειες. Πρέπει να στραφούμε προς τον Καναδά. Υπάρχει, ε, θα πρέπει να επιτρέψουμε τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες να ανταγωνίζονται ισοδύναμα σε μια πραγματικά διατλαντική αγορά και θα εργαστούμε για μια νέα πρόσβαση στην αγορά των υπηρεσιών. Επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι δεν θα καλυφθεί. Ούτε οι δημόσιες υπηρεσίες, ούτε οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Αυτό είναι σαφές. Ο δεύτερος πυλώνας της TTIP είναι οι ρυθμίσεις. Θέλω ένα πακέτο που να λειτουργεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και που θα ενισχυθεί, όχι να αποδυναμώνει το επίπεδο προστασίας στην Ευρώπη. Να περιλαμβάνει τρόπους να ενθαρρύνονται οι αρχές της Ευρώπης και των ΗΠΑ να συνομιλούν μεταξύ τους Καθώ καθώς θα διπλουθούν οι κανόνες που θα επηρεάσουν τη διατλαντική σχέση ευθύ εξ αρχής, από την αρχή της συνεργασίας και ελπίζουμε ότι θα αναπτυχθούν κανόνες όχι μόνο μεταξύ μας αλλά και διεθνώς. Θα συμπεριληφθούν συμφωνίες για την ε, μειωμένη εφαρμογή των ε, ρυθμίσεων σε αφορά τα αυτοκίνητα, τα εργαλεία, τον εξοπλισμό, κάποια ε, κάποιες συσκευές. Ας πούμε για τα αυτοκίνητα μπορούμε να δούμε τις διαφορές, τις διάφορες δοκιμές συγκρούσεων των αυτοκινήτων και τα διαφορετικά συστήματα. Η, η προσέγγιση διαφόρων διαφορών χωρίς να ε, διακινδυνευτεί ασφάλεια μπορεί να σημαίνει πολλά. Και επίσης τα διάφορες δοκιμές και τα πρότυπα που δημιουργούν ε, ε, ανώφελες ή περιτές διαδικασίες. Επίσης, οι διαδικασίες συμμόρφωσης στο, στα τελωνία κλπ. Υπάρχει απεριτή γραφειοκρατία. Επίσης, μονοφυριδική πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες και αυτό είναι βασικό και όχι μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που, είναι το 30% των εξαγω... που κάνουν το 30% των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Ο τρίτος πυλώνας της ρεαλιστικής TTIP θα καλύπτει κανόνες που θα έχουν παγκόσμια ε, επίδραση, ας πούμε, για την ενέργεια και τους πρώτες ύλες. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε πρόσβαση στις ενεργειακές πηγές των ΗΠΑ και να μας ανοίξει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας με τρόπο που να, γίνεται, ε, να έχει σεβασμό το περιβάλλον. Επίσης, οι γεωγραφικές ενδείξεις σε τρόφιμα, ε, στην, ε, η Absolute Vodka και φάρμακα. Όλα αυτά θα είναι ιστορικές συμβιβασμοί γιατί πάντοτε η ε, προσέγγιση των ΗΠΑ ήταν διαφορετική. Και βεβαίως ε, θα υπάρχει και ένας ρόλος ε, που θα επιτρέπει στην κοινωνία των πολιτών να, κάνει, να παρακολουθεί τα θέματα. ένα άλλο τομέας είναι οι επενδύσει Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα η Κομισιόν θα δημοσίευσει την ανάλυση μας ε, στις απαντήσεις αυτής της ε, θερινής δημοσίας διαβούλευσης για την προστασία των επενδυτών. Τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους θα συζητήσω μαζί σας εδώ, ελπίζω, και με τους Υπουργούς Εμπορίου για το τι πορεία θα ακολουθήσουμε. Έτσι ελπίζουμε ότι την Άνοιξη θα έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για αυτό το δύσκολο ζήτημα. Εάν συνεργαστούμε, με βέβαιο ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Και σίγουρα θα είναι πολύ σημαντικό το επίτευγμα αυτό. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Έχουμε και άλλα να κάνουμε εκτός από το TTIP. Ε, να σας επισημάνω ορισμένα. Η Ιαπωνία είναι η δεύτερη σημαντικότερη διαπραγμάτευση, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και έχει τεράστιες δυνατότητες να ανοίξει προς τους εξαγωγείς και τους επενδυτές μας. Εδώ χρειαζόμαστε μια φιλόδοξη συμφωνία που θα διευκολύνει πραγματικά το εμπόριο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς, αντιμετωπίζοντας τα θέματα των δασμών, των αριθμιστικών πολιτικών, των δημοσίων συμβάσεων και των γεωγραφικών ενδείξεων. Για να επιτευχθούν όλα αυτά Φυσικά η ουσία είναι σημαντικότερη από την ταχύτητα, αλλά υπάρχει περίπτωση να ολοκληρωθεί η συμφωνία αυτή και να συναυθεί μέσα στο επόμενο έτος εάν η Ιαπωνία συμφωνήσει με τις φιλοδοξίες μας και αυτό θα είναι καλό για τους καταναλωτές και για τους εργαζομένους και οι διαπραγματεύσεις με το Βιετνάμ είναι σημαντικές μεγάλη οικονομία, 90 εκατομμύρια άνθρωποι ε, πολύ συνδεδεμένη, διασυνδεδεμένη με την οικονομία της Ανατολικής Ασίας. Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν καλά και η κυβέρνηση του Βιετνάμ είναι διατεθειμένη να συνάψει συμφωνία στις αρχές του επόμενου έτους. Αυτό μπορεί να γίνει εφόσον προσφέρει περισσότερα το Βιετνάμ σε τομείς όπως οι υπηρεσίες, οι επενδύσεις, οι δημόσιες συμβάσεις, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι γεωγραφικές ενδείξεις, κάποιοι κανόνες ανταγωνισμού και οι δασμοί. Τέλος, έχουμε και την ευκαιρία να σημειώσουμε πρόοδο στο γύρο της Δόχα να τον ολοκληρώσουμε μάλιστα. Ε, τώρα πια δεν έχουμε τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζαμε στον ΠΟΕ. Η διαδικασία συνεχίζεται και την περασμένη εβδομάδα συμφώνησαν στον ΠΟΕ να προχωρήσει νέα συμφωνία για τη διευκολύνση του εμπορίου. Σημαντικό βήμα που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε τις υπόλοιπε ε, διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη καθυστερήσει αρκετά. Επίσης πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε επιτέλους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε το γύρο της ΔΟΧΑ παρότι έχουν περάσει 13 χρόνια από την έναρξή του, 13 ε, χρόνια που σημάδεψαν την παγκόσμια οικονομία δραματικά σε πολλές ε, χώρες, ε, εταιρείε, σε αναδυόμενες χώρες, σε αναδυόμενες οικονομίες, πολλές εταιρείε είναι τόσο ανταγωνιστικές όσο αμερικανικές, όχι περισσότερο. Στη Γεωργία έχουμε μεταρρυθμίσει τις πολιτικές μας με ελάχιστη και Κάποιε αναδιόμενες οικονομίες στο μεταξύ υποφελούνται από αυτό το νέο άνοιγμα και επεκτείνουν την παραγωγή τους. Άλλες όπως η Ινδία, έχουν σήμερα τόσο μεγάλη ανάπτυξη που τώρα πλέον έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν τα δικά τους προγράμματα επιχορηγήσεων. Η προσέγγιση λοιπόν της Ευρώπης ήταν πολύ σαφής. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη, ειδικότερα για τις φτωχότερε χώρε. Αλλά θέλουμε και ίσου όρου ανταγωνισμού οι εταιρείε πρέπει να ανταγωνίζονται με επίση επίσης με τους ομολόγους τους ε, σε τρίτες χώρες. Είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε το μερίδιο. Όπως ξέρετε, οι πιο φτωχές χώρες έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην ενιαία αγορά από την αρχή του γύρου το 2001. Αλλά πρέπει να φροντίσουμε επίσης οι εταίροι μας να δείχνουν και αυτοί ε, κάποια ε, ηγετικά ε, καθήκοντα πολλοί άνθρωποι έχουν βγει από τη φτώχεια λόγω του ανοίγματο των αγορών τη Ευρώπη και τη Αμερική και που έχει βασιστεί στο πνεύμα ηγεσία που έχουμε δείξει στον ΠΟΕ. Οι χώρε αυτέ σήμερα πρέπει να αντιληφθούν ότι η νέα του αυτή δύναμη του ε, αποδίδει επίση και ευθύνε ηγεσία παρόμοιου επίπεδου. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώ θα επιτύχουμε συμφωνία για να σημειωθεί η πρόοδο και να υποστηρίξουμε ε, το Γενικό Διευθυντή στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Εγώ θα προετοιμάσω ότι ε, έργο ε, ώστε να δούμε τι, πώς ακριβώς μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα. Αυτό με φέρνει στο τελευταίο μου σημείο. Τι γίνεται στο μέλλον, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Πρέπει να δράσουμε στρατηγικά. Πού θέλουμε να βρισκόμαστε, πού θέλουμε να βρίσκεται η Ευρώπη όταν εγώ θα φύγω από τη θέση μου Πώ μπορεί η εμπορική πολιτική να συμβάλλει στην υποστήριξη τη ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της παγκόσμιας ε, ολοκλήρωσης ε, στις ε, φτωχότερε αγορές, πώς μπορεί να ανταποκριθεί στι ανάγκε των πολιτών μα πώ μπορούμε να παρέχουμε μεγαλύτερε επενδύσει και ανάπτυξη μέσω του εμπορίου, πώ αντιμετωπίζουμε τι εμπορικέ σχέσει με τι αναδυόμενε χώρε και πώ συμφιλιώνουμε όλε τι διμερεί συμφωνίε με την προτίμησή μας για ανοιχτούς πολυμέρειες κανόνες. Πώς δημιουργούμε ευκαιρίες συντονίζοντας το τα διεθνή κανονιστικά καθεστώτα, προστατεύοντας ταυτόχρονα τους πολίτες μας. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Πρέπει επίσης να ορίσουμε προτεραιότητες. Δεν μπορούμε τώρα να φανταστούμε τις απαντήσεις για αυτές τις ερωτήσεις. Μέσα στους επόμενους μήνες θα δω πώς μπορούμε να μεταφράσουμε την εντολή του κυρίου Γιούνκερ σε έργα, σε μια νέα εμπορική πολιτική και θα παρουσιάσω σε μια ανακοίνωση τις απόψεις αυτές μέσα στο επόμενο έτος και θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις. Ελπίζω να μπορέσετε να συμβάλλετε σε αυτή την ανακοίνωση και εσείς όπως και τα κράτη-μέλη και η κοινωνία των πολιτών ώστε να τα γράψουμε τα πράγματα σωστά και να συζητήσουμε με συμμετοχή όλων, γιατί μπορούμε να εξυπηρετήσουμε την πολυμορφία των ευρωπαϊκών λαών μόνο εάν λάβουμε αυτές τις αποφάσεις μαζί. Προσδοκώ λοιπόν ε, για μια, να έχουμε μια όμορφη φιλία, να κάνουμε πολλές συζητήσεις σε πολυμερές και σε διμερές επίπεδο και ευχαριστώ φυσικά να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις σας. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά κύριε Επίτροπε. Τώρα καταρχήν στις κοινοβουλευτικές ομάδες θα δώσω τον λόγο σε ένα πρώτο γύρο και μετά στη συνέχεια εσάς κυρία Επίτροπε θα σας δώσω τη δυνατότητα να απαντήσετε στις παρεμβάσεις. Και έχω και μια ολόκληρη σειρά ευρωβουλευτών που ζήτησαν να παρέμβουν, αλλά σε ένα δεύτερο γύρο θα καλύψουμε τις παρεμβάσεις τους. Καταρχήν λοιπόν έτσι το ΕΛΚ θα λάβει τον λόγο πρώτο. Ο κύριος Κασπάρη έχει αρρωστήσει δυστυχώς. Ο κύριος Φιένερ θα θέσει την ερώτηση. Παρακαλώ θα το αντικαταστήσει. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε καλώς ήρθατε και εξ ονόματος του ΕΛΚ και θα έλεγα εξ όλων των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μας το λέγω. Καλώς ήρθατε. Προσβλέπουμε σε μια θετική συνεργασία μαζί σας στο μέλλον. Αλλά καλή και έντιμη και ακέραια. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα από καιρούς καιρών σίγουρα. Νομίζω μιλώ εξ όλων όταν σας λέγω ότι καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία σας για τη διαφάνεια. Πολύ σημαντική αυτή. Αλλά πρέπει να είναι και αποτελεσματική αυτή, να αποκτήσει σάρκα και οστά. Γιατί αυτό μετρά στο τέλος τέλος, το χειροπιαστό αποτέλεσμα. Επιπλέον δύο πράγματα είναι που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά που πρέπει να λάβετε υπόψη και θα ήθελα να σχολιάσετε. Πρώτο, το θέμα για την αξιοπιστία πώς θα δημιουργηθεί περισσότερη αξιοπιστία όσον αφορά τον ρόλο της ε, Ευρώπης ε, για, ως διαμεσολαβητού σε αυτές τις συμφωνίες, αλλά επίσης και την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής εμπορίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ένα όλο και μεγαλύτερο βαθμό αναλώνουμε χρόνο ως ε, εξετάζοντας κάποια θέματα αμυντικά. Δηλαδή ανησυχούμε περισσότερο και συζητούμε για τα αμυντικά θέματα πώς θα μπορούσαν να καλυφθούν και να αντιμετωπιστούν στις διαπραγματεύσεις. Όμως ο ρόλος μας στις διαπραγματεύσεις δεν είναι ποτέ λόγω αυτών των, αυτής της τάσης. Πρέπει πιο επιθετικά να μπορέσουμε να δράσουμε για να είμαστε επιτυχείς να μπορέσουμε να μεταθέσουμε το κέντρο βάρους όχι μόνο της πολιτικής εμπορίου αλλά και της συζήτησης και εδώ και στους πολίτες για μια πρωτοβουλία πιο επιθετική για τις δημόσιες προμήθειες ε, και αγορές και οποιοδήποτε άλλο θέμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να μετατρέψουμε το ρόλο μας πιο επιθετικά. Δεύτερον, για την αξιοπιστία να είμαστε ηγέτες στον ρόλο μας ε, ως ε, διαπραγματευτές και Έρχομαι από μια ομάδα όπου εξετάστηκε η ομάδα ε, από την επιτήρησή μας, την εποπτεία μας με για τη συμφωνία με τον Καναδά. Και βλέπουμε ότι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πήρε για μας για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε αυτή τη συμφωνία με τον Καναδά. Πέντε χρόνια, πέντε, εφτά ίσως κιόλα χρόνια για να μπορέσει να αποκτήσει σάρκα και οστά αυτή η συμφωνία. Αυτό είναι λοιπόν ε, το πρόβλημα για τους διαπραγματευτές. Μήπως ε, όταν θεωρούν ότι μπορεί να δώσει αποτελέσματα η πολιτική για το εμπόριο, αλλά μόνο μετά από 5 ή 7 χρόνια. Ε, αυτό πραγματικά υπονομεύει την αξιοπιστία μιας εμπορικής αποτελεσματικής πολιτικής και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Αλλά αν παίρνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να έχουμε μια σφαιρική συμφωνία με μια εντολή όπως εκείνη για τον Καναδά, για φανταστείτε πόσο χρόνο θα, πάρει, α, θα πάρουν άλλες συμφωνίες. Για να μην σκεφτούμε καν για την συμφωνία με τη ΣΥΠΑ το πόσο χρόνο θα απαιτούσε. Εσείς πιστεύετε ότι το χρονοδιάγραμμα το οποίο παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χρονοορίζοντας είναι ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα δεδομένου του πόσο καιρό χρειάστηκε για τον Καναδά. Και εσείς Επίτροπε τι μπορείτε να κάνετε για να επιταχύνετε τις διαδικασίες. Να αποδείξουμε στους πολίτες όχι μόνο ότι είμαστε ικανοί αλλά και ικανοί έγκαιρα να δώσουμε αποτελέσματα για μια τέτοια ευρεία σφαιρική συμφωνία. Για τους σοσιαλδημοκράτες παρακαλώ εσείς έχετε David τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δυστυχώς, Επίτροπε, φυσικά θέλω και εγώ να σας... Ε, συγχωρείτε. Ε, κυρία Επίτροπε, με χαρά σας υποδεχόμαστε. Θα έχουμε συνεργασία. Ε, θα είναι συγκρουσιακή και δημιουργική συνεργασία μας. Θέλω να αρχίσω με το μέλλον της εμπορικής πολιτικής. Όταν θα έχετε κάνει τις δικές σας σκέψεις και θα τις έχετε είτε γράψει είτε σκεφτεί ακριβώς ε, πώς θα είναι, μπορούσατε να επανέλθετε στην Επιτροπή μας για να συζητήσουμε, να δούμε πού θα συμφωνήσουμε, πού θα αλλάξετε ή πού εμείς ίσως θα αλλάξουμε ιδέα. Νομίζω ότι από κοινού πρέπει να καθορίσουμε πού θέλουμε να πάμε το επόμενο πενταετία, γιατί πρέπει να συνεργαστούμε, ε, αλλιώς θα είναι πιο κουραστική δουλειά και για τους δυο μας. Δεν θα μιλήσω για την, την διαφάνεια, πολύ, θα το κάνω αυτό. Θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω για την ε, προόδο για τη, στον τομέα της διαφάνειας και για δύο θέματα. Την ε, Σιγκαπούρη και το GSP+. Όσον αφορά τη Σιγκαπούρη, υπάρχουν φήμες, δεν ξέρω από πού προέρχονται, αλλά εν πάση περιπτώσει για να του αναφέρει ο τύπος κάτι θα συμβαίνει, ότι ενδεχομένως να αλλάξει άποψη ε, η Επιτροπή για την ε, προσφυγή κατά της ε, Σιγκαπούρης στα δικαστήρια. Ισχύει αυτό ότι δεν θα πάρετε, θα πάρετε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σχετικά επίσης με τη Σιγκαπούρη και αυτό το γνωρίζω από προηγούμενες συνομιλίες ότι εδώ δεν διαφωνούμε θα το ξαναδοκιμάσω όμως. Η συμφωνία με για τα προϊόντα και υπηρεσίες με τη Σιγκαπούρη είχε, είχε γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωριστή σε σχέση με τα με τις επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι πιο αμφιλεγόμενο θέμα από τα υπόλοιπα. Πάρα πολύ νωρίς στην θητεία σας θα μπορούσατε να πετύχετε ξεχωρίζοντας αυτά τα δύο και να περάσει η Σιγκαπούρη από το Κοινοβούλιο. Να μην γίνονται ε, συμβιβασμοί στο ένα που να αντικατοπτρίζονται στο άλλο σκέλος της συμφωνίας. Έτσι λοιπόν τα, τα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να προωθηθούν ως ανεξάρτητη συμφωνία. Σας παροτρύνω να το κάνετε αυτό και μάλιστα νωρίς. Άλλες ερωτήσεις σε σχέση με το GSP+. Όπως γνωρίζετε υπάρχει κάποια αμφισημία σχετικά με τις Φιλιππίνες και για κάποιες άλλες χώρες. Κάποιες από τις, κάποιοι από τους δισταγμούς προέρχονται από το γεγονός ότι μόλις μια χώρα, ε, όταν σε μια χώρα δοθεί το GSP+, δεν μπορεί να της αφαιρεθεί ε, και η ιστορία ε, δικαιώνει αυτούς που το υποστηρίζουν αυτό. Η Επιτροπή μας έχει διαβεβαιώσει ότι αν μια χώρα δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις θα της αφαιρεθεί το GSP+. Το GSP+. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, καλώς ορίσατε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια ερώτηση που μου έκαναν εμένα σε μια συνάντηση στην εκλογική μου περιφέρεια στο Midlands για τις μικρές επιχειρήσεις και η ερώτησή μου είναι έχει ανοίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επιχειρήσεις και πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο θα κάνουμε την εμπορική πολιτική τα επόμενα πέντε χρόνια θα καθορίσει το κατά πόσο θα θεωρηθεί γενικώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να κάνει δουλειές με τις επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε ότι πρέπει να συμμετέχουν στη χάραξη τη εμπορική πολιτική όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ο διάλογο είναι πολύ σημαντικό. Αλλά έχω και κάτι να προσθέσω στον καταλογό σα. Δράση. Χρειαζόμαστε πραγματικά να δούμε δράση, να δούμε αποτελέσματα. Και δεδομένου και τον όσων είπε ο κ. Φιέλνερ, έχουμε πολύ μεγάλα χρονοδιαγράμματα όσον αφορά το εμπόριο ε, μεγάλες μακροχρόνιες προθεσμίες ενώ ο κόσμος θέλει να βεβαιωθεί τώρα ότι θα υπάρξουν συναλλαγές νέες ευκαιρίες παντού και φυσικά η συμφωνία TTIP είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία με την οποία έχουμε να ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι να δράξουμε μια ευκαιρία μόλις αυτή φτάνει και ότι μπορούμε να επιταχύνουμε για να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάτι τέτοιο πολύ γρήγορα. Σκέφτομαι και τη Λατινική Αμερική όταν σκέφτομαι για όλες τις ευκαιρίες που έχουμε ε, για αποτελέσματα. Το ίδιο και με τη Σιγκαπούρη και την Ιαπωνία. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και χώρες όπως το Μεξικό που είναι έτοιμοι, που ήρθε και μας είπε είμαστε έτοιμοι να συνάψουμε μια νέα συμφωνία και να ε, την επεκτείνουμε περισσότερο από ό,τι παλιά. Είμαστε έτοιμοι για μια συμφωνία. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό μετά από τη Σύνοδο Κορυφής με το Μεξικό του χρόνου. Θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιο κείμενο του Συμβουλίου Επίσης, ε, ε, εστιαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να δούμε και τι γίνεται παγκοσμίως σε θέματα εμπορίου. Θέλουμε να θέσουμε παγκόσμια πρότυπα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτά που έχουν γίνει και με άλλε χώρε και ε, τι έχει γίνει με συμφωνίες ε, που δεν απασχόλησαν εμά, όπως η συμφωνία μεταξύ Κίνα και Αυστραλία αφορά γεωργικούς πόρους, ενέργεια, εξαγωγή προϊόντων, υπηρεσίες και επενδύσει Είναι σαφέ ότι η Αυστραλία είναι διατεθειμένη για παρουμε συμφωνίες με την Κορέα και την Ιαπωνία και είναι διατεθειμένη να κάνει δουλειέ. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να επεκτείνουμε ό,τι έχουμε δώσει ήδη σε συμφωνίες πλαίσια, αλλά να κάνουμε και συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών με χώρες όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία και να δράξουμε τις ευκαιρίες μόλις εμφανίζονται. Ναι, ε, ε, ε Μαρίτια. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κυρία Επιτροπέ. Έχουμε πλήρες θεματολόγιο ενώπιόν μας και είναι καλό που μιλάτε για διαφάνεια, η οποία πρωτοβουλία ξεκίνησε και πολύ γρήγορα με την καθοδηγητική σας θέση και την ε, εμπλοκή σας και τη συμμετοχή των εμπλεκομένων. Ε, πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν και θα πρέπει να ζητήσουμε από τους Αμερικανούς να διατηρηθεί αυτή η πορεία χωρίς βεβαίως να ε, συμβιβαζόμαστε στα θέματα ουσίας. Έχω διάφορες ερωτήσεις. Αυτή τη βδομάδα συζητάτε συμφωνία για την τεχνολογία της πληροφορικής. Θέλω να σας μιλήσω για την πιθανότητα μιας πρόοδου τις ερχόμενες δύο εβδομάδες, για την Ιαπωνία. Άλλη ερώτηση. Ενώ εμείς διαπραγματευόμαστε με την Ιαπωνία, η Ιαπωνία είναι ο μεγαλύτερος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εταιρική σχέση του ειρηνικού. Πολλοί λένε ότι η Ιαπωνία ε, καθυστερεί την TPP. Και το θέμα είναι πώς αυτό επηρεάζει τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις, εάν τι επηρεάζει δηλαδή, πώς επηρεάζεται η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιαπωνίας και TPP. Τέλος, Τις προηγούμενες εβδομάδες είδαμε μια πρόοδο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ε, είναι θαυμάσιο αυτό, τουλάχιστον για όσους ε, από εμά πιστεύουμε ότι οι πολυμερείς εμπορικές ε, συμφωνίες είναι αξιόλογες. Πώς βλέπετε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τώρα και πώς σκοπεύετε να κινητοποιήσετε την ηγετική θέση της Ευρώπης στον ΠΟΕ. Η Ινδία ήταν επίσης σημαντικός παίκτη. Σημαίνει αυτή η πρόοδος και μια, ένα νέο μέλλον για την εμπορική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας. Ευχαριστώ. Όλος ο κόσμος, ε! Ο Χέλμουντ ίσως θα προσθέσει και μια ανατολική διάσταση ενδεχομένως. Χέλμουτ. Πρόεδρε, θα διαρωτηθείτε. Ξεκινώ με την Ανατολική Ευρώπη. Η κατάσταση στην Ουκρανία και την Ρωσική Ομοσπονδία. Σαφέστατη πρόκληση για σας επίσης αυτή. Διότι έχουμε κοινή ευθύνη να συνεισφέρει το εμπόριο προς την ειρήνη. Και εδώ θα ήθελα να ξεκινήσω όμως με ένα άλλο θέμα που ε, ολοκληρώσατε την εισαγωγή σας και σας ευχαριστώ για αυτή την πλήρη ενημέρωση για τις προθέσεις σας να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γενικής Διεύθυνσης για το Εμπόριο και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ερώτηση σε σχέση με αυτά. Στην ακρόαση είπατε, πρώτο σημείο είναι για μας, ότι θέλουμε να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε το πολυμερές εμπορικό σύστημα ως προσέγγιση Σήμερα αυτό έχει περάσει σε υποδέστερη θέση. Έχετε κάποια σχέδια για τις οριζόντιες επιπτώσεις των διαπραγματεύσεων για το εμπόριο που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση όλα αυτά τα θέματα που θα μπορούν να συγκλίνουν μεταξύ τους. Γνωρίζουμε τι θα σημαίνει το TTIP για την προσχώρηση του Εκουαδόρ για παράδειγμα, την πρόσβαση του Εκουαδόρ την ε, συμφωνία επίσης ε, για την Κολομβία και το Περού και την ένταξη σε αυτό το πλαίσιο και του Εκουαδόρ του Ισημερινού. Ξέρουμε ποιες είναι οι αμοιβέ επιρροές ε, μεταξύ TTIP και των συμφωνιών ε- Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας για παράδειγμα. Πώς αλληλεπεριάζονται αυτά. Σχεδιάζει πραγματικά να κατανοήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σημαίνει για τις χώρες εταίρους, τις τρίτες χώρες και όλα τα 28 κράτη-μέλη όλα αυτά Φυσικά η Ελλάδα έχει κάποια ίσως άλλα ε, συμφέροντα ε, και στοιχεία που ε, εδώ η Γερμανία θα παρισέφερε. Πώς είναι δυνατόν να προσαρμοστούμε σε αυτή την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε κατά τον 21ο αιώνα. Το, η εναλλακτική εντολή για το εμπόριο και τις ε, μη οργανώσεις και υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει θετική συνεισφορά για το παγκόσμιο εμπόριο από πλευράς ε, της πραγματικής οικονομικής ανάπτυξης ε, από διάφορες περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σχεδιάζεται για να συμπεριληφθούν όλες αυτές οι πτυχές ε, και οι συμμετέχοντες να συμμετάσχουν σε μια πραγματική ημερήσια διάταξη ως θεματολόγιο για το εμπόριο. Και τρίτον για την λογική με την οποία προσεγγίζουμε την Συμφωνία Επενδύσεων και Εμπορίου με τις ΗΠΑ, τη Διατλαντική Συμφωνία, μιλήσατε για μια συνεργασία ρυθμιστική. Και αν και οι δύο πλευρές εκφράσουν και θα πάτε στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα, Επίτροπε, αν αναφερθεί, μην ανησυχείτε, δεν θέλουμε να τροποποιηθεί το κοινοτικό κεκτημένο πώς ρυθμιστικά θα προχωρήσει η ρυθμιστική συνεργασία ε, στο μέλλον για την τελευταία τελική διατύπωση. Τι θα σημαίνει για τοπικές αρχές, περιφερειακές αρχές, δήμους, κοινότητες να προσαρμόσουν τα συστήματα με μέσα στα οποία λειτουργούν στις προκλήσεις που θα δημιουργήσει μια τέτοια διεθνούς ε, χαρακτήρα συμφωνία. Και σε σχέση με τα συνδικάτα και τη Γερμανία για παράδειγμα, σε, ε, σε μια συνδιάσκεψη τα συνδικάτα είπαν να μην δεχθούμε τη ΣΥΤΑ αν συμπεριλαμβάνεται το ISDS. Δηλαδή αυτά αυτοί οι φόβοι πώς θα βοηθήσετε να πάψουν να υπάρχουν σε σχέση με τους ε, εργαζόμενους και την κοινωνία των πολιτών ώστε να βρεθούν λύσεις για τα προβλήματά τους από κοινού με τους εμπορικούς εταίρους μας ε, και που θα αποβαίνουν οι λύσεις αυτές υπέρ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ζανέτ. Ζανό. Ευχαριστώ Μπέρντ. Καλημέρα κυρία Επίτροπε. Παρουσιάσετε πολλά και ξεκινήστε με τη διαφάνεια και κάνατε μια πρόταση επί του θέματος αυτού. Ε, διαρκώς αξιολογούμε βέβαια το περιεχόμενο αυτής της πρότασης γιατί αντιλαμβανόμαστε τη γενική αρχή Διεύρυνση τη πρόσβαση στα έγγραφα, αλλά αληθεύει ότι μετά πρέπει να βάζουμε και τετραγωνάκια μπροστά σε κάθε τύπο εγγράφου, Ποιο μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό και ποιο όχι. Και αυτό αποτελεί κομμάτι και της αξιολόγησης που κάνουμε, αλλά αυτό που καθιστάται σαφέ κατά την άποψή μα, προφανέ μάλλον, είναι ότι δεν προχωρήσετε περισσότερο όπως σας επιτρέπουν οι Αμερικανοί. Ουσιαστικά στις αίθουσες ανάγνωσης ε, δεν προτείνεται τίποτα νέο. Για άλλη μια φορά Πρόκειται για το σύστημα για το οποίο έχει συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις Πολιτείες και κατά την άποψή μας αυτό το σύστημα είναι αμφισβητήσιμο. Διότι ναι, το να έχουμε πρόσβαση σε κάποιο πλήθος εγγράφων, μια χαρά εντάξει, αλλά η ουσία των εγγράφων είναι τα έγγραφα που ουσιαστικά θέλουμε, είναι τα ενοποιημένα έγγραφα των διαπραγματεύσεων και εσείς προτείνετε ε, να συνεχίσουν να έχουν σε αυτά πρόσβαση μόνο καμιά δεκαπενταριά ευρωβουλευτές και όταν εγώ ρωτώ δημόσια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον Υπουργό Οικονομικών μου έχετε το ενοποιημένο κείμενο των διαπραγματεύσεων, ελπίζω να το έχει, αλλά πραγματικά ξέρετε δεν μπορεί να πει ναι. Δεν μπορεί να πει έχω στο γραφείο μου αυτό το κείμενο των διαπραγματεύσεων. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν ένα δημοκρατικό πρόβλημα και για άλλη μια φορά θεωρούμε ότι το εγχείρημά σα αυτό υπέρ τη διαφάνεια δεν πάει παραπέρα από όσο σα επιτρέπουν οι Αμερικανοί. Τώρα πιο γενικά και υπόθηκε και από τον συναδελφό μου η, Γενική Συνέλευση, η Εθνική, Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας ε, αντιτέθηκε σε ένα ISDS σε αυτή τη συμφωνία και δεν είναι το πρώτο κοινοβούλιο στην Ευρώπη που εκφράζει την απόψή του για αυτό το θέμα. Ευτυχώς ε, έχουμε δει όλο και περισσότερες μελέτες αξιολόγησης αντικτύπου ε, των συμφωνιών ε, της ΣΕΤΑ και της TTIP και για την TTIP σύμφωνα με την τελευταία αμερικανική μελέτη λέει μείον 5.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και το κέρδος σε θέματα ε, ε, συναλλαγών είναι λιγότερες συναλλαγές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερες με, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τίθεται το ερώτημα, τι γίνεται με κάποια κεφάλαια αυτής της διαπραγμάτευσης που θέτουν σε κίνδυνο την δημοκρατική κυριαρχία και ε, η αμφισβήτηση των επιπτώσεων αυτής της συμφωνίας. Μήπως λοιπόν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνετε θα ήταν να, να ξεκινήσετε με μια νέα αρχή όχι μόνο τι μελέτε που λαμβάνετε από πανεπιστήμια και τα κέντρα μελετών, μήπω πρέπει να ξεκινήσετε να δώσετε μια νέα αρχή σε μια πραγματική εργασία μελέτη των επιπτώσεων αυτή τη διατλαντική διαπραγμάτευση. Και τέλο, πρέπει να σα ομολογήσω ότι για του οικολόγου, όταν μάθαμε ότι θα γίνετε επίτροπο, πάψαμε να ελπίζουμε πολλά και για το φιλελεύθερο κομμάτι των πεπιθυσιών σα. Αντιθέτως, ε, εκεί που μας δίνεται ελπίδες ε, είναι ο μόνιμος αγώνας ε, υπέρ της αηφόρου ανάπτυξη και των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Και αναφέρεται αυτά τα θέματα σήμερα, αλλά δυστυχώς σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν διαπραγματεύεται δεν επιθυμεί τα κεφάλαια αηφόρου ανάπτυξης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων να είναι δεσμευτικά. Εσείς θα αγωνιστείτε κατά αυτού για να αλλάξει. Όταν η Κομισιόν ε, προετοιμάζει κάποια διεύρυνση, κάποιον εξυγχρονισμό της συμφωνίας με το Μεξικό, θα λάβετε υπόψη το δημοκρατικό διακύβευμα που έχουμε σήμερα στο Μεξικό, το ίδιο για το Βιετνάμ. Μιλήσατε για 90 εκατομμύρια πολίτες του Βιετνάμ και εκεί μιλάμε για ένα εξαιρετικά προβληματικό πολιτικό καθεστώς, το ίδιο και στη Βερμανία. Και ε, δεν έχει λίστα τελειωμό. Δεν άκουσα στη συζήτησή σας τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγματική διάσταση ε, των συμφωνιών με αυτές τις χώρες ώστε να τηρηθούν τα, δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος, λιγότερο ίσως εύγλωτος από τον προλαλήσαντα. Έχω ε, ρωτήσει σε δύο ε, κατηγορίες. Εναρκτήρια ομιλία σας. Λέτε ότι το εμπόριο προκαλεί θέση εργασίας ε, και επενδύσεις και ανάπτυξη. Έχετε δίκιο. Αλλά προηγουμένως είχατε μιλήσει για την πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς η, εμπορική πολιτική σας θα προωθήσει την πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα συμβεί όταν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της πολιτικής ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον στόχο που έχετε θέσει για θέση εργασίας, ανάπτυξη και επενδύσεις. Η πολιτική ατζέντα θα επικρατήσει ή η θέση εργασίας, η ανάπτυξη και οι επενδύσεις που τόσο επιθυμούμε. Δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία η οποία επαναλήφθηκε πολύ εύγλωτα από τον συνάδελφο Helmut Scholz σχετικά με την ISTS και την TTIP. ISTS είναι η η διαδικασία ε, συμφιλίωσης των επενδυτών. Και η TTIP είναι η, η συμβολία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής είπε στις 22 Οκτωβρίου 2014 στο Στρασβούργο ζήτησα τον, από τον Φρανς Τίμερμαντ να με συμβουλεύσει επ' αυτού, δηλαδή για την ISTS δεν θα υπάρχει ρύθμιση ε, κράτους επενδυτή ε, στην TTIP. Οπότε ρωτάω, εσείς τώρα που εμπλέκεστε, εσείς είστε η Επίτροπος του Εμπορίου. Αναφέρεστε όμως για το, για το, βασικό, για το βασικό θέμα. Πολλοί ψήφισαν εναντίον σας, γιατί θεωρούσαν ότι δεν είστε κατάλληλη θέση. Οπότε μήπως θα έπρεπε να έρθει εδώ ο κύριος Τίμερμανς να απαντήσει στην ερώτηση τη δική μου και του κυρίου Σόλτς. Γιατί ο κύριος Τίμερμανς είναι αυτός που έχει την ευθύνη από ό,τι φαίνεται, όχι εσείς. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να απαντήσετε στον πρώτο γύρο των ερωτήσεων, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. πο... Ναι, η κυρία Λεπέν όμως, που ήθελε να παρέμβει. Συνάδελφοι, έχουμε ένα σαφή κανόνα. Στον πρώτο γύρο οι κοινοβουλευτικέ ομάδε έχουν το δικαίωμα να θέσουν ερωτήσει. Στον δεύτερο γύρο έχουμε 22 που έχουν ζητήσει τον λόγο να παρέμβουν. Και θα είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Λοιπόν, πρώτο γύρος. Τώρα απαντάτε εσεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινώ με την πρώτη ερώτηση του Κρίστοφερ Φιέρνερ. Συμφωνώ, παίρνει πολύ χρόνο για αυτέ τι διαπραγματεύσει. Όμως φυσικά με κάποιες ευκαιρίες μπορούμε να επιταχύνουμε τα πράγματα. Χρειάζεται όμως χρόνος. Έχουμε πολύ φιλόδοξο θεματολόγιο στην ημερήσια διάταξη. Θέματα που πρέπει να πραγματευτούμε με τους εταίρους μας τον Καναδά, τη είπα Είναι δυσχερέ εγχείρημα. Έχουμε πολύ περίπλοκο σύστημα. 28 κράτη-μέλη, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει από κάθε κοινοβούλιο, από κάθε κράτο μέλο να επικυρωθούν όλα αυτά. Χρειάζεται χρόνο. Αλλά στο μεσοδιάστημα εντωμεταξύ πρέπει να δώσουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Να δουν περί τίνο πρόκειται. Η διαφάνεια είναι ένα μέρο, ε, μία παράμετρο. Να δούμε, ορίστε, να πούμε, ορίστε, αυτό αναμένουμε να είναι η τελική έκβαση. Οι συνεργάτε μου και εγώ θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να αναφέρουμε στους ενδιαφερόμενους εμπλεκόμενους πού βρισκόμαστε σε αυτό το γύρο διαπραγματεύσεων. Ελπίζω θα μπορούμε να δείξουμε χειροπιαστά αποτελέσματα αυτών των διαπραγματεύσεων για να γνωρίζουν όλοι προς τα που κινούμαστε. Θα παίρνει χρόνο, θα πάρει χρόνο αυτό. Θα έχουμε το νομικό χτένισμα όλων αυτών που παίρνει και αυτό χρόνο, μεταφράσεις, διατυπώσεις, όλα αυτά απαιτούν χρόνο. Και το 2017 όταν θα έρθει η χρονική στιγμή να εγκριθούν όλα για να αρχίσουν να ισχύουν θα χρειάζεται αυτός ο χρόνος. Πρέπει να πούμε ότι το εμπόριο πρέπει να βρεθεί έτσι στο προσκήνιο και να δούμε πώς θα ενταχθεί στην γενικότερη πολιτική μας υπέρ της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της ανάπτυξης. Δεν υπάρχει αντίφαση σε αυτό και αυτό είναι μέρος τμήμα της πολιτικής μας και ελπίζουμε ότι και αυτό θα μπορέσει να ενταχθεί στο έγγραφο για την μελλοντική αυτή, ε, το μελλοντικό καθορισμό αυτών των πραγμάτων όπως ανέφερε και ο κύριος ε, ε, David Martin. Και με ιδιαίτερη χαρά θα μπορέσω να το συζητήσω μαζί σας αυτό ε, και με ποιο τρόπο θα μπορέσει να γίνει αυτό θα το μάθουμε και θα το προτείνει και ο Πρόεδρος αν θέλετε εξειδικευμένα να έχουμε μια συζήτηση επ' αυτού αν προετοιμάσετε κάποιο έγγραφο με ενδιαφέρει να ακούσω τις απόψεις σας επ' αυτού προτού προχωρήσουμε στην τελική διατύπωση Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια τελική διαβούλευση κατά τα τέλη του επόμενου έτους. Θα έχουμε ένα, πλήρη έτος, ένα πλήρες έτος για να συζητήσουμε προτεραιότητες, πώς όλα αυτά τα θέματα και παράμετροι θα ενταχθούν, διμερεί, πολυμερεί, θέματα, μονομερείς πρωτοβουλίες και αυτόνομες ε, αυτοτελεί συμφωνίες επίσης. Και όσον αφορά την, ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το ΔΕΚ και τη Σιγκαπούρη. Δεν γνωρίζω σε ποιο άρθρο αναφέρεστε, αλλά ο προκάτοχός μου, Κάρεντε Χούχτε, που αποφάσισε να προσφύγει στο Ευρωδικαστήριο, δεν ε, απεστάλλει όμως το θέμα αυτό σε σχέση με την, ε, το διάστημα πριν την αλλαγή, την, πριν πάρει τα ενία της η νέα Επιτροπή. Και είπε ο κύριος Γιούνκερ ας δούμε τι θα γίνει σε σχέση με αυτό ε, στο παραπέντε ας το πούμε έτσι είναι πραγματικά πολύ μικρό το χρονικό διάστημα πιεστικός, πιέζει πολύ ο χρόνος αλλά θα δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει σε σχέση με αυτό για την διαφορετική άποψη για την Σιγκαπούρη γνωρίζω την άποψή σας ότι είναι μια ξεχωριστή μονάδα και ότι πρέπει από κοινού να αντιμετωπιστεί για το JSP Plus ε, υπάρχει κάτι που πραγματικά πιστεύω σε αυτό και είναι αυτό είναι ένας τρόπος να μπορέσουμε να εντάξουμε τις φτωχότερες χώρες για το πώς μπορούν στο παγκόσμιο εμπόριο να έχουν έναν ρόλο που θα έχει νόημα. Αηφορία, ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα. Ξέρετε ότι πρέπει πολλές συμβάσεις να υπογραφούν πρωτού γίνει κάποιος δεκτός σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Μετά δεν σημαίνει ότι όλα έγιναν και τελείωσαν. Πολλές από τις χώρες αυτές, κάποιες από αυτές έχουν προβλήματα. Μπορούν όμως να τεθούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο όπου θα υπάρχει διαρκής επιτήρηση, εποπτεία και διάλογος και μπορούμε να ε, ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. αν υπάρχουν παραβιάσεις θα δράσουμε, αλλά όταν θα υπάρχει η δυνατότητα να εμπλέξουμε αυτές τις ε, χώρες, την κοινωνία των πολιτών, τα συνδικάτα, τις, ε, του, διάφορες οργανώσεις για να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να προαγάγουμε αυτά τα πράγματα θα αποβούν πιο ε, θα είναι μεγαλύτερο το όφελος για τους πολίτες πολίτες αυτών των χωρών. Δεν θα έχω καμία ε, επιφύλαξη αν υπάρχουν συστηματικές παραβιάσεις και παραβάσεις να προσφύγω και να χρησιμοποιήσω το όπλο του παγώματος ή των κυρώσεων. Ας δούμε όμως πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά όχι μια υποχρεωτική, ένα υποχρεωτικό πάγωμα άμεσα μόλις κάτι έχει συμβεί, να δούμε ακριβώς ε, τι συμβαίνει. Αν ρωτήσατε αν θα είναι ανοιχτό για τις ε, επιχειρήσεις, πρέπει πολλές εσωτερικές μεταρρυθμίσεις να γίνουν για να διασ διασφαλίσουμε ότι θα δρέψουμε όλα τα ωφέλη από την οδηγία για την ενιαία εσωτερική αγορά και τις μεταρρυθμίσεις που υποσχεθήκαμε τόσα χρόνια ότι θα προχωρούσαμε. Αλλά είμαστε ανοιχτοί στους εταίρους μας, για τους εταίρους μας και εκείνοι πρέπει να ανοίξουν τις αγορές τους. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά πρέπει να εμπλακούμε σε αμφίδρομη δράση με τον κόσμο γύρω μας. Αναφέρατε το Μεξικό. Μίλησα με τους αρμόδιους τηλεφωνικά την προηγούμενη εβδομάδα. Αποστήλαμε ερωτήματα σε σχέση με αυτό το ενεξελίξει εγχείρημα για να δούμε ποιε είναι οι θέσει του. Αναμένουμε τι απαντήσει του. Υπάρχει λοιπόν διάλογο. Και όταν θα βρούμε ότι έχουμε το ίδιο επίπεδο φιλοδοξιών και προθέσεων θα μπορέσουμε να ξαναξεκινήσουμε αυτέ τι διαβουλεύσει ε, κατά το επόμενο έτο. Διότι το επιθυμεί και το Μεξικό για την ε, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία είναι εξαιρετική εταίρη ε, Να δούμε τι μπορούμε να, ε, ποια ωφέλη θα μπορούν να υπάρξουν ε, μέσω μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου διότι το πιο, τα πιο ευαίσθητα θέματα εκεί είναι φυσικά τα θέματα τα γεωργικά για τη γεωργία. Να δούμε δηλαδή σε σχέση με τα ωφέλη και τις απώλειες τι ακριβώς γίνεται, τι, ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Αυτό είναι μέρος της εξίσωσης που προσπαθούμε να επιλύσουμε σε σχέση με αυτές τις χώρες. Τώρα α, κάνα, θέσατε μία ερώτηση για το ε, το ETA και αύριο θα έχουμε διαπραγματεύσεις στη Γενέβη που θα ξαναξεκινήσουν για το θέμα του ETA. Πρόοδος που πιέσαμε εμείς να ε, σημειωθεί και σε σχέση με, τις, με τους εταίρους μας ε, υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει ακόμα να επιληθούν όσον αφορά ε, εμπορεύματα και ο στόχος μας είναι, μια και οι διαβουλεύσεις θα ξεκινήσουν αύριο στη Γενέβη και θα συνεχιστούν για μια εβδομάδα, ελπίζουμε ότι κάτι χειροπιαστό θα μπορέσει να απορρεύσει και θα βρεθούν λύσεις σε αυτά τα ζητήματα. Σημαίνει αυτό ότι επιστρέφει η Ινδία, ίσως κάποιοι θα το θεωρούσαν αυτό. Είχαμε χαμηλού επίπεδου δραστηριότητες σε σχέση με τις ε, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις με την Ινδία και θα θέλαμε να γίνει αυτό, να ενταχθεί. Δεν, θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί όμω. Να δούμε, θέλει να φτάσει εκεί η Ινδία και να το πετύχει αυτό και τότε θα ανταποκριθούμε εμεί. Για τον ΠΟΕ Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, όπω είπα αρχικά, για ε, τον ΠΟΕ, η συμφωνία για το μέσο για τη διευκόλυνση του εμπορίου υπεγράφει την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ θετικό αυτό και υπάρχει και η προοπτική να ολοκληρωθεί ο γύρος της Δόχα κατά τα τέλη του 2015. Θα υπάρχει μια άτυπη υπουργική συνάντηση στον Ταβός, θα συνεχιστούν ε, οι επαφές και σε σχέση με την συνάντηση όσον αφορά την Γενέβη την επόμενη εβδομάδα στόχος είναι να υπάρξει υπουργική συνάντηση κατά το 2015. Θα, θα ανοιχνεύσουμε και θα ε, προσπαθήσουμε να ταυτοποιήσουμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν στη Γενέβη αυτό για να ολοκληρωθεί η Ντόχα. Σε εσά ε, η πολυμερή ημερήσια διάταξη είναι πολύ σημαντική για μένα. Είπατε ότι έφτασε από πρώτο, πρώτη προτεραιότητα ε, σε τρίτη, τέταρτη. Αλλά χαίρομαι πολύ που συνεχίζονται τώρα οι προσπάθειες. Ίσως υπήρχαν επιφυλάξεις αλλά τώρα έχει πράγματι αποτροχοπεδηθεί η κατάσταση και βρίσκεται πάλι, δρομο, έχει δρομολογηθεί εκ νέου. Φυσικά πολλές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις υπό το πνεύμα του ΠΟΕ έγιναν, αλλά όχι υπό την αιγίδα και τη στέγη του ΠΟΕ. Πρέπει όμως να ενταχθούν όλα αυτά υπό την αιγίδα και στέγη του ΠΟΕ. Εκεί ανήκουν. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, σε αυτό το αίσιο πέρας, σε αίσιο τέλας. Η δική μου εκτίμηση είναι προσπαθούμε με αξιολογήσεις ε, για αυτές τις χώρες να δούμε ποιε προοπτικές υπάρχουν υπάρχουν. Υπάρχουν τόσες πολλές ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και βρίσκονται όλες υπό εξέλιξη παγκόσμια που είναι πολύ δύσκολο να ξέρει, να γνωρίζει κανείς για αυτό τον μεγάλο σύνθετο ιστό τι ακριβώς συμβαίνει και να έχει μια συνολική ε, εικόνα για το δίκαιο εμπόριο. Ναι, πράγματι μπορεί να έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα για το JSP+, Plus, ε, το JSP-SYN ε, ε, διευρυμένης ε, μορφής και εμβέλειας. Και έτσι λοιπόν πράγματι είναι πολύ χρήσιμη αυτή η προσέγγιση. Μπορούν να διαδραματίσουν ένα ρόλο για την κατάθεση στοιχείων για να διαπιστωθεί αν υπάρχει παραβίαση αηφορίας, θεμελιωδών δικαιωμάτων, ελευθεριών σε σχέση με τις χώρες αυτές, ώστε να πρέπει τότε να δράσουμε. Λυπούμε πρόεδρε, αλλά ήταν τόσες πολλές, τόσες ερωτήσεις που πρέπει να συνεχίσω δεν μακρηγορώ, για το ρυθμιστικό πλαίσιο. Εκεί πραγματικά είναι το κεφάλαιο που μπορούμε να έχουμε τα μεγαλύτερα ωφέλη, αν τα πάμε καλά, χωρίς να υποβαθμίσουμε τα περιβαλλοντικά ως προδιαγραφές ε, ε, από πλευράς γνώμονα που θα θέσουμε και να δούμε για παράδειγμα σε σχέση με τις ε, ε, ε επιθεωρήσεις ε, κάποιων βιομηχανιών crash test σύγκρου, δοκιμές σύγκρουσης για αυτοκίνητα για γιοταχή προσπαθούμε όλα αυτά να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο ή αν παρισφρέουν για πρώτη φορά να ξεκινήσουν από μια κοινή προσέγγιση από κοινά, θεμέλια να εξετάζονται. Τώρα για τη διαφάνεια. Επιτρέψτε μου να πω κύριε Ζαντό εσείς θα δείτε περί τίνος πρόκειται. Τώρα προσπαθούμε και στόχος μας είναι στο διαδίκτυο να είναι πολλά έγγραφα διαθέσιμα για την παιδαγωγική την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε ώστε να είναι επωφελής για τους πολίτες, να είναι όλα αυτά προσπελάσιμα για τα κράτη-μέλη, για τους ε, πολίτες. Όλα αυτά θα δώσουν μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια στα όσα συζητούμε. Η δυνατότητα προσπελασιμότητας αυτών των εγγράφων για τους ευρωβουλευτές. Προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο να το καταφέρουμε. Στόχος μας όμως είναι όλοι οι ευρωβουλευτές να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα για να μπορούν να τα συμβουλεύονται. Και αυτό φυσικά θα ας το πω έτσι, θα είναι μια ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης και δεν θα υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί. Δηλαδή δεν θα είναι τόσο διαβαθμισμένα ή περιοριστικού χαρακτήρα αυτά τα έγγραφα για να τα συμβουλευτεί κανείς. Φυσικά θα πρέπει και οι τεχνικές λύσεις για τους ε, παράδειγμα ευρωβουλευτές και τους ε, υπουργούς να μην χρειάζεται να πάνε σε ένα ειδικό αναγνωστήριο για να τα ε, συμβουλευτούν. Θα μπορούσε να υπάρχει και μια ηλεκτρονική δυνατότητα ώστε σε ένα συγκεκριμένο μέσο συγκεκριμένων συσκευών ε, και χώρων να μπορούν να, τα να συμβουλευτούν αυτά τα στοιχεία. Τώρα για το ISDS. Μάλιστα, πράγματι, έχω συνειδητοποιήσει τις επικρίσεις που έχουν ασκηθεί. Και επίσης ε, γνωρίζω ότι η συμφωνία ε, ΣΥΤΑ έχει θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε από τα κράτη-μέλη και επίσης ε, για την ε, ε, Καναδική Συμφωνία έχει ληφθεί ένα πολύ σημαντικό η ΣΥΤΑ, η Συμφωνία με τον Καναδά ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για να υπάρξει πλαίσιο διαφάνειας, ανοιχτό πλαίσιο ώστε να εγγυηθούμε ότι το δικαίωμα, ας το πω έτσι, της, ε, ασφάλειας για τους πολίτες ε, ε, δεν θα έχει τέτοια, τέτοιο ρόλο ώστε άλλα δικαιώματα όπως για παράδειγμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων να περιφρονούνται. Και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε, θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Όμως ε, το ε, ΣΕΤΑ έχει ολοκληρωθεί, δεν ξανανοίγει, ούτε απομένουν εκκρεμότητες. Και φυσικά μπορείτε να προσκαλέσετε τον κύριο Τίμερ μας να έρθει εδώ και να διαβουλευτείτε μαζί του. Κανένα πρόβλημα. Μπορώ να σας διασφαλίσω όμως με τον πρόεδρο Γιούνκερ και τον Φρανς Τίμερ μας ε, συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Δεν έχουμε διαφορές απόψεων, δεν δεν αποκλίνουν οι απόψεις μας. Είναι φυσιολογικό θα έλεγα σε σχέση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιος για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για την προάσπιση των αξιών μας, για καλύτερες διατάξεις και ρυθμίσεις, να ενημερώνεται και αυτός και να έχει συντονιστικές αρμοδιότητες από αυτών των θεμάτων για το ISDS για παράδειγμα. Διότι πραγματικά εδώ περί αυτού πρόκειται. Όλοι οι αντιπρόεδροι έχουν θέματα σε υψηλότερα επίπεδα ευθυνών από ότι οι υπόλοιποι ε, επίτροποι. Είναι ένας τρόπος αυτός όχι να υποβαθμίζονται κάποιοι να αποκλείονται, αλλά να υπάρχει συντονισμός αρμοδιοτήτων κατά τον βέλτιστο τρόπο. Θα προσέλθει αν τον προσκαλέσετε. Εγώ όμως είμαι η Επίτροπος αρμόδια για το εμπόριο και τις εμπορικές σχέσεις. Σίγουρα θα συνεργαστούμε μαζί με τον κύριο Τίμερμασά, αλλά δεν παρεκκλίνουν οι απόψεις μας. Έχω τις δικές μου αρμοδιότητες και θα πρέπει να αυτό να το ανεχτείτε καμιά φορά. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε 21 άτομα που ζητούν το λόγο. Αυτό σημαίνει ότι μόνο επειδή έχουμε 22 λεπτά, έχουμε τη δυνατότητα να σας δώσουμε μόνο ένα λεπτό στον καθένα. Αλλιώ δεν θα προλάβει η Επίτροπος να απαντήσει. Σκεφτείτε λοιπόν κατά πόσο είναι απολύτως αναγκαίο να κάνετε ερώτηση τη Ήδη απαντήσαμε τόσο πολλά στο πρώτο γύρο. Κύριε Ρίγκλερ, είστε πρώτος. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για τις ε, απόψεις και την ενημέρωση. Θεωρώ κύριε Πρόεδρε είναι απαραίτητη αυτή η ερώτηση. Θέλω η κυρία Επίτροπος να αγγίξει ένα θέμα που δεν συζήτησε σήμερα, την Κίνα, σημαντικό μας εταίρο. Τρεις ερωτήσεις ε, για αυτό την εταιρική σχέση. Πρώτα απ' όλα, οι σχέσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας ε, έχει πολλά επίπεδα. Έχουμε διαλόγους, ε, σχέσεις σε επίπεδο κράτους μέλους, κομισιών, πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο κομμάτων, στο πλαίσιο πολλών πρωτοβουλειών που ξεκίνησαν ήδη 20 χρόνια πριν. Θεωρείτε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος ώστε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή φωνή στην Κίνα. Κάτι τέτοιο θα ήταν καλό τι προβλέπετε από αυτού. Δεύτερη ερώτηση. Το ζήτημα της πρόσβασης στην αγορά και των φραγμών που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά. Και το τρίτο ζήτημα, ένα ενδεχόμενο πώς προβλέπετε να εξελιχθεί ο διάλογος για την επενδυτική συμφωνία ε, με την Κίνα και επίσης ε, η κατάσταση στην Ταϊβάν. Ε, το Κοινοβούλιο ε, έκανε ένα ψήφισμα πριν από ένα χρόνο για τις σχέσεις με την Ταϊβάν. Ε, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουμε κάποιο διάλογο με την Ταϊβάν. Ευχαριστώ κύριε Κέπρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε. Οι εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χρειάζονται σήμερα 7 με 10 χρόνια. Χρειάζεται να πάρετε πόρους από αλλού στον προϋπολογισμό για να υποστηρίξετε τη διαπραγματευτική ομάδα και κάτι άλλο Θεωρείτε ότι χρειαζόμαστε και άλλον διαπραγματευτή ε, για την Ινδία πέραν ε, ξεχωριστά από τον διαπραγματευτή της TTIP ε, γεγονός που σημαίνει ότι η Ινδία θα ακολουθήσει την TTIP και αυτό θα χρειαστεί περισσότερα χρόνια δηλαδή θέλω να, δώσω, να στείλω ένα μήνυμα ότι την Ινδία τη βλέπουμε σοβαρά και θα, προσπαθήσω, θα θέλαμε να μην καθυστερήσει να επιταχύνουμε τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ κύριε Σίκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο Σικού. Ε, ε, κυρία Μάλμστραμ, όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην προηγούμενη συζήτηση σας παρουσίασα κάπου στις σκέψεις μου τα στατιστικά στοιχεία μας λένε ότι το 3% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μόνο επιτυγχάνουν να αποκτήσουν μια έδρα στο εξωτερικό. Η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μας δεν σκέφτεται καν το ενδεχόμενο διεθνοποίησης. Και το 98% του παραγωγικού του αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό πέραν του καταμερισμού και της διαθεσιμότητας των πόρων να σκεφτούμε να έχουμε μια πολιτική η οποία να οδηγεί και στη σύναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Θεωρώ ότι πέραν της διαφάνειας, πέραν των διαφόρων πτυχών και διαστάσεων που έχουν οι συμφωνίες αυτές, ε, οι συμφωνίες αυτές ε, πρέπει να βοηθήσουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν με θετικά αποτελέσματα. Σας ρωτάω λοιπόν ποια θα είναι η πολιτική σας μέσα στην επόμενη πενταετία όσον αφορά αυτό το στόχο. Ευχαριστώ. Merci, Madame Ευχαριστώ κυρία Λεπέν. Ωραία κυρία Επίτροπε και εγώ σας καλωσορίζω. Προϊθανότητα δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ σε τίποτα. Σας το ανακοινώνω. Έχω 51 δευτερόλεπτα που πολύ ευγενικά μου εκχωρεί ο κύριος Πρόεδρος παρότι είμαι η επικεφαλής της μεγαλύτερης αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από μία από τις μεγαλύτερες χώρες του, ε, της Ευρώπης, στη Γαλλία. Ευχαριστώ για τη γενναιοδορία Είμαι σοκαρισμένη για το πώς δημιουργείται απόλυτη αδιαφάνεια όσον αφορά ότι το πει, έκανα ένα αίτημα τον Ιούλιο που πετάξετε στα σκουπίδια στο πλαίσιο αυτής της δημοκρατικής διαδικασίας ε, και μετά έστειλα μια επιστολή πριν από τρεις εβδομάδες ώστε να αποκτήσω πρόσβαση στην αίθουσα ανάγνωσης παρά τη θέση μου, παρά το όσα αντιπροσωπεύω, παρότι σας ενοχλούν και παρά το ότι είμαι μέλος της Επιτροπής αυτής δεν απέκτησα πρόσβαση σε αυτή την γνωστή, τη φημισμένη αίθουσα ανάγνωσης. Ναι, Στείλατε λοιπόν μια επιστολή γεμάτη καλές προθέσεις, κερδίζετε λίγο χρόνο και εξάλλου δεν ε, αποφασίζετε να έχουμε πλήρη διαφάνεια. Αυτό είναι η δημοκρατία σας. Όμως η δημοκρατία είναι πλήρης διαφάνεια, είναι η κυριαρχία του λαού που μέσω των εκπροσώπων του μπορεί να πρέπει να γνωρίζει ακριβώς ποια είναι η πρόοδος των εργασιών που γινόνται ώστε να μπορέσει να γίνει συζήτηση στην εν λόγω χώρα. Για να τελειώσω, συγγνώμη μου δίνω λίγα ακόμη δευτερόλεπτα, θα ήθελα να μάθω κατά πόσο η μελέτη για την οποία μίλησε ο κ. Ζαντό προηγουμένως, η οποία είναι πολύ ε, ε, σοβαρή όσον αφορά τις συνέπειες ε, για το TTIP που θα έχει πτώσει του ΑΕΠ σε πολλές χώρες, ειδικά στη χώρα μου, στη Γαλλία, άνοδο της ανεργίας, μείωση φορολογικών εσόδων, κίνδυνο αστάθειας. Έχετε διαβάσει αυτό το έργο που αντιτίθεται στη μελέτη της ε, Κομισιόν που προβλέπει μια ισχνή ανάπτυξη του 0,4% του ΕΠ ή θα το πετάξετε και αυτή τη μελέτη στα σκουπίδια όπως το ψήφισμα που εγώ υπέβαλα. Ευχαριστώ. Hello, uh, Commissioner, and uh, I come to... Κύριε Επίτροπε, γεια σας και μπαίνω στην ουσία κατευθείαν. Έχετε δεσμευτεί υπέρ της διαφάνειας. αυτό είναι σημαντικό θα εφαρμόσετε την διαφάνεια που ανακοινώνατε για την TTIP και σε άλλες διαπραγματεύσεις. Αναφέρομαι στο PISA. Δεν έχουμε την εντολή, δεν έχουμε δει την εντολή, δεν έχουμε το ε, κανονιστικό σκέλος της συμφωνίας και ελπίζουμε ότι θα δημοσιευθεί, διότι μόνον όταν μπορούν να δουλέψουν πάνω στα κείμενα οι ε, βουλευτές μπορούν να διαλύσουν τις υποπτήσεις. Όλα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα και όχι άλλα ε, Όχι κατά περίπτωση. Έχω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε αυτή τη στιγμή. Τι συζητείτε όσον αφορά το κεφάλαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Φαίνεται, φαίνεται χωρίς να έχουμε τα έγγραφα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν υποβάλει προτάσεις που περιλαμβάνουν και παραθέτω κανόνες ροής δεδομένων που ε, κάνουν εξαίρεση για την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων. Γνωρίζετε τη θέση μου και στο παρελθόν αλλά και τώρα και τη θέση μας. Μιλάω εξ ονόματος αυτού του σώματος. Γνωρίζετε τη θέση του σώματος και δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτό θα περάσει. Επίσης ενημερωθήκαμε από την, ήδη από την περασμένη πέμπτη. Μοιάζει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν κάνει μια περιοριστική πρόταση στο Συμβούλιο ε, Εμπορίου Επιρεσιών του ΠΟΕ για να υπάρχει το ηλεκτρονικό εμπόριο στο πλαίσιο του προγράμματος εργασία είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επανέλθω σε δύο-τρεις απαντήσεις της Επιτρόπου που δεν ήταν επαρκείς. Πρώτον, ο Ντέιβιτ Μάρτιν, ρώτησε για τη Σιγκαπούρη. Γνωρίζω τη θέση σας, είπατε πρέπει να τη συζητήσουμε. Δηλαδή ποια είναι η θέση σας, γιατί ε, εμεί έχουμε ξεκάθαρα ε, επιχειρηματολογία για τον διαχωρισμό. Ποια είναι η θέση της Επιτρόπου. Δεύτερον, αυτό που δεν μου φάνηκε απόλυτα σαφή, το ISDS σε σχέση με την συμφωνία ΣΕΤΑ, ε, είπατε ναι και μετά θα, συζητήσουμε. Δηλαδή τι σημαίνει, θα συζητήσουμε ή δεν θα συζητήσουμε. Και τρίτον, είσαστε υπέρ της TTIP, η οποία πρέπει να είναι ρεαλιστική. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει μια ρεαλιστική TTIP. Ε, νομίζω ότι θα έχετε καταλάβει ότι πολλοί από εμά είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και σύμφωνα με πρόσφατες ε, μελέτες διαπιστώθηκε ότι η ευτυχία που μας υποσχέθηκε η Κομισιόν και η, ο προκατοχός σας δεν, είναι ακριβώς ε, δεν έχει πραγματοποιηθεί και τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε και μια να εφαρμόσουμε την αρχή της επιφύλαξης γιατί υπάρχουν υποθέσεις αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και απειλές για τους μισθωτούς, για την τεχνογνωσία και για πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, πώς απαντάτε σε αυτά. Ευχαριστώ κύριος Μάρος. Η ISTS έχει σαφώς εξαντληθεί ως θέμα, περνάω κατευθείαν στη Σιγκαπούρη. Ε, μία φιλική προειδοποίηση, αν μου επιτρέπετε. Ίσως να είναι λάθος τακτικής, σοβαρό λάθος τακτικής, να μην ακούσετε την πρόταση του David Μάρτιν, όχι επειδή είναι του David Μάρτιν, αλλά επειδή είναι καλή πρόταση. Ο τομέας των ε, ε, αγαθών και των υπηρεσιών να αντιμετωπιστεί χωριστά. Καμιά φορά ακούγεται σαν εμείς εδώ να έχουμε παγιδευτεί στην απόφασή μας να διαχωρίσουμε και ότι προκαταλαμβάνουμε τη, με τη θέση μας αυτή μελλοντικέ συμφωνίες. Πολλοί εδώ θα ψήφιζαν υπέρ οποιασδήποτε καλή συμφωνίας που θα ε, ερχόταν εδώ αν αυτή η ISDS ε, σε σχέση με τη Σιγκαπούρη. Δεύτερον, περιμένετε ομαλή μετάβαση ε, για, την Κίνα στον τομέα της αγοράς εργασίας του 2016. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σας κάνω μια ερώτηση για ένα θέμα που δεν έχουμε συζητήσει ακόμα. Να σας ρωτήσω κατά πόσο η Κομισιόν έχει την πρόθεση να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για να ξεμπλοκάρει το φάκελο του εξυγχρονισμού των ε, μέσων υπεράσπισης που γνωρίζουμε ότι έχει μπλοκάρει στο Συμβούλιο. Αλλά στο πλαίσιο της πολύ θετική σας προσέγγισης ε, σεβασμού των, θεσμικών, ε, των θεσμών και συνεργασίας θεωρούμε ότι το έργο του Κοινοβουλίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν αξίζει τίποτα. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι απαραίτητο ώστε να δημιουργήσει μια ισορροπία και καλή ε, διοργανική συνεργασία. Καλό είναι λοιπόν η Κομισιόν να δράσει ενεργά ώστε να ξεμπλοκάρει τα πράγματα και έτσι οι εργασίες του παρόντος κοινοβουλίου να αναγνωρίζονται και όχι να χάνονται. Με αυτή τη μέθοδο θα ενισχύσουμε και την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Λαντσπάγης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Έχω ένα πρόβλημα, μια ιδέα η οποία γεννήθηκε το μυαλό των ηγετών του Κρεμλίνου το 2010 τον, την τον κοινό ευρωπαϊκό χώρο από τη Λισαβόνα μέχρι τον Βλαδιβοστόκ. Και βλέπω ότι αυτή ξαναμπαίνει στο κοινοβούλιο και στα διάφορα θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Οπότε αγαπητοί επίτροπε, η ερώτησή μου είναι τι πιστεύετε από αυτού εσείς. Υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθεί κατά κάποιο τρόπο αυτή η ιδέα περνάμε από το δεν συνεργαζόμαστε ως συνήθως στο περισσότερα με λιγότερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις ξεκάθαρες θέσεις της Επιτρόπου και συμπεριλαμβανομένης και της έμφασης στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανάπτυξη και τη διαφάνεια στα πλαίσια της TTIP. Ως μόνιμος εισηγητής που για τη Ρωσία που συντάσσει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για τη Ρωσία. Γνωρίζουμε την προσάρτηση της Κρυμαίας και την κλιμάκωση της κατάστασης στην Ανατολική Ουκρανία, η οποία έχουν αφήσει σε στασιμότητα τις θέσεις ε, της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας, πράγμα που επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι η ρωσική οικονομία ε, βρίσκεται σε πτώση λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαίου στο πλαίσιο λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνει ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί ένας διάλογος. Οπότε έρχομαι σε ένα ερώτημα που είναι διερευνητικό αλλά και προσπαθεί να δείξει ποια θα είναι οι προοπτικές συνεργασίες ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Θα δούμε ποιοι θα είναι φυσικά οι όροι της κατάπαυσης του πυρός στα πλαίσια της συμφωνίας του Μίνσκ και αν τηρηθούν αυτοί. Οι προτάσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί έχει γίνει μια προσπάθεια συμπεριλάμβουν και τις ΗΠΑ αλλά χωρί σοβαρέ συνέπειε. Λοιπόν, εσεί Επίτροπε, πώ βλέπετε την πιθανή σημασία τη διατήρηση του διαλόγου με τη Ρωσία και τι είδου φιλοδοξίε έχει από αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που ήρθατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ουσιαστικά είναι κάτι το αυτονόητο όμως αυτό να προσέρχεστε εδώ. Μία και μόνο ερώτηση έχω. Δεν είναι πραγματικά ερώτηση, είναι παρατήρηση. Αν ακούει κανείς εδώ τι λένε οι συνάδελφοί μας και όταν τα βλέπει όλα αυτά υπάρχουν τόσα πολλά τόσα πολλά σχέδια και προγράμματα με διαφορετικές περιφέρειες, με διαφορετικές περιοχές που όλα θέλουμε να τα καταφέρουμε. Και εσείς κάνετε λόγο εδώ για διαφάνεια. Αλλά μόνο όσον αφορά την TTIP και όχι για τα υπόλοιπα. Υπάρχει κάτι άλλο πέρα από διαφάνεια. Ωραίο είναι να υπάρχουν στο διαδίκτυο αυτά. Όμως ε, οι σελίδες αυτές, αλλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται μια πολύ καλή στρατηγική για την επικοινωνία με τους πολίτες επικοινωνιακά εμείς ως Ευρωβουλευτές τα καθημερινά, κάθε εβδομάδα είμαστε σε επαφή με τους ψηφοφόρους μας, με τους πολίτες στις πιο διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης. Εσείς ζείτε εδώ στην εφελοκοκυγία των Βρυξελών, ωραίο για σας αυτό, αλλά πρέπει να επικοινωνήσετε με τους πολίτες. Εκείνοι θα έχουν επιρροή στην συμπεριφορά του πώς θα ψηφίσουν, ψηφίσουμε, όχι μόνο εμείς αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια. Και αυτό όχι για την TTIP μόνο ζήτημα, αλλά για όλα τα άλλα εγχειρήματα και προγράμματα και σχέδια που έχετε, που εμείς θα συνεργαστούμε για αυτά τα επόμενα χρόνια και θα συζητήσουμε για αυτά. Αλλά ευχαριστώ για τον ανοιχτό χαρακτήρα, την ευθύτητα και τη διαφάνεια από πλευρά σας. Δεύτερον, είμαι ίσως η μόνη, αλλά είμαι υπέρ του ότι το ISDS πρέπει να δημιουργηθεί, να ε, εγκριθεί με μια τροποποιημένη μορφή δεν είμαι μόνη μου με αυτές τις απόψεις, ακόμα και αν οι αντίπαλοι έχουν ισχυρότερη φωνή από τη δική μου. Ευχαριστώ. Sorry. Um, I was listening to, to... Συγγνώμη, άκουγα τη δερμηνία, ε, κυρία Κιρτον Τάρλινγκ. Μας ικανοποιεί που λέτε ότι θα κάνετε μια νέα αρχή. Θα ήθελα να συμφωνήσω με πολλά από τα όσα είπε η συνάδελφος η κυρία Ρέντινγκ. Μια από τις βασικές μου ανησυχίε ε, καθώς εστιάζουμε όλη την προσοχή στην TTIP, ένα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι διαπραγματεύσεις ε, έχουν γίνει λίγο υπόγεια και η πιθανή συμφωνία teaser θα παίξει το ίδιο σημαντικό ρόλο όσο και η TTIP σε τελική ανάλυση. Θα θέλαμε λοιπόν να δοθεί η ίδια διαφάνεια και στην συμφωνία ΤΙΖΑ όπως και στην ΤΙΤΙΠ. Ένα βασικό ζήτημα τώρα οι δημόσιες υπηρεσίες για να πάρουμε τον κόσμο με το μέρος μας όσον αφορά αυτές τις διαπραγματεύσεις πρέπει να έχουμε απόλυτη σαφήνεια για το τι, είναι, τι έχει συμφωνηθεί εσωτερικά και εξωτερικά δηλαδή να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις προσφορές της Ευρώπης ε, στην ΤΙΖΑ, στην ΤΙΤΙΠ και σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία. Ευχαριστώ κύριε Στιτόσο. Τέμοζα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα ε, κύριε Επίτροπε ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει περίπτωση να επανεξετάσουμε την προσφυγή μας για την ε, συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Εγώ σας συνιστώ να μην προσφύγετε στο δικαστήριο διότι Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τα διάφορα αρχεία τα οποία υπάρχουν και με τη Σιγκαπούρη ε, και άλλες ασιατικές χώρες. Ε, κυρία Μινέρ, κυρία Μάλμστρομ, υποσχεθήκατε διαφάνεια και εμείς ε, καλωσορίζουμε αυτή τη βελτίωση. Ωστόσο, αυτέ οι συμφωνίε ελευθερών συναλλαγών έχουν τόσο τεράστιε επιπτώσει στι ζωέ των Ευρωπαίων πολιτών που χρειαζόμαστε κάποια καλύτερη προσπάθεια ώστε αυτή η συζήτηση να γίνει δημόσια πού πάμε με αυτή την Ήπειρο. Δημιουργούμε μια τεράστια νέα εσωτερική αγορά που θα έχει τεράστιες επιρροές για τα ε, δικαιώματα των εργαζομένων, τις υπηρεσίες που παρέχονται τα προϊόντα. Πριν από τη συνάντηση άκουσα τον ε, κύριο διαπραγματευτή σας, τον Μάριο Πετροτσόνα, να μιλάει για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και τι κρίμα θα ήταν τα Εθνικά Κοινοβούλια να έχουν, να έχουν να πούν κάτι για τη συμφωνία με τον Καναδά, διότι μπορεί να διτεθούν. Και καταλαβαίνω τις ανησυχίες του, γιατί η αντίθεση προς το ISDS ε, όλο ένα και αυξάνεται. Από τα γερμανικά συνδικάτα, η Γαλλία επικρίνει όλο και περισσότερο το ζήτημα αυτό και το δικό μας Εθνικό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει δύο ψηφίσματα για το ISDS και τη διαφάνεια το να προωθούμε αυτές τις συμφωνίες ε, και το ISDS ε, δεν είναι λύση, απλά διευρύνει το χάσμα μεταξύ της πολιτικής ελίτ και του κοινού. Στις ε, κάτω έχουμε το Brady Match Happily και Discussion, μια ευρεία κοινωνική συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια στις ε, κατοχώρες. Κάναμε ένα δημοψήφισμα συνταγματικό όπως γνωρίζετε. Μπορούμε να το κάνουμε. Χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Απλά οι άνθρωποι με τους οποίους συζητάτε δεν είναι όλοι με τους οποίους πρέπει να συζητήσετε. Θέλουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη οικονομία ή να ακούσουμε τους ανθρώπους και να δούμε τι λένε. Θέλω τις απόψεις σας. Μαρία, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Υπάρχει κάποιο χάσμα σε σχέση με το παρελθόν. Ο κύριος ε, Ντεχούχτ ε, δεν μας είχε συνηθίσει να συζητάμε σε διαφάνεια, αλλά δεν μπορεί η διαφάνεια να είναι μόνο marketing. Έχω μια απλή ερώτηση. Το ελεκτικό συνέδριο σήμερα το πρωί μας έδειξε την έκθεση, μας προσέσε την έκθεση για τις ε, μελέτες αντικτύπου και ζήτησε να εμβαθύνονται αυτές, ε, να δημοσιοποιούνται, να επικρίνονται και να γίνονται με τη συνεργασία της Eurostat. Είστε έτοιμοι να αλλάξετε αυτές ε, τις μελέτες αντικτύπου, όχι μόνο για την TTIP, αλλά για το σύνολο των συμφωνιών που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Το δεύτερο που θέλω να πω, χθε στο πλαίσιο της ακρόασης για την απασχόληση στο πλαίσιο της TTIP, συζητήσαμε διάφορα όπως τα κοινωνικά δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά δικαιώματα. Επ' αυτού Είστε έτοιμοι και ο συνάδελφός μου Γιάννη Ξαντώ το ρώτησε. Είστε διατεθειμένοι να υιοθετήσετε μια δεσμευτική ε, πορεία όσον αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα. Και τέλος, σε σχέση με το όμως μας είπε το ηλεκτρικό συνέδριο σήμερα το πρωί, παρατηρούμε την ανικανότητα της Κομισιόν αυτή τη στιγμή να υλοποιήσει έναν αποτελεσματικό έλεγχο για τα αγαθά στο πλαίσιο των ελευθερών συναλλαγών. Έχετε τέτοια πληροφορία και αν ναι, πώς η Κομισιόν θα υλοποιήσει τον έλεγχο για το να έχουμε συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών χωρίς δυνατότητα ελέγχου δεν είναι κάτι ιδιαίτερα αποτελεσματικό θεωρώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Σίλβα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Δεν μπορώ παρά να διακρίνω ως εισηγητής για τη συμφωνία με την Ιαπωνία ότι η κυρία Επίτροπος στην παρουσίασή της στην αρχική αναφέρθηκε στην Ιαπωνία αμέσως μετά την ε, ITTIP και συμμερίζομαι την αξιολόγηση αυτής της συμφωνίας που είναι λοιπόν πολύ αξιόλογη από οικονομικό, υπό πρίσμα και στρατηγική. Και σημειώνω την αισιοδοξία σας επίσης γιατί είπατε ότι είναι πιθανό να ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις του χρόνου 2015. Παρότι υπάρχει αβεβαιότητα πολιτική στην Ιαπωνία με εκλογές που θα γίνουν εσπεσμένα. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρόοδος που επετεύχθη από την ε, Ιαπωνία για την άρση των μη δασμολογικών ε, ε, φραγμών δεν είναι το τέρμα της διαδρομής και ότι υπάρχουν και άλλα κρίσιμα θέματα που πρέπει να επιληθούν για μια ισόρροπη συμφωνία. Μπορείτε να μας πείτε τους τομείς εκείνοι ποιοι είναι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί και έχει απαιτήσει διαπραγματευτικά επ' αυτών ή αν θεωρεί ότι σε αυτούς τους ευαίσθητους τομείς αυτοκινητοβιομηχανία, αγροτροφικός τομέας για παράδειγμα αν είναι δυνατόν να επιτεθεί σε μια τόσο σύντομη χρονική περίοδο η ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάιφριντ, ίσως θα έπρεπε να αποχωρήσω, να ζητώ συγγνώμη. Κάπως έχω οργιστεί πρέπει να πω, λέει ο κύριος Λάιφριντ. Έχω εμπλακεί στην TTIP, στην ΣΕΤΑ με τον Καναδά και όλο τον πολιτικό μου βίο με άλλες πολιτικές συμφωνίες στην Ευρωβουλή. Όμως σε σχέση με το θέμα της ε, διαφάνειας ε, που ε, δεν είμαι σε σχέση με τη διαφάνεια υπεύθυνο της ομάδας μας για αυτά τα θέματα όμως άκουσα με ιδιαίτερη χαρά ότι θα είναι όλα λέει διαφανή, όλα θα είναι καλύτερα και θα επιτευχθεί η διαφάνεια και είπα ορίστε τι γίνεται πήρα ένα email, ένα μήνυμα και είναι η βοηθός μου που μου λέει ότι λυπούμε αλλά μπορεί να μην δοθεί μια θετική απάντηση στο έτοιμά σας και γι' αυτό δεν θα είναι δυνατόν να έχει πρόσβαση ο κύριος Λάιχτφριντ σε αυτά τα έγγραφα. Τι είναι αυτό, αυτό είναι διαφάνεια. Μήπως είναι γραφειοκρατική επιβάρυνση που δεν ξέρουν ε, οι γραφειοκράτες τι επιθυμούν οι υπεύθυνοι διοικητικά ηγέτες τους. Δεν το ξέρω τι είναι, αλλά πείτε μας τι είναι. Είναι αυτό διαφάνεια, αν λέτε εσείς, ε τότε μην κάνουμε λόγο. Να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται έτσι. Δεν είναι ακριβώς καθόλου τόσο διάφανα τα πράγματα αν συνεχίζουν έτσι. Ευχαριστώ. Και θα ξαναδοκιμάσω αύριο να δούμε μήπως βελτιωθούν τα πράγματα. Πάρω καλύτερη απάντηση. Εσείς παρακαλώ. Yeah, Κάποιες παρατηρήσεις και ερωτήματα. Ήμουνα καθηγητής πανεπιστημίου ε, στο ε, ε, πανεπιστήμιο. Είδα τα ερωτήματα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και τα συνέκρινα αυτά με τη συζήτηση και τα ερωτήματα και τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν εδώ. Αν υπολογίσω τις φοβίες, φόβους, ε, επιφυλάξεις, προγνώσεις, ε, ποτέ δεν θα είχαμε καταλήξει στην οικονομική κοινότητα, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Να το πούμε αυτό. Αυτοί οι φόβοι που διατυπώνονται και τότε ήταν ισχυροί στο παρελθόν δεν ήταν τίποτα καινούργιο. Και όμως παρόλα αυτά δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και αυτό το θυμόμαστε. Και μετά γίνεται εδώ λόγος για θυσίες. Ακούω ποσοτικές αναλύσεις για την TTIP. Κανείς δεν μπορεί να ποσοτικοποιήσει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του TTIP. Γιατί όλα αυτά εξαρτώνται από τις συνθήκες πλαίσιο. Κάθε μεγαλύτερη αγορά δίνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Μεγαλύτερη παραγωγικότητα οδηγεί σε απώλειες. Κλείνουν επιχειρήσεις, χρεοκοπούν. Τι να κάνουμε. Και αυτό είναι στη ζωή. Ποιε συνοδευτικέ πολιτικές θα κάνω εγώ, ώστε από την TTIP να ε, υπάρξει επιτυχές αποτέλεσμα, να στεφθεί με επιτυχία. Αν δεν κάνει κανείς τίποτα και δεν επενδύσει στην κατάρτιση, στην εκπαίδευση, σε όλα αυτά, τότε θα είναι απώλεια η TTIP. Αν έχουμε ανοιχτό πνεύμα προσέγγιση στην TTIP και δράσουμε ενεργά, τότε θα στεφτεί με επιτυχία. Όταν κάνετε λόγο για θυσίες και θύματα, να θυμόσαστε ότι τα συνοδευτικά μέτρα για τέτοιες συμφωνίες είναι αταποφασιστικά. Ο Παύλο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί Επίτρεπε, θα ήθελα να μιλήσω μόνιμο ε, επιτροπο, ε, ε, εισηγητής για τη συμφωνία με το Μερκοσούρ. Να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με αυτή τη σημαντική συμφωνία με το Μερκοσούρ. Θα ήθελα επίσης από πλευρά σας να μας δώσετε μια αξιολόγηση αξιολόγηση για τις ε, πρόσφατες εκλογές που έγιναν στην Ουρουγουάη και στη Βραζιλία. Πιστεύετε ότι βοηθούν να προχωρήσουν, να προαχθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις που παρατάθηκαν περισσότερο από ό,τι είχατε υπολογίσει ή ποια είναι η αξιολόγησή σας. Μήπως είναι αντίθετη. Ναι, Επίσης θα μας πείτε την ε, δική σας θέση για τον εξυγχρονισμό της συμφωνίας με τη Χιλή. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Σας ευχαριστώ. Εσείς παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ και για την επίσκεψή σας εδώ που μας επισκεφθήκατε στην ε, Επιτροπή Ίντα και σε σχέση με τα όσα είπατε για το Ευρωκοινοβούλιο θέλω να αναφέρω το θέμα της διαφάνειας και σε σχέση με την ανακοίνωση που μας απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέγνωσα πολύ προσεκτικά το έγγραφο και ανέμενα κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτή η ανακοίνωση δείχνει ότι υπάρχουν κάποιοι φόβοι από πλευρά της Επιτροπής για την ΑΚΤΑ τέθηκε το ζήτημα διαφάνεια το 2012 και θεωρώ ότι αυτή η ανακοίνωση στην πραγματικότητα, με αυτή την ανακοίνωση υπόσχεστε μεγαλύτερη διαφάνεια. Ε, είναι σαν να προσπαθείτε να τραβήξετε την προσοχή μας σε κάτι πέρα από αυτή τη συμφωνία. Τα μυστικά έγγραφα ούτω ή άλλω δεν πρόκειται να βγουν από τα θεσμικά όργανα, δεν θα μπορέσουν να διανεμηθούν χωρί τη Συμφωνία των ΗΠΑ και η διαφάνεια είναι λίγο μισή, αν μου επιτρέπετε. Θα ισχύει για τις συνεδριάσεις των επιτρόπων ίσως, αλλά όχι για τις συνεδριάσεις των υπαλλήλων της Digitrade με τους λομπίστες. Ε. Και μην ξεχνάμε ότι η διαφάνεια δεν είναι το μόνο πρόβλημα της TTIP. Κάτι τελευταίο, στο κείμενο διάβασα ότι αντικείμενο του ίδιου του κειμένου είναι να επιτευχθεί η συνένεση των πολιτών για την TTIP. Εγώ θεωρώ ότι δικό σας καθήκον ως θεσμικών οργάνων είναι να ενημερώνετε τους ε, πολίτες και όχι να τους πείθετε. Φραν Σάντσες. Ευχαριστώ. Να δούμε αυτή τη μελέτη της, του Πανεπιστημίου Ταφτς στις ΗΠΑ μια και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η μελέτη, μια και βασίζεται στο πρότυπο των Ηνωμένων Εθνών για την παγκοσμιοποιημένη πολιτική. Είναι το πιο αντικειμενικό έγγραφο από όσα έχουμε μέχρι σήμερα. Θα ήθελα να μου πείτε, με αυτά τα στοιχεία που είναι τόσο απογοητευτικά, τα οποία προσφέρονται, δεν θα έπρεπε κάτι να επανεξετάσετε σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις της ε, TTIP. Δεύτερη ερώτηση δρατώμενη της ευκαιρίας ε, της παρουσίας στην αίθουσα των μη κυβερνητικών οργανώσεων που αγωνίζονται για τα κράτη της Αφρικής. Θέλω να ξέρω, θα συνεχίσει να πιέζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρξει πρόοδος ε, σε σχέση με αυτά τα θέματα για αυτές τις χώρες. Και τελευταία ερώτηση για την εμβέλεια και το, ε, τη σημασία των ορικτών. Ε, είσαστε πρόθυμοι να υιοθετήσετε μια θέση που θα δεσμεύεται ώστε να υπάρχουν δεσμευτικές υποχρεώσεις ευχαριστώ. Yes, thank you. Ε, ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη στον κύριο Ζαντό. Δεν μπόρεσα να ακούσω όλη την ερώτησή σας. Σήμερα μιλώντας στον Μάρτιν, είπα ότι υπάρχει ε, GSP Plus και θέλουμε όλες οι ε, συμφωνίες ελευθερών βορείου στο μέλλον να έχουν κεφάλαια βιος, ε, βιωσιμότητας, αηφορίας για την εργασία και το περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, ανάλογα με το ποια, για ποια χώρα πρόκειται, θέλουμε να έχουμε και σωστή επιτήρηση. Το ζητήσαμε και για τις Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά ε, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς. Πολλές χώρες του κόσμου, κυρίως σε χώρες που δεν είναι πλήρης δημοκρατίας ή και χειρότερα, έχουμε ξεκινήσει ένα διάλογο είτε για ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε, ε, κάνουμε προσπάθειες και για άλλες ε, συμφωνίες σύνδεσης και θέλουμε το εμπόριο να μπει πιο ολοκληρωμένα στη γενική εξωτερική πολιτική και γι' αυτό συνεργάζομαι με την κυρία Μολγκερίνη ώστε το εμπόριο να αποτελέσει σημαντικό σκέλος της εξωτερικής πολιτικής ώστε να έχουμε διαρκή διάλογο. Οι εμπορικές συμφωνίες είναι ένας, μόνο τρόπος αξιολόγησης. Δεν μπορεί να αλλάξει ε, θεμελιωδώς η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μόνο μέσω του εμπορίου. Είναι ένα κομμάτι του πάζελ. Να δούμε πώς μπορούμε να εμπλακούμε με τα κράτη-μέλη και την κοινωνία των πολιτών, διεθνεί οργανισμού όπως ε, το Διεθνές Γραφείο και άλλους για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια είναι τα προβλήματά μας για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με ένα σύστημα και με διαφανή και υποχρεωτικό τρόπο. Να μην αρχίσουμε τις αναστολές αυτός νομίζω ότι είναι ένας τρόπος που συμπεριλαμβάνει, λαμβάνει υπόψη του και τα συμφέροντα των ανθρώπων που υποφέρουν. Φυσικά απαιτείται διαρκής επιτήρηση και αυτό θα συζητηθεί σε μελλοντικά έγγραφα. Πώς μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερο στην αηφορία μέσω του εμπορίου. Κυρία Λεπέν, χωρίς να ξεκινήσω, να εισέλθω στη συζήτηση που ξεκινήσατε με τον κύριο Πρόεδρο, πρέπει να σας πω ότι θα έχετε πρόσβαση σε περισσότερα έγγραφα μέσω διαδικτύου για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, όπως επίσης και σε όλα τα έγγραφα που, στο, στα οποία το, στο παρελθόν πρόσβαση είχε ένας πολύ μικρός αριθμός ευρωβουλευτών, θα είναι προσβάσιμα σε όλους από εδώ και στο εξή. Φυσικά πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για να λειτουργήσει το σύστημα, για να δούμε μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Εν πάση περιπτώσει αυτό θα είναι ένας τρόπος για να σας δείξουμε εσάς και στους ε, εκλογείς σας, στους ψηφοφόρους σας και στους πολίτες τους οποίους εκπροσωπείτε τι ακριβώς συζητείτε και τι δεν συζητείτε. Και φυσικά θα υπάρξουν και τακτικές αναφορές για την προόδο των διαπραγματεύσεων ώστε να εξασφαλιστεί ότι τελικά η συμφωνία αυτή ε, θα είναι συμφωνία που μπορεί να εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κράτη-μέλη και γι' αυτό απαιτείται διαφάνεια. Η διαφάνεια δεν είναι μόνο στα λόγια, είναι κάτι που οδηγεί σε ένα διάλογο, μια ανακοίνωση που πολλοί από εσά αναφέρθηκαν. Ε, ένας διάλογος με τους πολίτες. Και εγώ δεν ζω μόνο ε, σε αυτή τη φούσκα. Ε, πολύ συχνά έρχομαι σε επαφή με τους πολίτες πολλών χωρών αφού με τις ανησυχίες τους και προσπαθώ να τις ακούσω είτε σε προσωπικό επίπεδο και συμφωνώ απολύτως μαζί με εσά και με πολλούς άλλους συναδέλφους ότι χρειάζεται ανακοινώσεις, όχι μόνο ενημέρωση αλλά και επικοινωνία με τους πολίτες, όχι μόνο για τη Συμφωνία για τις ΗΠΑ αλλά και με άλλες χώρες και σε άλλους τομείς. Κυρία Ρέντινγκ, όσον αφορά τη ΤΙΣΑ, ναι, δεν είναι δημόσια η εντολή. Ελπίζω να μπορέσει να γίνει. Δεσμεύτηκα ε, με τους υπουργού Εμπορίου για θέματα ε, διαφάνειας πριν από μία εβδομάδα. Υποστήριξαν την πρωτοβουλία και αναγνώρισαν ότι όχι μόνο στην TTIP αλλά και γενικότερα στο εμπόριο χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια αλλαγή νοοτροπίας και ελπίζω θα καταφέρουμε να ε, δημοσιεύσουμε την εντολή. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Πάρα πολλά έγγραφα της συμφωνία αυτής είναι δημόσια αλλά όχι η εντολή. Όσον αφορά το συγκεκριμένο, συγκεκριμένο αφορά στην προστασία των δεδομένων, το έγγραφο έχει κυκλοφορήσει. Τα περισσότερα κράτη-μέλη ε, έχουν σχολιάσει. Για μα είναι απόλυτα σαφή ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε οτιδήποτε που θα διακινδυνεύσει την προστασία στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει η Συμφωνία Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που ξέρετε ότι έχουμε συμφωνήσει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα επισέλθουμε σε καμία συζήτηση που θα διακινδυνεύσει τα προσωπικά δεδομένα στην ΤΙΖΑ. Αυτό το σημειώνουμε, αλλά νομίζω ότι κανένας δεν θέλει να εμπλακεί σε κάτι τέτοιο. Όσον αφορά την Κίνα, βεβαίως είναι σημαντικός εταίρος. Δύσκολος εταίρος, αλλά σημαντικός και αναφέρθηκα σε αυτήν όταν είπα ότι πρέπει κάπως να σκεφτούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις αναδυόμενες αυτές οικονομίες και σαφώς η Κίνα είναι μία από αυτές. Όσον αφορά τις συμφωνία για τις επενδύσεις προχωρούμε, όμως δεν έχει κλείσει. Αποτελεί προτεραιότητα. Προσπαθούμε να ανοίξουμε λίγο την αγορά τους σε ευρωπαϊκές επενδύσεις και στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Και όταν συμβεί αυτό μπορούμε να μελετήσουμε το πώς θα προχωρήσουμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς να ξεκινήσουμε συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Κίνα. Πρέπει πρώτα να γίνει η συμφωνία ε, επενδύσεων για να αυξήσουμε την πρόσβαση που έχουμε στην αγορά. Για την Ταϊβάν, επίσης σημαντικός εταίρος, έχουμε επαφές μαζί τους μέσω της ΤΙΖΑ και της ΙΤΑ ε, την περασμένη εβδομάδα νομίζω είχαμε ένα σεμινάριο για τον τομέα των υπηρεσιών και το πώς μπορούμε να ε, συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Έχουμε τακτικές επαφές για, και συζητήσεις για τα εμπόδια στο εμπόριο κλπ. Ε, αυτά τα διερευνούμε και προσπαθούμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Να δούμε μέχρι που θα πάμε προς το παρόν. Είναι ε, διαρκής εταίρος με τακτικό διάλογο. Ινδία. Ο κύριος Κάμπος ρώτησε για την Ινδία, ναι. Ε, όπως γνωρίζετε είχαν γίνει συζητήσει επί πολλά χρόνια, είχαν όμως παγώσει τα τελευταία χρόνια, που δεν, όχι για λόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν επιλογή της Ινδίας. Για τον λόγο αυτό δεν είχαμε θεωρήσει απαραίτητο πέρυσι να, ξεκινήσουμε, να στήσουμε μια πλήρη διαπραγματευτική ομάδα. Αν τώρα μοιάζει ότι θέλουν να επανέλθουν και στη συζήτηση μαζί μας, θα δούμε πώς θα οργανωθούν οι διαπραγματευτικές μας ομάδες. Αλλά προς το παρόν, αφού δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις εν εξελίξη, δεν είναι θέμα που μας έχει απασχολήσει. Όμως θα είναι απολύτως ευπρόσδεκτο όταν αν ε, δώσουν ενδείξει ότι θέλουν να επανέλθουν. Τώρα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει ειδικό κεφάλαιο στην TTIP και ε, θεωρώ ότι πρέπει σαφώς να ξεκαθαρίσουμε πώς μπορούμε να ε, συνεισφέρουμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να εφαρμόσουμε ρήτρες που θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς μπορούμε να ε, βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τις ε, δυνατότητες που προσφέρουν οι εμπορικές συμφωνίες, ας πούμε με την Κορέα, για την Κίνα. Επίσης, καθεστώς οικονομίας αγοράς. Δεν... Αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να θέσω τον Ιανουάριο σε ψηλή προτεραιότητα με τους άλλους συναδέλφους της Κομισιόν για να το συζητήσουμε. Υπάρχουν κριτήρια, τεχνικά κριτήρια, τα οποία δεν έχουν ε, τηρηθεί ακόμα, δεν εκτηρούνται και πρέπει στην Επιτροπή να συζητήσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα και θα επανέλθουμε στη συζήτηση μαζί σας. Τώρα, ε, τα Trade Defensive Instruments στο Συμβούλιο και την, ε, την προηγούμενη εβδομάδα έδειξε ότι υπάρχει πλήρης, πλήρες αδιέξοδο μισή-μισή. Ε, Η Ιταλική Προεδρία έκανε ηρωική προσπάθεια να ξεμπλοκάρει, αλλά δεν, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο, τους είπα, να έρθει στον τριμερή διάλογο, τίποτα. Σήμερα συνομίλησα με τους εκπροσώπους της επερχόμενης Λετωνικής Προεδρίας. Ε, μας είπαν ότι θα κάνουν ότι μπορούν να ξεμπλοκάρουν την κατάσταση, αλλά είναι πολύ μπερδεμένο. Αν έχετε κάποια ιδέα για το πώς μπορεί να ε, ξεμπλοκαριστεί το θέμα, ευπρόσδεκτη. Ε, Σιγκαπούρη. Εσείς, ναι. Σημείωσα. Ε, τη διαπραγματευτήκαμε ως μία συμφωνία. Εάν τώρα την διαχωρίσουμε στα δύο, θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να τεθεί ενισχύ, γιατί δεν τη διαπραγματευτήκαμε έτσι. Και δεν θέλουμε να προχωρήσουμε έτσι σε αυτό το τομέα. Θέλουμε να έχουμε μια φιλόδοξη συνολική ατζέντα για αυτά. Θα ήταν λοιπόν ατυχές να, ε, να ξεχωρίσουμε το επενδυτικό σκέλος. Γνωρίζω όμως την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από αυτού. Το εμπόριο από τη Λισαβόνα στο Βλαδιβοστόκ και εγώ το διάβασα. Πολύ ωραίο όραμα. Ωραίο όραμα αλλά δεν νομίζω ότι είναι ένα όραμα που θα το δούμε να υλοποιείται σύντομα. Πρώτον, συζητούμε με τη Ρωσία και χωρίς να σας ε, αναφέρω τις λεπτομέρειες, η Ρωσία έχει καταλάβει ε, μέρος μιας ανεξάρτητης χώρας, εκεί κλιμακώνονται τα πράγματα, άρα το να ξεκινήσουμε εμπορικές συμφωνίες ε, δεν θεωρούμε ότι είναι κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο. Αλλά και πιο πρακτικά μιλώντας, ε, δεν έχει ξεκινήσει, ή δεν έχει ενταχθεί στον, στον ΠΟΕ και δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Υπάρχουν πράγματα ε, που γίνονται και τα οποία επηρεάζουν ε, σημαντικά την ευρωπαϊκή οικονομία. Η οικονομία δεν είναι εύκολος εταίρος. Ξέρω ότι στο μέλλον μπορεί κάτι να συμβεί, είναι ένα ωραίο το όραμα, αλλά προς το παρόν δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Τώρα, όσον αφορά την ε, κρίση, την, του δικαστηρίου, ναι, η Κομισιόν διάβασε το έγγραφο. Κάποιες από τις μεθόδους ήδη άλλαξαν, ήταν λίγο ξεπερασμένες, ήδη άλλαξαν κάποιες μέθοδοι, αλλά ήδη προσπαθούμε πώς θα πάρουμε υπόψη μας αυτές τις, ε, ε, αυτές τις παρατηρήσεις για να συνεχίσει η παρακολούθηση αυτών των συμφωνιών. Η Ευρασία, ναι, νομίζω το... Ε, ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία, νομίζω το ανέφερα αυτό. ISDS. ISDS. Ε, υπάρχει αυτό το σκέλος στην συμφωνία με τον Καναδά. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο να αντιμετωπίσουμε το SDS στην, στην, στην ε, συμφωνία με τον Καναδά αποτελεί σοβαρή βελτίωση στον τρόπο που λειτουργεί τώρα. Αυτό υπάρχει επιτάπητος και δεν πρόκειται να χαλάσει. Αυτό που συμβαίνει στην TTIP είναι ότι υπάρχει αυτή η διαβούλευση, όπως είπα ευθύς εξ αρχής. Θα κάνουμε μια ε, περιληπτική παρουσίαση αυτών των διαβουλεύσεων πριν τα Χριστούγεννα και ακόμη θα έχουμε τα αποτελέσματα, την ανάλυση, στις διαφορετικές εναλλακτικέ λύσεις και πώς θα προχωρήσουμε. Γιατί όπως γνωρίζετε τα κράτη-μέλη ε, ε, έχουν ζητήσει να συμμετέχουν συμφωνία θέλουν και οι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά ο κύριο Γιούνκερ ήταν απόλυτα σαφή και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Πρέπει να υπάρξει μια πλήρη μεταρρυθμισμένη ISDS σε σχέση με το, τα όσα ισχύουν τώρα. Και από αυτό έχουμε δουλέψει. Γενικά για την TTIP. Επίκυνται διάφορες μελέτες. Ε, γνωρίζω τη μελέτη στην οποία αναφερθήκατε. Χρησιμοποιεί διαφορετική μεθοδολογία. Βεβαίως, δεν είναι ομόφωνα όλα τα κράτη-μέλη με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το ψήφισμα του 2012 που λέει ότι η μάλλον δεν θα υπήρχε όλη αυτή η συμφωνία αν δεν ήταν κάτι καλό αυτό. Επί, ώρες επί ωρών διαπραγματεύσεων δεν θα, δεν, θα γίνονταν, δεν θα είχαν γίνει αν δεν ήταν κάτι το καλό. Γιατί πιστεύουμε ότι θα μας φέρει θέσεις εργασίας ε, και ανάπτυξη και επενδύσεις. Πολύ περισσότερο από ότι άλλες. Και το να ε, ξεπεράσουμε τους δασμούς, τη γραφειοκρατία και τις επιπλοκές, το άνοιγμα της αγοράς, ιστορικά πάντοτε ήταν εποφέλες. Τώρα διάφορες μελέτες δείχνουν διαφορετικά αποτελέσματα, όμως η συντριπτική πλειοψηφία των μελών δείχνει ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για την Ευρώπη και το πιστεύουμε αυτό και ελπίζω ότι στην επαφή μου μαζί σας και με άλλους και με την κοινωνία των πολιτών θα μπορέσω να πείσω ότι αυτό το οποίο διαπραγματευόμαστε και αυτό το οποίο δεν διαπραγματευόμαστε θα είναι επωφελές για τους πολίτες, τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εν γέννη. Όμως ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο να κάνουμε μια νέα αρχή στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων στις αρχές Φεβρουαρίου με τους Αμερικανούς. Τέλος, για το Μεξικό. Ε, σας ευχαριστώ που μου το θυμήσατε. Μερκοσούρ, Μερκοσούρ. Ποιος ρώτησε? Ναι. Μερκοσούρ οι υπουργοί των, χωρών Μερκοσούρ συμφώνησαν ότι θα κάνουν μια νέα κοινή προσφορά για να αναβιώσουν κάπως τις διαπραγματεύσεις. Είναι ευπρόσδεκτη. Συμφωνήσαμε ότι θα συναντηθούν σύντομα οι επικεφαλής των αντιπροσωπιών για να δουν ποιο θα είναι το επίπεδο των επιθυμιών και κατόπιν μπορούμε να αρχίσουμε. Έχουμε θετικές ενδείξεις και από τη Βραζιλία που είναι και αυτές ευπρόσδεκτες για τη Χιλή παρόμοια προσπάθεια όπως και με το Μεξικό, αλλά δεν έχουν προχωρήσει εξίσου πολύ ακόμα. Η συμφωνία με τη Χιλή πρέπει και αυτή να επικαιροποιηθεί. Γίνεται ανταλλαγή επιστολών και συζητήσεις για το πού βρισκόμαστε, ποιο επίπεδο θέλουμε να φτάσουμε, πού θέλουμε, τι θέλουμε να πετύχουμε, ένας εξυγχρονισμός δηλαδή σε ανώτερο επίπεδο. Αν διαπιστώσουμε ότι οι στόχοι μας είναι συμβατή και οι φιλοδοξίε μας συμβατέ, θα προχωρήσουμε. Είναι κάτι που θα μου είναι πρόσδεκτο, αλλά και πάλι δεν έχουμε φτάσει ε, ε, εκεί. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο πριν ξεκινήσουμε. Japan, yes. Ε. Λοιπόν, για την Ιαπωνία μάλιστα. Έχουμε κάποια θέματα τα οποία απομένουν ε, με την Ιαπωνία. Δημόσιες προμήθειες, μη ε, δασμολογικά μέτρα, γεωγραφική όρη προέλευσης ε, και θέματα που δεν έχουν επιληθεί ακόμα. Πολλά απομένουν. Είναι όμως μια θετική ατμόσφαιρα επικοδομητικού χαρακτήρα και έχουν δεσμευτεί για να προχωρήσουμε. Ξέρω ότι θα έχουμε εκλογές στην Ιαπωνία, α, το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε ποια θα είναι η έκβαση, αν θα υπάρξει αλλαγή κυβέρνηση και διαπραγματευτών. Θα πρέπει να αναμείνουμε να δούμε. Αν όχι όμω και δεν υπάρξουν αλλαγέ και συνεχίσει η ομάδα όπω είχε στην σύνθεσή τη, θα συνεχίσουμε κι εμεί τι διαπραγματεύσει. Το περιεχόμενο η ουσία είναι πιο σημαντική από τη χρονική στιγμή που θα γίνουν οι διαπραγματεύσει. Κατά τα τέλη του 2015 ή αρχέ 2016 ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Θα επανέλθουμε με έκθεση όταν θα έχουμε προχωρήσει χωρίς Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο η παρέμβαση. Νομίζω το ανέφερα προηγούμενα. Είπα ότι δεν είναι αυτόματη η διαδικασία. Έχουμε κάποια κριτήρια τα οποία δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί, δεν έχουν επιτευχθεί και θα αρχίσει κατά την έναρξη του ε, επόμενου έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητά αυτά τα θέματα. Θα υπάρξει ξεχωριστή απόφαση γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σε, ευχαριστούμε Σεσίλια και πράγματι ο Χάμφρι Μπόγκαρ ως Ρίκ στην Καζαμπλάνκα πράγματι είπε είναι η αρχή μιας υπέροχης φιλίας αυτή. Και τι ωραία εποχή συνεργασίας μεταξύ μας. Ελπίζω ότι θα προσέρθει στην δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή αρκετές φορές στο μέλλον. Σε ευχαριστώ και θα σε ξαναδούμε σύντομα. Γεια. παρακαλώ. Συνεχίζουμε με τις εργασίες μας. Ο κύριος Λάιχτφριντ, διαδικαστικό παρακαλώ εσείς. Mr. President, thank you very much. So... Uh, ευχαριστώ. Έχω την εντύπωση που αποκόμισα ότι η Επίτροπος δεν ε, αισθάνεται την υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση ε, που επικρατεί εδώ. Ορθό αυτό, έστω. Λοιπόν, θέλω να ξαναθέσω το ζήτημα. Πότε θα είναι δυνατόν επιτέλους ε, να έχουμε πρόσβαση σε αυτή την αίθουσα για να συμβουλευτούμε αυτά τα έγγραφα, τα διαβαθμισμένα. Και θα ήθελα να προαναγγείλω και να πω αύριο θέλω να πάω 10 η ώρα το πρωί εκεί. Λοιπόν, να είστε εκεί να δούμε τι θα συμβεί. Θα έχουμε πρόσβαση ή όχι. Πρόεδρος, λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, ε, φυσικά αυτό είναι ε, σοβαρό ερώτημα, σοβαρό ζήτημα. Και σήμερα διεξοδικά σε σχέση με τους συντονιστές καλύψαμε το θέμα για τις διαπραγματεύσεις για τη διαφάνεια και αναφέρθηκαν διεξοδικά στοιχεία εκεί. Τώρα να τα επαναλάβουμε αυτά. Ωραία. Αφενός λοιπόν πρόκειται για το εξής. Διότι τα, ότι τα έγγραφα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις, μια και έχουν υποβληθεί στις ΗΠΑ, τότε θα δημοσιευθούν, θα δημοσιοποιηθούν. Μας είπαν. Αυτή είναι η δέσμευση που δόθηκε. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές προσαρμογές. Από την 1η Πρώτου 2015 όμως, όταν αυτά τα έγγραφα θα έχουν κατατεθεί όλα στις ε, ενώπιον των ΙΠΑ, τότε θα είναι δυνατόν να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Δεύτερον, θέλουμε να διασφαλίσουμε και αυτό πάντα ήταν το αίτημα του Ευρωκοινοβουλίου, η διεκδίκησή του. Όλοι οι Ευρωβουλευτές θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα. Εντάξει, Μέχρι σήμερα η παλαιότερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αρνηθεί κάθετα αυτό το αίτημα και είχε διαφοροποιήσει μεταξύ κάποιων λίγων ευρωβουλευτών που θα είχαν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, αυτή τη στιγμή είναι 13 αυτοί οι ευρωβουλευτές και, και κάποιοι άλλοι ευρωβουλευτές που αναπερίπτωση εκ αν οι αρμοδιότητες τους καλύπτουν τέτοιου είδους έγγραφα θα είχαν πρόσβαση σε αυτά. Σύνολο δηλαδή 28 και τώρα πρέπει να δούμε η, η μετάβαση, η γεφυροποίηση πώς θα διοργανωθεί. Δεν γίνεται και είναι αθέμητο πιστεύω η γραμματεία μας όπως μέχρι σήμερα τα έγγραφα αυτά να τα προετοιμάζει σε έντυπη μορφή για να είναι διαθέσιμα σε όλους τους 751 ευρωβουλευτές. Δεν γίνεται αυτό, είναι ανέφικτο. Ένα πρώτο βήμα πρέπει να διοργανωθεί ταχύτατα και μετά να υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα κάθε ευρωβουλευτής. Πρώτο έτοιμά μας να πούμε, όχι μόνο αυτοί οι 28 ευρωβουλευτές θα έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα, αλλά όλα τα μέλη της Επιτροπής ΕΝΤΑ, ΙΝΤΑ θα έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά τα έγγραφα οι συν, εμπλεκόμενες συναρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές θα έχουν και εκείνες πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα. Και έτσι δεν θα υπάρχει κάποιο θέμα τριβής ποιοι θα έχουν πρόσβαση και ποιοι όχι. Μπορούμε αυτό να συμφωνήσουμε επ' αυτού. Και το θέμα του αναγνωστηρίου ή της αίθουσας που έθιξε ο κύριος Λάιχτφριντ έτσι νομίζω επιλύεται. Σε τεχνικές διαπραγματεύσεις είμαστε, διαβουλεύσεις Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι τεχνικές προϋποθέσεις θα επιτευχθούν, να είναι το προσωπικό τα στελέχη εκεί ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί η προσπελασιμότητα. Το αργότερο από 1η Ιανουαρίου 2015 λοιπόν αυτό το πρώτο βήμα, η πρώτη φάση θα έχει επιτευχθεί ώστε κάθε ένας από εσά ευρωβουλευτές της ΙΝΤΑ να έχετε πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα αυτά. Εντάξει πάμε τώρα στο σημείο 11 για να συνεχίσουμε με αυτό δασμολογική, ο υπεύθυνο από το Εκουαδόρ περιμένει να εξετάσουμε αυτό το σημείο για να το παρακολουθήσει. Είναι το ζήτημα της σταθεροποίησης της δασμολογικής δηλαδή κατάστασης για τον Ισημερινό επειδή ο Ισημερινός το Εκουαδόρ θα έχανε το καθεστώς αυτό αυτής της χώρας για αυτές τις συναλλαγές δασμολογικά αλλά όμως ε, θα ενταχθεί στη συμφωνία με το Περού και στο μεσοδιάστημα θα υπάρχει ένα κενό, μία οπή ε, και δεν θα καλύπτεται το Εκουαδόρ και η δασμολογική εισπράξη αυτών των δασμών θα δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό πρότεινε ο εισηγητής Helmut Scholz να βρεθεί μια λύση για να προχωρήσει το θέμα αυτό. Όμως το θέμα είναι περισσότερο νομικού χαρακτήρα. Κατά πόσο δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά εξουσιοδότηση πράξης ε, ή εκτελεστικές πράξεις μπορεί να χρησιμοποιήσει και δόθηκε εντολή στην νομική υπηρεσία του σώματος του Ευρωκοινοβουλίου να μας πει τι συμβαίνει. Και υποστηρίζει σαφώς την άποψη του Ευρωκοινοβουλίου η νομική υπηρεσία. Δηλαδή ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει κατά εξουσιοδότηση πράξη να ε, ε, κατατίθενται και να εγκρίνονται. Δίνω λοιπόν τώρα στον εισηγητή Σόλτ τον λόγο να μας πει τα σχετικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ για την προετοιμασία, στο πω έτσι, ή τις διάφορες παρατηρήσεις που έγιναν, τροπολογίες που κατατέθηκαν στο σχέδιο έκθεσης που κατά τις τελευταίες διαβουλεύσεις που είχαμε εξετάσαμε. Γι' αυτό δεν θα επανεξετάσω και δεν θα ξαναρχίσω την παρουσίαση όλων αυτών των γενικών θεμάτων και γενικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε με αυτό το σχέδιο έκθεσης για αυτή τη ρύθμιση που έχουμε μπροστά μας για τον Ισημερινό, το Εκουαδόρ όσον αφορά δασμολογικές διευκολύνσεις και τελωνιακές ε, ε, διευκολύνσεις. Αυτά πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν και προχωρούμε για το χρονικό διάστημα που πιέζει ήδη έγινε λόγος. Και επανέρχομαι σε αυτό, θέλω να επανέλθω σε αυτό και ευχαριστώ ρητά ότι ο κύριος Υπουργός του Ισημερινού και αντιπροσωπεία του Υπουργείου από τον Ισημερινό τον συνοδεύει και παρίστανται εδώ με πολυάριθμους εκπροσώπους ε, επιχειρησιακών κύκλων επιχειρήσεων και από τον Ισημερινό αλλά και από εισαγωγή ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπορικούς εταίρους από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται σε, αντα... συναλλαγές και συναλλάσσονται με τα προϊόντα αυτά, με το... για τα προϊόντα αυτά με το τον Ισημερινό. Έχουμε σε διάφορα χρονικά σημεία επανειλημμένα συζητήσει το τι σημαίνει αυτό Δηλαδή, ο χρονορίζοντας που έχουμε μπροστά μας για να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη κατάσταση και τις ανάγκες των πολιτών του Ισημερινού και όλους, όλων των εμπλεκομένων stakeholders, αλλά επίσης και για τους πολίτες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους αφορούν αυτά τα προϊόντα που εισάγονται. Ακόμα και ή να το πω διαφορετικά. Συμφωνήσαμε και είπαμε ότι σε αυτή τη συνεδρίαση απόψε θα συζητούσαμε για τις τροπολογίες και για τις συμβιβαστικές τροπολογίες, θα ανταλλάσσαμε απόψεις. Αύριο ήδη θα ψηφίζαμε αυτές τις τροπολογίες. Θα ήθελα να προτείνω στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με την ψηφοφορία, άσχετα ποια θα είναι η έκβαση στο τελικό αποτέλεσμα των ψηφοφοριών, εγώ ως συζητητής παρακαλώ αμέσως, αμέσως να περάσουμε στις επίσημες διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο ώστε αυτό το χρονορίζοντα, αυτή την προθεσμία που υπάρχει να μπορέσουμε να, την καταφέρουμε, να καταφέρουμε να την τηρήσουμε για το, τον Ισημερινό. 1η Ιανουαρίου 2015. Δηλαδή ήδη η κατάσταση εξαίρεσης που ισχύει για το Εκουαδόρ η, η, διευκόλυνση ας το πω έτσι όσον αφορά ίσπραξη τελωνιακών δασμών έχει κάποια οικονομική σημασία και θα πρέπει αμέσως να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή η διευκόλυνση. Με το Συμβούλιο λοιπόν, με την Ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου ήρθα σε επαφή, συζήτησα μαζί τους και είναι πρόθυμοι να οδηγηθούν σε ολοκλήρωση σε πρώτη ανάγνωση μαζί μας. Να υπάρξει δηλαδή συμφωνία μεταξύ μας ώστε ή δυνατόν να έχουμε το τελικό κείμενο στο οποίο θα συμφωνήσουμε και να εγκριθεί και να προχωρήσουμε μετά δηλαδή την ψηφοφορία του Ιανουαρίου να μπορέσουμε το Φεβρουάριο να έχουμε προχωρήσει και να πούμε ότι αυτή θα είναι η ρύθμιση η οποία θα αρχίσει να ισχύει από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Διεξοδικά τα ανέφερα λοιπόν όλα. Σήμερα με την ακρόαση με την κυρία Μάνστρεμ είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και την κατάσταση όσον αφορά την Ανατολική Ευρώπη, την Ανατολή και με τις μειωμένες δασμολογικές, ε, με τις ε, χαμηλές τιμές πετρελαίου και την κατάσταση που είναι μια οικονομία που βασίζεται στα δολάρια, η οικονομία του Εκουαδόρ, καθίστανται πιο ακριβές οι εξαγωγές. Οι εξαγωγές των προϊόντων του Εκουαδόρ παγκόσμια Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Ισημερινό, το Εκουαδόρ, με αυτή τη διευκόλυνση την δασμολογική, αμέσως από την 1η-1η Ιανουαρίου 2015, να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο όσο είναι αναγκαίο μέχρι ότου να ε, ενταχθεί στην συμφωνία με το Περού και στο πλαίσιο των διατάξεων για τη συμφωνία με το Περού. Το αργότερο κάπου έξι μήνες μετά την έναρξη σε ισχύ αυτής της ε, ε, κατεξαίρεση ρύθμισης για το Εκουαδόρ προβλέπεται να γίνει αυτό το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Κανείς δεν γνωρίζει από μας αν αυτό το πλαίσιο, αυτός ο χρονορίζοντας θα τηρηθεί. Αυτό το τι θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2017. Αν δεν τα καταφέρουμε, κανείς δεν το γνωρίζει. Είναι μια κατάσταση που βρίσκεται εκρεμή υπό καθεστώς αβεβαιότητας και αν τροχοπεδηθεί ε, μια τέτοια συμφωνία πάλι θα τεθούν εκ νέου ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν όχι μόνο εδώ σε εμά, αλλά και στο, στον Ισημερινό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις πτυχές και η θέση της Επιτροπής ε, Εμπορίου ήταν η πρακτικότητα, ο πρακτικός χαρακτήρας, ε, η λειτουργικότητα να διασφαλίζεται σε θέματα εμπορίου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να δράσουμε προς το συμφέρον όλων των εμπλεκόμενων και ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει αυτό με τέτοιο τρόπο ώστε οι πολίτες του Ισημερινού και οι πολίτες και των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποφεληθούν. Κατά τούτο λοιπόν επιχειρηματολόγησα εγώ με τις παρατηρήσεις μου σε σχέση με αυτή την, το σχέδιο έκθεσης και είπα ότι το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων πρέπει να τεθεί στο προσκήνιο, να προαχθεί ώστε ταχύτατα να μπορέσουμε εμείς όπως και το Συμβούλιο να είμαστε σε θέση άμεσα να αντιδράσουμε και να λάβουμε μέτρα και να δούμε αν υπάρχουν θέματα παγώματος ή ε, ε, κάποιας ε, οποιασδήποτε καθυστέρησης να ρυθμίζονται με τέτοιου είδους πράξεις Νομίζω και με τους σκιώδεις εισηγητές είχαμε ένα πολύ ζωντανό διάλογο και εργαστήκαμε σε βάθος για να προχωρήσουμε τα πράγματα. Αδειμονώ να δω ποια θα είναι η θέση των σχεδόν εισηγητών και να δούμε αύριο τι θα γίνει στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Έχετε τον λόγο εσείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Φίσα Σαϊσελά Χέλμουτ έγινε μια σε ανάλυση όλων των συμφερόντων που βρίσκονται εδώ ενώπιον μας οικονομικών, πολιτικών, νομικών, και στο τέλος τέλος ε, λάβαμε την απόφαση να υπερψηφίσουμε αυτό το κείμενο το οποίο παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να απορρίψουμε δηλαδή όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Το κάνουμε αυτό για να διευκολύνουμε ταχύτατη έγκριση του κανονισμού που θα επιτρέψει να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της κατάργησης ε, των δασμολογικών προτιμήσεων. Δεν γινόταν διαφορετικά. Πολύ προσεκτικά διάβασα τη γνωμοδότηση των νομικών υπηρεσιών του Ευρωκοινοβουλίου θα μπορούσαν νομικά να δικαιολογήσουν εξουσιοδότηση πράξης ως ένα μέσο για να εφαρμοστεί ο κανονισμός σε περίπτωση φυσικά ε, κατάργησης των δασμολογικών προτιμήσεων. Όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου κατέληξε σε διαφορετικά συμπεράσματα για αυτό το θέμα. Αυτό δείχνει την δυσκολία να καθορίσουμε ποιο είναι το πιο ενδεδειγμένο μέτρο το οποίο θα έπρεπε να υιοθετηθεί σε μια τέτοια περίπτωση. Κάνουμε λόγο για μια προσωρινή ρύθμιση για να αντιμετωπιστεί μια ξεχωριστή κατάσταση. Πολύ ξεχωριστή κατάσταση για μια χώρα που έχει ανάγκη αυτών των προτιμήσεων λαμβάνοντας υπόψη τους εξής παράγοντες. Να υπάρχει μια συνεκτικότητα και συνοχή με παρόμοιους ε, κανονισμούς όπως για το Πακιστάν, την Ουκρανία, τη Μολδαβία, Όλα αυτά τα επιχειρήματα και όλοι αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις και το πιεστικό χρονοδιάγραμμα οδήγησαν την ομάδα μου να υποστηρίξουν κάποιες από τις τροπολογίες του εισηγητή και εν πάση περιπτώσει θέλω να τον, να τον συγχαρώ για την προσπάθεια που κατέβαλε για αυτό το χαρτοφυλάκιο. Στην περίπτωση που έχουμε μπροστά μας υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα πολιτικού και εμπορικού χαρακτήρα που πρέπει να λάβουμε υπόψη η έγκριση κάποιων από τις τροπολογίες από το Ευρωκοινοβούλιο θα οδηγούσε σε μια καθυστέρηση της έγκρισης του κανονισμού κατά δύο μήνες τουλάχιστον. Και θα μπορούσαμε να φτάσουμε και σε τρεις ή τέσσερις μήνες από τα, ε, που θα εξαρτάται αυτό από τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου. Και εδώ τώρα σε σχέση με ε, ε, ε, αναδρομικής εφαρμογής από την 1η Πρώτου του 2015 σε σχέση με τους δασμούς και εδώ έχουμε υπόψη το 24% η αβεβαιότητα σε σχέση με τους τελωνιακούς δασμούς και οι δυσκολίες που θα είχαν οι εισαγωγείς για τα ποσά τα οποία θα είχαν ήδη πληρωθεί θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομία του του Είναι πιθανόν αντί να πληρώσουν το επιπλέον 24% των αγαθών αυτό αυτών οι εισαγωγείς να στραφούν σε άλλε χώρε για να εισαγάγουν τα προϊόντα του. με αποτέλεσμα να ε, ήθελαν ίσως να επιστρέψουν στην ε, αγορά του Ισημερινού μετά την έγκριση του κανονισμού. Σε σχέση με αυτέ τι προτιμήσει, λαμβάνοντα υπόψη ότι τα στοιχεία που προτείνονται στι τροπολογίε δεν αλλάζουν ουσιοδό την πρόταση του κανονισμού η ομάδα μα πιστεύει ότι η καλύτερη βοήθεια για τον Ισημερινό είναι να δουλέψουμε και να υιοθετήσουμε άμεσα την πρόταση κανονισμού. Γι' αυτό θα απορρίψουμε όλες τις τροπολογίες λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ως κοιόδης εισηγητής για τους σοσιαλδημοκράτες λαμβάνω εγώ τον λόγο. Και εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη άμεσα να δράσουμε. Είναι αυτονόητο ότι δεν θέλουμε να υπάρξει κάποιο κενό που θα αφήσουμε να δημιουργηθεί. Από την άλλη πλευρά όμως είναι σαφές επίσης ότι πραγματικά δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιο προηγούμενο εδώ όσον αφορά την απεμπόληση δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό όπως και σε όλα τα άλλα νομοθετικά εγχειρήματα πρέπει να αποσαφηνίσουμε το ότι πάντα τότε όταν υπάρχει θέμα νομοθεσίας πρέπει να απαιτείται ε, λύση κατεξουσιοδότηση πράξεως. Και είχαμε και τον τριμερή διάλογο σε σχέση με τα εξωτερικά στατιστικά στοιχεία, πράγμα το οποίο νομοθετικά, ας το πω έτσι, από πλευράς του έχει και τις, τον ειδικό χαρακτήρα του. Όταν νομοθετούμε όμως τότε το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει με κατεξουσιοδότηση πράξη που πρέπει να υποβάλλεται, να κατατίθεται. Έτσι θα εγκρίνουμε λοιπόν. Αλλά με τη σαφή ένδειξη κύριε Υπουργέ αναφέρθηκε αυτό ότι αν αυτή, αυτό το αίτημα τύχει πλειοψηφικής έγκρισης άμεσα, αμέσως μετά την ψηφοφορία θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις μας, οι διαβουλεύσεις μας με το Συμβούλιο για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει καμία καθυστέρηση χρονική. Αυτά είχα, ήθελα να πω. Έχετε εσείς τώρα τον λόγο πάλι. Παρακαλώ. Uh, thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γενικά η ομάδα του ECR είναι φυσικά υπέρ της πρότασης της Επιτροπής θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να συμπληρωθεί, να καλυφθεί το κενό μεταξύ 1η Ιανουαρίου του 2015 και της χρονικής στιγμής όπου αυτή η νέα FTA, η διευρυμένη FTA θα τεθεί σε ισχύ. Δεν έχουμε λοιπόν πρόβλημα με αυτό. Γενικά είμαστε υπέρ της πρόθεσης του ε, ελεύθερων συναλλαγών όταν αυτό είναι δυνατόν. Έχουμε κάποια ελάσσονα σημασία προβλήματα, θα έλεγα, όσον αφορά την αυριανή ψηφοφορία. Το ένα πρόβλημα αφορά τι συμβαστικέ τροπολογίε 1 και 2. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να εισάγουμε κάτι το οποίο μπορεί να παράσχει τη δυνατότητα να εισαχθεί αργότερα κάτι, κάποιο πράγμα προστατευτικής φύσης, ε, κάποια μέτρα προστατευτικά που μπορεί να επηρεάσουν ε, το εμπόριο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Συνεπώς ε, πιστεύουμε ότι τίποτα τέτοιο δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη διατύπωση αυτών των τροπολογιών. Έχουμε μία φράση που λέει ότι θα πρέπει να απέχει από νέα δασμούς ή χρεώσεις και ξέρω, ή μέτρο και ξέρω ότι ο εισηγητής θέλει να διαγραφεί η λέξη μέτρα. Εμείς θεωρούμε ότι υπό συνθήκες μπορεί και τέτοιο να προσφέρει ένα περιθώριο εισαγωγή τέτοιων μέτρων προστατευτισμού που για μας δεν είναι επιθυμητά. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα όσον αφορά τις κατεξοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Αναφερθήκατε και εσείς αυτό. Έγινε νομική ανάλυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που, είναι πλήρως, που αιτιολογεί πλήρως τη χρήση των εκτελεστικών πράξεων και το ρόλο του Κοινοβουλίου, ενώ η νομική ανάλυση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, από όσο ξέρω, θεωρούν ότι το σωστό είναι το αντίθετο. Θεωρούμε ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή για μάχες μεταξύ θεμισμικών οργάνων. Ούτε θεωρούμε ότι πρέπει εμεί να προκαλέσουμε τσακωμού. Ε, προτείνουμε λοιπόν να υποστηρίξουμε την άψη τη Κομισιόν για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν είναι η ώρα για να έρθουμε σε διένεξη. Αυτά είχα να πω εγώ από πλευρά μα. Γενικά υποστηρίζουμε την πρόταση και καλωσορίζουμε το γεγονό ότι ο σημερινό είναι άλλη μια χώρα που θα ε, παρατείνει ε, ε, τη συμφωνία της και θα υπερισχύσει αυτή, θα είναι ευρύτερη αυτή η συμφωνία που έχουμε με την Κολομβία και το Περού. Ευχαριστώ κύριο ε, Ταμόζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγγνώμη κύριε Σόλτς, αλλά οι φιλελεύθεροι πιστεύουν ότι αυτό που εμείς υιοθετηθούμε είναι αυτό το οποίο προηγούμενα ο συνάδελφος ανέφερε. Και τώρα θα μιλήσω την γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κύριος Φίσας ε, σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Για να είμαι σύντομος λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι το ελεύθερο εμπόριο είναι το μόνο δυναμικό που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αυξηθεί οικονομικά μετά από την κρίση χρέους. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο και πρέπει να ανοίξουν οι αγορές μας ε, και γι' αυτό οι φιλελεύθεροι είναι πρόθυμοι να συζητήσουν τις τροπολογίες και θα καταψηφίσουμε αύριο όλες αυτές τις τροπολογίες διότι θεωρούμε ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος εδώ να καθυστερήσουν οι τροπολογίες την έναρξη σε ισχύ αυτής της συμφωνίας γι' αυτό, γι αυτό θα καταψηφίσουμε τις τροπολογίες εδώ και σας ευχαριστούμε όλοι για το έργο που επιτελέσατε που ήταν πραγματικά αξιόλογο κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος. Σας ευχαριστώ. Uh, uh, uh. Ευχαριστούμε. Τώρα η πράσινη, η σκιώδης των πρασίνων δεν είναι εδώ. Θα πάρει τον λόγο η Επιτροπή λοιπόν. Αν επιθυμεί να παρέμβει. Κύριε Γιώργενσεν, θέλετε να παρέμβετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα να πω ότι κατανοούμε απόλυτα την επιθυμία του Κοινοβουλίου να μην του κάνουμε εκπλήξεις όσον αφορά την υλοποίηση αυτού του κανονισμού. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ακόμη και αν το Κοινοβούλιο τελικά δεχθεί να συμφωνήσει με την πρόταση της Κομισιόν, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να είμαστε όσο διαφανείς επιθυμείτε και να σας ενημερώνουμε ώστε να συμμετέχετε κι εσείς και να διατηρήσετε ενημερωμένοι από το θέμα του Ευχαριστώ. Πάντα τόσο διάφανη όπως πάντα, as usual, όσοι ήθιστε. Μάλιστα. Και τώρα έχω την τιμή να δώσω τον λόγο κατ' εξαίρεση στον Υπουργό του Ισημερινού για δύο λεπτά. Αν επιθυμείτε να προσφωνήσετε τους Ευρωβουλευτές, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να μιλήσω όμως στην γλώσσα μου σε αυτή την παρέμβασή μου. Πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα είναι τιμή και χαρά να είμαι ενώπιον σας. Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στις Βρυξέλλες στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχαμε τη χαρά να, ε, είχα την τιμή και τη χαρά να σπουδάσω κοινοτικό δίκαιο και γνωρίζω εκ του σύνεγγυς ε, το πώς λειτουργεί η Ευρώπη και η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Να σας υπενθυμίσω όμως ότι παρόμοιες διαδικασίες ενισχύονται αυτή την εβδομάδα στη Νότια Αμερική. Η ε, Νοτιοαμερικανική Ένωση Χωρών που αρχίζει στην έδρα της ε, να λειτουργεί με τα γραφεία της στο Κίτο, πρωτεύουσα του σημερινού. Θα είναι το επίκεντρο της ε, νοτιοαμερικανικής ολοκλήρωσης ε, και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα μπορέσουν να ενισχυθούν οι σχέσεις της UNASUR, της Ένωσης Νοτιοαμερικανικών Χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα στο Εκουαδόρ. Μιλήσατε προηγούμενα και είπατε όλα όσα έπρεπε να αναφερθούν. Για μας είναι ανάγκη αυτή η δυνατότητα να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός με κατεπήγοντα χαρακτήρα για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κύρια αγορά για τα εξαγώγημα προϊόντα από τον Ισημερινό εκτός του πετρελαίου πολλά από αυτά τα προϊόντα δεν μπορούν να υποκατασταθούν ή να διατεθούν σε άλλες αγορές ε, βραχυπρόθεσμα. Εξαρτώμεθα από τις ευρωπαϊκές αγορές στην Ευρώπη. Όλα όσα εξάγουμε σε σχέση με τα κυριότερα μας προϊόντα υποεξαγωγή πάνε στην Ευρώπη και ουσιαστικά υπό το γενικό σύστημα, γενικό σύστημα ε, ε, δασμολογικών προτιμήσεων. Γι' αυτό είναι αναγκαία αυτή η κατεξαίρεση ρύθμιση. Και εδώ θέλω να υπενθυμίσω εκείνοι που θα χάσουν βραχυπρόθεσμα αν δεν ε, και προχωρήσει αυτή η συμφωνία θα είναι οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Ισημερινού θα είναι οι κοινότητες και συνεταιρισμοί γεωργών και παραγωγών του Ισημερινού που εξάγουν κυρίως τα προϊόντα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως μέσω του δίκαιου εμπορίου, στο πλαίσιο του δίκαιου εμπορίου. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους κύριοι Ευρωβουλευτές ότι εμείς είμαστε αλυσοδεμένοι. Η αλυσίδα δεν, δεν τερματίζει στην πλευρά του ε, Ισημερινού ή μέσω του ωκεανού. Ε, συνεχίζεται προς την ε, Ευρώπη με πολλές επιχειρήσεις ε, που παρακολουθούν αυτά τα προϊόντα και τα ε, χρησιμοποιούν διότι έχουν πολύ μεγάλη πρόσθετη αξία και είναι συμπληρωματικά σε σχέση με τα όσα παράγει η ευρωπαϊκή παραγωγή και υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση από καταναλωτές αυτών των προϊόντων. Εμείς λοιπόν είμαστε μια χώρα που δεν πουλάει φθηνά προϊόντα αλλά προϊόντα ποιότητας και αν πρέπει βραχυπρόθεσμα να καταβάλουμε δασμολογικές ε, ε, επιβαρύνσεις ε, τότε αυτό θα είναι ιδιαίτερα αρνητικό για μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Σόξ για την εξαιρετική δουλειά που επετέλεσε και εμεί θέλουμε να ζητήσουμε να κατανοήσουν όλα τα μέλη της, Ευρωπα... της δικής σας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής την εμβέλεια αυτής της απόφασης που θα λάβετε και εμείς σεβόμενοι τα δικαιώματα που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διαβουλεύσεις με άλλα θεσμικά όργανα όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο παρακαλούμε, εκφράζουμε την παράκληση να λάβετε υπόψη το τι σημαίνουν όλα αυτά για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες του Εκουαδόρ να έχουν αυτό το μηχανισμό τάχιστα στη διάθεσή τους, κατεπηγόντως. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε λέει κύριος Λάγκα, κύριε Υπουργέ. Θα έλεγα ο κατεπήγον χαρακτήρας εδώ έχει γίνει πια κάτι το οποίο συνειδητοποίησαν όλοι. Φυσικά πολλά θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει ως προβλήματα αν αποκινούμε την Κολομβία και το Περού και την, το Οικουαδόρ είχαμε τότε υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Δεν έγινε όμως αυτό τότε. Εν πάση περιπτώσει μπορούμε να σας διασφαλίσουμε κύριε Υπουργέ ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας αυτό το, ε, σε αυτή τη διαδικασία να μην υπάρξει κενό ή τρύπα. Σόλτς, Σόλτς, σύντομα, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ Μπέρντ. Με την τελευταία παρατήρηση συμφωνώ απόλυτα. Όλοι συνειδητοποιούμε και γνωρίζουμε γιατί ο Ισημερινός δεν ακολούθησε την Κολομβία και το Περού σε αυτή τη συμφωνία. Και αυτό είναι το θέμα το οποίο κινεί τον Ισημερινό και σε σχέση με την συμφωνία αυτή αλλά και με το θέμα αυτό. Το θέμα είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε την προηγούμενη φορά και να το αναφέρω σύντομα και τώρα. Πρέπει η γενική συζήτηση να διεξαχθεί και στους δύο τομείς να λυθούν υπόψη αυτά τα θέματα και τα θέματα για τον Ισημερινό όπου διεξάγονται ευρύτερες συζητήσεις για το νόημα μιας τέτοιας ρύθμισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε εμά από δικής μας πλευράς. Γι' αυτό η πρόταση των κατεξουσιοδότηση πράξεων είναι ένα δημοκρατικό μέσο το οποίο θα εξυπηρετήσει όλες τις πλευρές προς όφελος μιας λύσης που θα είναι πραγματικά επωφελής για αμφότερες τις πλευρές. Και έτσι να το δουν και οι πολίτες και για τη διαφάνεια που ακριβώς με το παράδειγμα προηγούμενων συμφωνιών αναφέραμε. Και αυτό έχει το νόημά του και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και λαμβάνεται υπόψη στην γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Είπα ότι η νομική βάση για το Εκουαδόρ, για τον Ισημερινό, είναι διαφορετική από ό,τι για την Ουκρανία ή τη Μολδαβία ή το Πακιστάν. Δεν μπορούμε ισοπεδωτικά να τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Εμείς θέλουμε ο Ισημερινός το επαναλαμβάνω δεν είναι παιχνιδάκι άθυρμα δεν είναι μπαλάκι το οποίο παίζουμε στο ένα γήπεδο και το άλλο θέλουμε και για τους πολίτες ε, του Ισημερινού και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσουμε υπεύθυνα ευχαριστώ ωραία ευχαριστώ αύριο θα ψηφίσουμε λοιπόν στις 10 η ώρα στην αυριανή συνεδρίαση σας ευχαριστώ πολύ περνάμε στο σημείο 12 Πρόκειται για την χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Και αυτό το έχουμε συζητήσει. Έχουμε δέκα τροπολογίες που κατατέθηκαν. Δίνω τον λόγο στον εισηγητή μας, κύριο Σορίν Μόισα. Παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ πολύ σύντομος και ε, δομημένος. Μια υπενθύμηση για όλους. Ε, το θέμα εδώ αφορά τη χορήγηση στη Μολδαβία στο πλαίσιο των ήδη υπαρχουσών ε, ε, γενικευμένων ε, προτιμήσεων κάποιες μειοστασμών για κάποιες ποσότητες μήλων, δαμασκίνων και σταφυλιών επιτραπέζιων κάτω των 10.000. Έχουμε λάβει ήδη κάποιες τροπολογίες από την κυρία Λεπέν θα τις χωρίσω τις τροπολογίες σε τέσσερις κατηγορίες ε, και θέλω να τις συζητήσουμε σοβαρά κατά κατηγορία. Η μία κατηγορία αφορά την ε, τροπολογία 1 που λέει ότι αν εγκρίνουμε αυτήν την τροπολογία με κάποιο τρόπο θα είναι να, σαν να εγκρίνουμε το κίνητρο της ε, Μολδαβίας για να γίνει μέλος της Ένωσης ε, σε κάποια χρονική στιγμή. Ωστόσο αυτό αφορά, ξέρετε, κάποιες μικρές ποσότητες από Δαμάσκηνα και Μήλα. Δεν αφορά κάποια πολιτική σύνδεση της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα δεν αφορά την προσχώρηση της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική σύνδεση της Μολδαβίας, όπως και για τις υπόλοιπες ε, άλλες χώρες και της Ευρώπης, δεν είναι απαραίτητα κάτι που οδηγεί στην προσχώρηση. οι γενικευμένες προτιμήσεις οι πολιτικοί ενδιαφερόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Μολδαβία όταν προσεγγίζονται ε, ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω σε κάθε τέτοια περίπτωση θα υπάρχουν 28 βέτο από κράτη-μέλη για να ορίσουμε μια χώρα ως πιθανό υποψήφιο, για να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις, να ξεκινήσουμε και να κλείσουμε κάθε κεφάλαιο και να επικυρώσουμε τη συνθήκη στο τέλος. Η Μολδαβία δεν ε, βρίσκεται καν πολύ κοντά, δυστυχώς, ανάλογα με τις απόψεις του καθένα, βέβαια. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι κρυφό, δεν ε, υπάρχει κάποια ενέδρα που επίκειται, δεν υπάρχει κάτι που ορίζει το μέλλον της Μολδαβίας. Ε, με κάποιο θέμα ε, ε, προσχώρησης αφορά τα μήλα, τα δαμάσκηνα, τα σταφύλια και κάποιους στοχούς αγρότες που θα υποφεληθούν χωρίς να προκαλέσουν κάποια ζημιά καθόλου μάλιστα στην ευρωπαϊκή αγορά. Η δεύτερη κατηγορία τροπολογιών είναι 4, 5, 6 και 8 που ουσιαστικά απορρίπτουν τις εκχωρήσεις με διάφορους τρόπους ε, δεν συμφωνούμε. Αν τις εγκρίνουμε είναι σαν να λέμε δεν συμφωνούμε με την πρόταση της Κομισιόν οπότε δεν θέλουμε να χωρίσουμε αυτές τις προτιμησιακές ρυθμίσεις στη Μολδαβία. Οι 2, 3, 9 και 10 τώρα τροπολογίες κάνουν έκκληση για έρευνες από την Κομισιόν για το κατά πόσο η Μολδαβία τηρεί τους κανόνες ε, πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά η Μολδαβία εδώ θεωρείται ότι είναι ένοχη οπότε υποτεθεί ή πρέπει αμέσως ή μόλις τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός να ξεκινήσουμε τις έρευνες. Να διαβεβαιώσω όλους ότι ο αρχικός κανονισμός που εμείς τροποποιούμε έχει διατάξεις για αναστολή του προτιμησιακού καθεστώτος σε περίπτωση που η Μολδαβία δεν τηρεί τους κανόνες καταγωγής και σε αυτή την περίπτωση η Κομισιόν ε, εφόσον έχει πρέπει να έχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σε μια κοινωνία δικαίου λοιπόν δεν επιτεθέμεθα σε, απλά σε χώρες και ανθρώπους ε, πρέπει να υπάρχουν κάποια διάστα στοιχεία ότι κάτι πάει λάθος και υπάρχει και ένα ξεχωριστό άρθρο για τα μέτρα ε, διασφάλισης σε περίπτωση που οι εισαγωγές από μια συγκεκριμένη χώρα από τη Μολδαβία στη συγκεκριμένη περίπτωση αποδειχθεί ότι ζημιώνουν την αγορά μας, την εσωτερική αγορά, τότε έχουμε τα κατάλληλα μέσα για να παρεύουμε. Αυτά είναι μικρά TRQ, μικρές δυσμαλογικές ποσοστώσεις που πολύ εύκολα μπορούν να απορροφηθούν και μόνο από τη ρουμανική αγορά. Οπότε είναι απίθανο να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο, αλλά να διασφαλίσω, να διαβεβαιώσω του συναδέλφου και την κυρία Λεπέ, τα μέτρα υπάρχουν ήδη σε περίπτωση που χρειαστούν. Και μετά υπάρχει η τροπολογία 7, η οποία αναφέρεται σε μια τεχνική προσαρμογή στο νέο τελωνιακό κώδικα της Ένωσης, που τεχνικά είναι σωστή η τροπολογία όπως προτείνει η κυρία Λεπέν, αλλά είναι περιττή διότι καλύπτεται ήδη από το κείμενο της Κομισιόν. Η πρόθεση πίσω από αυτό είναι ότι αν δεχθούμε οποιαδήποτε τροπολογία πρέπει να ακολουθήσει τριμερής διάλογος με την Κομισιόν και το Συμβούλιο και θα χάσουμε παραπάνω χρόνο. Η αντίφαση που διακρίνει αυτές τις τροπολογίες είναι ότι αν τις δεχθούμε όλες απορρίπτουμε ουσιαστικά όλες τις εκχωρήσεις και ξεκινάμε σε βάθος ε, έρευνες κατά των φτωχών Μολδαβών και αυτό θα ήταν λίγο σουρεαλιστικό. Θερμά λοιπόν παροτρύνω τους συναδέλφους να συμφωνήσουν ότι ε, είναι απλά μια πολύ λογική λύση να απορρίψουμε όλες τις τροπολογίες. Δηλαδή να δεχθούμε τον κανονισμό όπως τον προτείνει η Κομισιόν. Και καλό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στην ε, Επιτροπή Πολιτικής Τζάι την περασμένη, Δευτέρα, την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν χωρίς τροπολογίες και η Κομάγκρη που συνήθως είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική στην απελευθέρωση του εμπορίου και της γεωργίας ε, ενέκρινε την πρόταση της Κομισιόν χωρίς καμία τροπολογία με συντριπτική πλειοψηφία 35 ψήφοι υπέρ, 5 κατά και 2 αποχές σήμερα το πρωί μόλις. Οπότε πιστεύω ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ε, ε, για να μπορέσουμε να δεχθούμε την πρόταση και να κρίνουμε την πρόταση της Επιτροπής όσο έχει χωρίς τροπολογίες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στον σκιώδη του κ. Βέγκλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μια σκέψη πρώτα και μετά πιο συγκεκριμένα στις τροπολογίες. Ναι, φυσικά εκτιμάμε ιδιαίτερα το, η δουλειά του κυρίου Σιγητή και τις εξηγήσεις που μόλις ακούσαμε για τις 10 τροπολογίες. Πριν από αυτό όμως θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή αυτή εδώ παλαιότερα επίσης αποφάσισε υπέρ μέτρων τα οποία βοήθησαν τη δημοκρατία της Μολδαβίας και το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μολδαβίας. Το ερώτημα έχει τεθεί από πολλούς ε, συναδέλφους και τον Χελμουτσούλης που είναι εδώ. Παλιότερα τα μέτρα αυτά έχουν αυτά αποτελέσματα, ορατά. Είναι σημαντική ερώτηση. Χθε συναντήθηκα με τον πρέσβη της Μολδαβίας εδώ στις Βρυξέλλες και μου έλεγε για τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια, τις διεργασίες ε, στο τομέα της ε, ε, Γιατί θα θυμάστε ότι είχαμε δώσει και διαστήματα για εισαγωγή ίνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μου είπε ο ότι η εινοποιία αναζητά νέε τεχνολογίες και τρόπους προσαρμογής στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό είναι μια σκέψη για να απαντήσω σε κάποιε ανησυχίε. Τώρα όσον αφορά τι τροπολογίες θεωρώ ότι ο κ. Σιγητή μας έδωσε επαρκείς εξηγήσει. και το ΕΛΚΑ ε, θα καταψηφίσει και τις 10 τροπολογίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σαβαλιά. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. ε, καταλαβαίνουμε αυτό το πολύ ε, εξαιρετικό μέτρο και αυτή την έκφραση αλληλεγγύης φιλίας με τη Μολδαβία. Πιστεύουμε ότι έχει πολύ περιορισμένο πεδίο, καλύπτει μόνο τρία προϊόντα. Τα περισσότερα από αυτά το πιθανότερο είναι να απορροφηθούν από την αγορά μίας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν βέβαια αυτή η χώρα στην προηγούμενη περίπτωση Ρουμανία δεν διαμαρτυρηθεί. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε κανένα λόγο να διαφωνήσουμε. Έτσι λοιπόν σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με τον εισηγητή και με την Κομισιόν και θα ψηφίσουμε κατά οποιασδήποτε πρότασης που προσπαθεί να αντιτεθεί ή να περιορίσει με κάποιο τρόπο αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση Αυτά έχω να πω προς το παρόν. Ευχαριστώ. Οι φιλελεύθεροι δεν παρίστανται. Ο Χέλμουτ λοιπόν έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι σύντομος. Ήδη την τελευταία φορά σε σχέση με τον εισηγητή στην τοποθέτηση του για την τροποποίηση του κανονισμού σε σχέση με την μετατροπή δηλαδή συμμεριστήκαμε την άποψή του και συμφωνήσαμε μαζί του ταυτόχρονα θέλω όμως να καταστήσω σαφές ότι για το μέλλον θα πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν ας το πω έτσι από πλευράς των αγαθών αυτών της δημοκρατίας της Μολδαβίας να υπάρξει μια δυνατότητα που θα διασφαλίζεται για να προχωρήσει μια τέτοια συμφωνία. Δηλαδή όχι μόνο για γεωργικά προϊόντα από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξουμε τις πύλες μας, αλλά να συνεισφέρουμε γενικότερα η Δημοκρατία της ε, Μολδαβίας ε, να μπορεί να δρά και να εξαγάγει με υψηλότερης αξία προϊόντα. Ευχαριστώ. Μάλιστα σας ευχαριστώ και οι πράσινοι δεν παρίστανται. Τώρα η κυρία Λεπέν. Παρακαλώ κυρία Λεπέν. Κύριε Ισηγητά, σχετικά με τα επιχειρήματά σας. Κάποια στιγμή υπάρχει το δικαίωμα, υποστηρίζουν το δικαίωμα τροπολογίας ε, με επιχειρηματολογία που αφορά τη δημοκρατία. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ε, αυτό που λέμε, ε, το, την ανάγκη να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του λαού της Μολδαβίας αλλά ελάχιστο ακούω για την υπεράσπιση των λαών της Ευρώπης. Γιατί εμείς εδώ γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε, για την ε, ε, υπεράσπιση των ε, συμφερόντων των λαών της Ευρώπης. Και εγώ συμπαθώ την Μολδαβία, αλλά εδώ συζητάμε για κατεξαίρεση κάποια στιγμή μέτρα, αλλά κατεπήγοντα μέτρα, εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, αλλά τελικά καταλήγουμε λίγο-λίγο να κάνουμε ένα σοβαρό αποτέλεσμα. Λοιπόν, βεβαίως δημιουργούμε, δεν υπάρχει αμφιβολία, κίνδυνος να υπάρξουν προβλήματα για τους δικούς μας αγρότες. Ας πούμε, εδώ αυτό που βλέπω εδώ και γι' αυτό έχω υποβάλει τροπολογίες είναι ότι διαφυσβήτητα δυστυχώς η κατάσταση Μολδαβία μοιάζει με την κατάσταση στην Ουκρανία στη διάρκεια της κρίσης. Δηλαδή αν υπάρχει ένα μέρος που στρέφεται προς τα δεξιά ε, στην, ε, σε εκλογέ ε, της Κυριακής υπάρχει ένα κόμμα που κοιτάζει προς, τα, προς Ανατολάς πολιτικά η υπόθεση της ένταξης της, των σχέσεων της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκαλεί διαφωνίες στο ιστορικό της χώρας. Έτσι λοιπόν εμείς είμαστε υποχρεωμένοι με βάση την εμπειρία μας να διαπιστώσουμε ότι οι ελεύθερες ε, ε, συναλλαγές και οι εμπορικές συμφωνίες είναι πάγοντα ένα είδος πολιτικής ε, σύγκλησης. Δεν είναι ο ρόλος και φυσικά δεν, είναι, δεν μιλάμε κατά ανάγκη για περαιτέρω διεύρυνση. Εδώ και καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συγχαίουν ε, σκόπιμα αυτά τα δύο πράγματα. Και το άλλο είναι η μεγάλη δυσκολία που έχουν οι αγρότες μας όταν βλέπουν τις τιμές να καταραίουν και αυτό είναι που με απασχολεί περισσότερο και υπάρχουν ε, ε, αντίπεινα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία. Οι δικοί μας αγρότες ε, υποφέρουν, αυτούς πρέπει να υποστηρίξουμε κυρίως Πεναντί τους έχουμε ευθύνη και δεν νομίζω ότι σε περίοδο κρίσης της γεωργίας όπου, στην οποία είμαστε, βρισκόμαστε εντός, να δίνουμε ευνοϊκή μεταχείριση σε άλλα προϊόντα, όποια και αν είναι αυτά και από που και, οπουδήποτε και αν προέρχονται. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνει μια έρευνα της Κομισιόν αν, για να διαπιστωθεί αν μια τέτοια συμφωνία δεν θα συνεπάγεται περαιτέρω δυσκολίε για τους ε, αγρότες μας, αλλά αυτό μου φαίνεται ήδη περί τι δαπάνη. Ευχαριστούμε πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω το εξαιρετικό έργο του εισηγητή και του Σκιώδους που θεωρώ ότι συνόψαν εξαιρετικά το στόχο και τη φύση των ε, τροπολογιών. Ε, ναι, υπενθυμίζω ότι πράγματι υπάρχουν μέτρα έρευνα σε περίπτωση που χρειαστεί, σε περίπτωση απάτη, σε περίπτωση προβλήματων εισαγωγών. Προβλέπονται ήδη στο βασικό κανονισμό. Οπότε οι τροπολογίες αυτές δεν προσθέτουν τίποτα. Όσον αφορά τα δύο επιχείρηματα τη κυρία Λεπέν, Πρώτα απ' όλα την ε, διαφωνία αυτή περί της Μολδαβίας να υπενθυμίσω ότι τίποτα στην Συμφωνία Σύνδεσης και τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών που έχει υπογράψει τη Μολδαβία δεν εμποδίζει τη Μολδαβία να έχει οικονομικές και εμπορικές προνομιακές σχέσεις με όλους τους εταίρους με τους οποίους έχει αυτή τη στιγμή προνομιακές συμφωνίες συμπεριλαμβανομένες φυσικά και της Ρωσίας και του εταιρού τη κοινότητα ανεξαρτητών κρατών. Αντιθέτω έχουμε ενθαρρύνει τη Μολδαβία, ναι Το πρόβλημα είναι όμω ότι η Ρωσία τα πράγματα τα βλέπει διαφορετικά, γιατί η Ρωσία πράγματι άρχισε, ε, εφάρμοσε μέτρα εμπάργκο μέσω ψευδών ε, μέτρων ε, φυτογενομικών μόλις υπέγραψε τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση η Μολδαβία. Δεύτερον, όσον αφορά τις δυσκολίες ε, για τους Ευρωπαίους Γεωργούς, να επενθυμίσω ότι οι ποσότητες για τις οποίες μιλάμε εδώ είναι αμελητές σε σχέση με το μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς. Αντιστοιχούν στο 0,8% για τα μήλα, δηλαδή το σύνολο των ε, μήλων της Μολδαβίας, ε, εάν το 100% αν το εξήγαγαν στην Ευρώπη θα αντιστοιχούσε σε 0,8%. 1,4% για τα δαμάσκηνα και 1% για τα σταφύλια. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι η Ρωσία η οποία ε, λαμβάνει μέτρα κατά των εξαγωγών στην Ευρώπη. Πρόκειται για κυρώσεις ε, που ε, έχουν, βασίζονται σε κινήσεις προστατευτισμού. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Συγητής. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα για το οποίο συμφωνώ με την κυρία Λέπεν. Είμαστε εδώ για να υπερασπίσουμε τους Ευρωπαίους, τους πολίτες μας και τους Ευρωπαίους Γεωργούς. Εγώ ήμουν επικεφαλής του γραφείου του Επιτρόπου Γεωργίας στην τελευταία επιτροπή και υπεράσπισα στεναρά τους Γεωργούς και τους Γεγάλους Γεωργούς. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση πραγματικά δεν υπάρχει καμία διαφωνία, διότι η Ρουμανία για παράδειγμα φέτος παράγει 3 μίλα λιγότερα, 22% μείωση της παραγωγής και από αυτά τα τρία λιγότερα μόνο ένα μπορεί να δικαταστήσει η Μολδαβία. Συνεπώς πραγματικά δεν υπάρχει κίνδυνος, οποιοδήποτε κίνδυνος για την ευρωπαϊκή αγορά γενικότερα, ούτε καν για τη ρουμανική αγορά, πόσο μάλλον για τη γαλλική, την ιταλική κτλ. Αλλά ακόμα και αν ε, πρόκειται να υπάρξει κάποια επιρροή στην τιμή στην Ευρώπη, εμείς έχουμε συμφέροντα πολύ ευρύτερα από τη σταθερότητα της Μολδαβίας. Είναι συμβολική η κίνηση γιατί πραγματικά είναι αμελητές ποσότητες. Ακόμη και αν επηρεαζόταν η τιμή που δεν πρόκειται, θα άξιζε τον κόπο για να βοηθήσουμε στη σταθεροποίηση μιας αγροτικής κοινωνίας με μια πολύ μικρή κίνηση που δεν μας κοστίζει τίποτα στηρίζει και τα δικά μας συμφέροντα. Υπάρχουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στη Μολδαβία. Έχουμε θέματα συμφέροντα που αφορούν την ασφάλεια στα σύνορα της Μολδαβίας. Ε, δεν επιθυμούμε την υπερβολική μετανάστευση από τη Μολδαβία. Λοιπόν, είναι ελάχιστη η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε και η θυσία. Συμφέρει εμάς ως Ευρωπαίους. Κάνουμε μια κίνηση που για αυτούς είναι σημαντική, αλλά που εμάς δεν μας κοστίζει σχεδόν τίποτα. Συμφωνώ μαζί σα. Ναι, πρέπει να εργαζόμαστε για τον εαυτό μα, να εκπροσωπούμε του Ευρωπαίου, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά έχετε άδικο. Δεν ρηψοκινδυνεύουμε ε, τίποτα την κατάσταση τη ευρωπαϊκή αγορά καθόλου, ούτε την κατάσταση των Γάλλων Γεωργών. Ευχαριστούμε πολύ. Σα ευχαριστούμε. Αύριο, αύριο θα ψηφίσουμε. Θα ήθελα όμω αυτό που είπε ο εισηγητή στην πρώτη του παρέμβαση να το τονίσω να το υπογραμμίσω. Μια επιστολή πήρα από το Συμβούλιο, στην οποία στο Συμβούλιο την έγκριση χωρίς τροπολογίες σε αυτό το αίτημα προαναγγέλει. Και κατά τούτο λοιπόν ταχύτατα θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και να το διευθετήσουμε. Λοιπόν, όπως είπα, ψηφίζουμε αύριο. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Το οποίο είναι το υπαριθμό 13. Πρόκειται εδώ για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και τη στρατηγική για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Να σας αναφέρω επ' αυτού ότι αποφασίστηκε από τους συντονιστές να μην συνταχτεί γνωμοδότηση για την ε, έκθεση που είναι αρμόδια για αυτήν η Επιτροπή Εξωτερικών, ΑΦΕΤ, Εξωτερικών Υποθέσεων. Και αυτό επειδή διότι δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε με την ΑΦΕΤ, την Επιτροπή Εξωτερικών, να υπάρχει μια σαφής διαχωριστική γραμμή όσον αφορά τις αρμοδιότητες εκάστοτε γενικού πολιτικού χαρακτήρα για την ΑΦΕΤ και ειδικού εμπορικού χαρακτήρα για την ΙΝΤΑ, τη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Και έτσι τέλος αποφασίσαμε ότι η ΑΦΕΤ θα συντάξει μια γενική έκθεση γενικού πολιτικού χαρακτήρα χωρίς, χωρίς να υπάρχουν πτυχές που αφορούν το εμπόριο σε αυτήν χωρίς να θίγονται τέτοιου είδους πτυχές. Και εμείς από πλευράς μας ως Επιτροπή Εμπορίου θα συντάξουμε μια ξεχωριστή έκθεση ή ψήφισμα, θα δούμε τι θα κάνουμε ακριβώς, ως Επιτροπή Εμπορίου. Μόνοι μας εμείς ώστε τις δικές μας αρμοδιότητες να τις διασφαλίσουμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την ξεχωριστή έκθεση ή ψήφισμα. Κατά τούτο θα επικεντρωθούμε λοιπόν στα ε, θέματα που αφορούν το εμπόριο στην αναθεώρηση της ε, πολιτικής, ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Αλλά αυτό και σε περίπτωση μιας γνωμοδότησης θα συνέβαινε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Όμως είναι μια συνετή λύση πιστεύω αυτή. Διότι αν μόνο μια γνωμοδότηση συντάσαμε τότε η Επιτροπή Εξωτερικών <clears throat> σε σχέση με τη δική μας νομοδότηση θα μπορούσε να ψηφίσει για θέματα δικής μας αρμοδιότητας. Δεν θα είχαμε ηχέγγυα στο τέλος τέλος οι δικές μας απόψεις να εντασσόντουσαν με κατοχύρωσή τους στην, κοινή, στην έκθεση αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Επιτροπής αφετά. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν εμείς. Θα συντάξουμε ή ξεχωριστή έκθεση ή ψήφισμα. Θα γίνει η συζήτηση λοιπόν να κάνουμε κάτι ξεχωριστό εμείς ως Επιτροπή Εμπορίου στο μέλλον. Και δίνω λοιπόν τον λόγο στους δύο συνεισήγητες. Πρώτα στην κυρία Μαρία Αρένα. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ούτω ή άλλω αυτό που προτείνεται μου φαίνεται ενδιαφέροντα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει να ε, εστιάσουμε την προσοχή μα στη συνοχή των πολιτικών γιατί όταν μιλάμε για πολιτική γειτονία και το υπενθύμισε η κυρία Επίτροπος προηγουμένω, η διάσταση του εμπορίου ε, όπω εννοείται εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πολιτικό σύνολο πλαίσιο ε, που, στο οποίο βασίζεται η πολιτική και η δημοκρατική εξέλιξη στις χώρες. Τώρα για την πολιτική γειτονία και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την πτυχή του Νότου Εκεί θα επικεντρωθώ. Στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας υπάρχει μια σημαντική αρχή που λέει ότι όσο πιο πολλές προόδους κάνει μια χώρα όσον αφορά το σεβασμό των δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλύτερη πρόσβαση έχει, τόσο καλύτερη πρόσβαση θα έχει στην ευρωπαϊκή αγορά. Πρέπει να μείνουμε πιστοί σε αυτή την αρχή που υπερασπίζει την, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες. Μετά από τις διάφορες επαναστάσεις που είχαμε γύρω από τη Μεσόγειο, σήμερα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς ε, ποια υπήρξαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ε, εμπορικής πολιτικής σε αυτό, στις χώρες και σε αυτό το πλαίσιο. Αναφέρομαι φυσικά σε κάποιες χώρες με τις οποίες έχουμε ήδη συμφωνίες αλλά και σε άλλες όπου μόλις τώρα ξεκινούν ε, οι, συμφωνίες, οι συμφωνίες είναι νέες ναι, οι συμφωνίες. Να υπενθυμίσω την κατάσταση του Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Έχουμε συμφωνίες εδώ και χρόνια. Ορισμένες συμφωνίες έχουν επικαιροποιηθεί, αναβαθμιστεί στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που έχουν γίνει. Ενδιαφέρον θα ήταν να ζητήσουμε κάποια αξιολόγηση των συμφωνιών αυτών βάσει των όσων ανέφερα προηγουμένω. Πώ δηλαδή αυτές ε, οι συμφωνίε ενίσχυσαν τι δημοκρατικέ αξίε και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σύνολο αυτών των χωρών. Είναι σημαντικό να γίνει αυτό σήμερα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ Μαρία. Και τώρα ο κύριο Λαντσπέργκη για το ανατολικό κομμάτι γειτονία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποιος πριν από λίγες μέρες μου είπε ότι ζούμε στην εποχή των τίτλων στις εφημερίδες. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συντάξει κανείς μια έκθεση σε, όταν ζει εποχή, σε τέτοια εποχή, όταν βρίσκεσαι σε χώρες όπως η Ουκρανία ή η Γεωργία που τα γεγονότα ε, ακολουθούν το ένα το άλλο με μεγάλη ταχύτητα. Θεωρώ ότι ήταν ε, πετυχημένη η πορεία ε, με τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας όσον αφορά το more for more, δηλαδή που μπορούμε να προσφέρουμε και περισσότερη υποστήριξη. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος για μας. Ιδίως τώρα που συζητάμε για την Ουκρανία, μια ατζέντα για μεταρρυθμίσεις που πρέπει να ανακοινωθεί σύντομα, ενδεχομένως και αυτό το μήνα, αυτό εμπίπτει στα θέματά μας. Όμως υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα το οποίο το ανέφερα στην κυρία Μάλμστρομ ότι δηλαδή αν τώρα ιδίως ε, συζητηθεί το θέμα της ενισχυμένης συνεργασίας ή της ανανέωσης συνεργασίας με τη Ρωσία σε μια στιγμή που υπάρχει η κρίση στην Ουκρανία, κατά την άποψή μου θα μπορέσει να ε, θα οδηγήσει στο να ε, καταστραφεί η ανατολική εταιρική σχέση. Δηλαδή η Ρωσία έχει εισβάλει σε μέρη της Ουκρανίας, δεν τηρεί τη συμφωνία της με τον ΠΟΕ όπως είπε και η κυρία Μάλμστρομ. Αν τώρα ε, εμβαθύνουμε στη συνεργασία μας με τη Ρωσία, ποιο είναι το μήνυμα που θα στείλουμε στους εταίρους των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Πρέπει λοιπόν πρώτα να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με τη Ρωσία, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιο δρόμο θα ακολουθήσει η ανατολική εταιρική σχέση. Όπως είπα προηγουμένως, ο σωστός δρόμος είναι αυτός που ακολουθούσαμε πριν, αλλά εξαρτάται από το τι θα κάνουμε με τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Κύριο Ζαφράντη, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο από εμά θα θέλαμε να παρέμβουμε εξ ονόματος ECR. Ίσως μπορούμε να το κάνουμε ένας τώρα να παρέμβει και ο άλλος ε, στη συζήτηση μετά. Διαρωτώ με θα επιτρέπατε και σε άλλους να συμμετάσχουν έτσι. Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Δίνω λοιπόν τον λόγο στον συνάδελφο από το Βέλγιο και εγγράψτε με σας παρακαλώ στον κατάλογο αγορητών για υστερότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν να σας... Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Πράγμα. Επιμερίσαμε αυτές τις αρμοδιότητες και εγώ θα επικεντρωθώ στην ε, νοτιότερη ε, πτυχή της πολιτικής γειτονίας που είναι πολύ σημαντική αυτή η πολιτική για την ομάδα ECR και για το κόμμα μου για την ε, πολιτική αυτή που πρέπει να επανεξεταστεί για δυνατότητες βελτίωσης που μπορούν να απορρεύσουν εμείς ε, θεωρούμε ότι έχει αποφασιστική σημασία αυτό το στοιχείο και τα εξή άλλα υπόλοιπα στοιχεία. Οικονομική ολοκλήρωση. Πρέπει να θέσουμε το ερώτημα κατά πόσον μπόρεσε να προωθήσει την ε, οικονομική ολοκλήρωση η μέχρι σήμερα ακολουθηθήσα πολιτική. Δεύτερον, αυτό που ανέφερε η κυρία Ρένα, τα θέματα δημοκρατίας. Πάντα στόχος μας ήταν να ενδυναμωθεί η δημοκρατία σε αυτή την περιοχή του κόσμου, ιδιαίτερα μετά από τις ταραχές στον αραβικό κόσμο. Θα συνιστούσαμε να εξετάσουμε κατά πόσον το εμπόριο μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο για την ανάπτυξη, την ενδυνάμωση της δημοκρατικής συνιστώσας. Τρίτο, βελτίωση, αλλά εξίσου σημαντικό και αυτό το θέμα, βελτίωση των υποδομών η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησαν σχέδια και προγράμματα στις ε, εμπλεκόμενες χώρες με την βοήθεια των οποίων οι εσωτερικές υποδομές μπόρεσαν ε, να αρχίσουν να δημιουργούνται. Πρέπει να ρωτήσουμε, συνεισέφεραν για την οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών αυτές οι υποδομές. Είναι αποφασιστική σημασία σε αυτό. Τέταρτο, ΜΜΕ, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο των ΜΜΕ. Πρέπει να δούμε πώς μπορούν να διεθνοποιηθούν εντός εισαγωγικών η ΜΜΕ για να διαδραματίσουν ένα ευρύτερο ρόλο. Και ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχω υπόψη μου κατά πόσον έχει υπόψη η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης να κάνει κάτι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτή τη συνιστόσα. Τελευταίο ζήτημα, Γεωργία πολλές από αυτές τις ε, χώρες γειτονίας εξάγουν γεωργικά τους προϊόντα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πρόκειται για μικρές μονάδες, γεωργικές μονάδες και όχι για μεγάλους παραγωγούς. Αυτή η μικρής κλίμακας ε, γεωργοί μπορούν σε σχέση με τις φυτοϊγειονομικές προϋποθέσεις και κτηνιατρικές προϋποθέσεις έχουν δυσκολίες να τις υλοποιήσουν. Πώς μπορούμε εμείς συμβουλευτικά να δράσουμε ώστε να μπορούν να βοηθηθούν να υλοποιήσουν αυτούς τους κανονισμούς και να τους σεβαστούν η μικρή αυτή παραγωγή. Αυτά τα πέντε αιτήματα θέλουμε να παρουσιάσουμε και μας ικανοποιεί το ότι μια ξεχωριστή έκθεση θα συντάξουμε και όχι γνωμοδότηση για λογαριασμό άλλων. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Δεν έχουν ζητήσει άλλοι τον λόγο. Ο Χέλμουτ λοιπόν θα λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ Μπέλτ. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τους σκιώδεις που απουσιάζουν. Όμως κάποια σημεία, τρία σημεία πολύ σύντομα, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις από αυτόν. Ναι και απόψε στην ακρόαση με την κυρία Μάνστρομ διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο. Πιστεύω ότι στην πολιτική γειτονία και προς, προς Ανατολάς και προς Νότον πρέπει πολύ σοβαρά να δούμε ποιες αλλαγές ε, μπόρεσε, μπόρεσε να προαγάγει για μια στενότερη συνεργασία μεταξύ ε και των εμπλεκόμενων χωρών και τι συνεισέφερε για την εσωτερική σταθεροποίηση και την δημοκρατία, εκδημοκρατισμό αυτών των χωρών. Και βρίσκω εγώ τουλάχιστον, χωρίς να επισέλθω στα επιμέρους σημεία, το αποτέλεσμα ότι δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό, για να μην πω ότι είναι και απογοητευτικό κιόλας. Όταν λέει ο τύπος, τα μέσα ενημέρωσης λένε ότι με τη δίκη του Μουμπάρακ στην Αίγυπτο, ας το πούμε, και η τελευταία προσπάθεια εκδημοκρατισμού στην Αίγυπτο με την ε, Αραβική Άνοιξη απέτυχε και υπονομεύτηκε, ε, πρέπει να διατυπώσουμε το ερώτημα. Πώς θα διαμορφωθεί μελλοντικά η οικονομική συνεργασία με τις χώρες του Νότου και τις χώρες προς Ανατολάς. Αν δούμε τη Μέση Ανατολή που δεν εδώ, ε, δεν εμπλέκεται άμεσα εδώ, αλλά και αυτό μας αφορά. Αν δούμε και τι συμβαίνει στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, για να μην πούμε τίποτα για τη Λιβύη. Κατά τούτο λοιπόν τα ερωτήματα αυτά, τι μπορεί να συνεισφέρει το εμπόριο και τι δεν μπορεί να συνεισφέρει, δηλαδή που το εμπόριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό μέσο άσκησης πολιτικής, αλλά πρέπει να υπάρξουν γέφυρες, γεφυροποίηση για μια πολιτική εταιρική σχέση, ας το αποκαλέσω έτσι. Και στη Μέση Ανατολή δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά τα πράγματα. Στη Δε Ανατολή απόλυτα δυσάρεστη η κατάσταση. Ουκρανία, Λευκορωσία, Κάυκασος και όλα αυτά θέτουν το ερώτημα. Η δική μας η έκθεση δεν μπορεί να συνεισφέρει αυτή που θα συντάξουμε ουσιοδός ώστε να προπαρασκευαστεί η Σύνοδος Κορυφής για αυτά τα θέματα. Θα έχουμε συγκεκριμένο χρονοορίζοντα, συγκεκριμένες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το δεχόμαστε δηλαδή εμείς οι Αμερικανοί να ε, ε, παρακολουθούν τα θέματα πυρηνικής ενέργειας στην Ουκρανία και των αντιδραστήρων και οι Ευρωπαίοι να αρτεθούν στο περιθώριο. Μόνο κάποια θέματα θέλω εδώ να σκιαγραφίσω. Αδειμονώ για τη συνεργασία, για το έργο, για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. παρακαλώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο. Και για την Ανατολική και για την Νότια γειτονία. Θεωρώ ότι η κατευθυντήρια αρχή για μας ακόμα και στην εμπορική πολιτική πρέπει να είναι ότι δεν ε, ταιριάζει το ένα η μία εκδοχή σε όλους κάθε φορά. Αν δούμε κάθε χώρα χωριστά μπορούμε να εντοπίσουμε τις διαφορετικές τους θέσεις και τα διαφορετικά τους ε, συμφέροντα. Οι χώρες της ανατολικής γειτονίας. Ακόμα και αυτές που είναι στον Κάφκασο, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, έχουν διαφορές μεταξύ τους. Οπότε μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τη μία από την άλλη. Πρέπει να τις ε, αξιολογήσουμε χωριστά και όχι να τις ρίξουμε όλες στο ίδιο καλάθι. Αυτό καμιά φορά δεν δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ήδη ακούσαμε την υπεριαλιστική όρεξη της Ρωσίας. Είναι σαφές ότι υφίσταται απέναντι σε συγκεκριμένες χώρες ανατολικά. Και πρέπει να αποφύγουμε τα σφάλματα. Είναι απαραίτητο να προσαρμοστούμε στο ότι έχουμε κάνει κάποια και δεν θα πρέπει να στριμώχνουμε τις χώρες στη γωνία όπου θα πρέπει να αναγκαστούν να επιλέξουν ή το ένα ή το άλλο. Να μπορούν να βρουν έναν τρόπο ώστε να διατηρούν εξίσου καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα να μην αποξενώνονται από άλλους ε, πιθανούς δεσμούς ή ευκαιρίες ή προσεγγίσεις. Όσον αφορά την νότια γειτονία, η όλη διαδικασία ξεκίνησε όταν στις περισσότερες από τις χώρες αυτές κυβερνούσαν ε, λαϊκοί ε, δικτάτορες ή αυταρχικοί ηγέτες που ζούσαν σε μεδανικό χρόνο. Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς όμως τα κόμματα αυτών των ανθρώπων έχουν, τα έχουν διαδεχτεί ομάδες ε, ριζοσπαστικές. Βεβαίως υπάρχουν και παραδείγματα όπως στην Ισίας που έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, ένα πολυκομματικό σύστημα, ε, σχεδόν ελεύθερες εκλογές που τηρούν διάφορα πρότυπα η Λιβύη, όπου υπάρχει πλήρης αποτυχία του ίδιου του κράτους θα έλεγα στην Αίγυπτο. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση η Αίγυπτος. Ε, τώρα ε, υπάρχει σταθερότητα για την οποία πληρώθηκε βαρύ τίμημα και σαφώς το τίμημα είναι ο περιορισμός κάποιων ε, ατομικών ή πολιτικών δικαιωμάτων και αυτές οι χώρες πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά περίπτωση, ενώ βεβαίως η Συρία βρίσκεται σε πλήρη διάλυση και σε πόλεμο. Πρέπει να βρούμε τις θετικές περιπτώσεις, να συνεργαστούμε μαζί τους, να βρούμε κάτι απτό και συγκεκριμένο και να μην ε, με κανένα τρόπο στηρίξουμε στοιχεία που είναι εχθρικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είχα να πω νομίζω. Ποτέ δεν ήμουν υποστηρικτής του να χρησιμοποιείται το εμπόριο ως εργαλείο πολιτικής, όμως σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να δικαιολογείται. Και κυρίως θα πρέπει κάθε χώρα να την αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά με βάση τις προτιμήσεις της, τη συμπεριφορά της, τη στάση της και την κατάσταση ε, στην οποία βρίσκεται τα πρότυπα ε, που έχει πετύχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει κάποιος από πλευράς Επιτροπής. Α, θαυμάσια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Um, thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ας ξεκινήσουμε από την Ανατολή. Πράγματι πολλά έχουν γίνει μεταξύ των συνόδων κορυφής του Βίλνιους και της Ρήγα. Κάποια θετικά, κάποια λιγότερο. Σαφώς λοιπόν ε, καλωσορίζουμε αυτή τη μελλοντική έκθεση και θα συνεργαστούμε στο μέγιστο βαθμό. Σίγουρα διαφορετική διαδρομή έχουν ακολουθήσει οι ανατολικοί εταίροι, η Γεωργία και η Μολδαβία έχουν συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών και τις εφαρμόζουν. Η Ουκρανία την προετοιμάζει για το χρόνο, η Λευκορωσία και οι Αρμενία έχουν ακολουθεί την ε, ευρασιατική οδό. Δεν τις τιμωρούμε φυσικά, συνεχίζουμε να τις βοηθάμε. Δεν άρουμε καν τις ε, προτιμησιακές ε, ρυθμίσεις όσον αφορά την Αρμενία. Και το Αζερμπαϊτζάν έχει εκφράσει την επιθυμία να αντικαταστήσει τη συμφωνία σύνδεσης που προτείναμε με μια, ένα στρατηγικό θεμοτολόγιο Συνεπώς με αυτές τις χώρες ε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε φάση αναθεώρησης της πολιτικής προσαρμόζοντας την, στις περιστάσεις και στις επιθυμίες τους. Να πω τώρα όσον αφορά τα ερωτήματα του κυρίου Λόνας. Πρώτον, ναι, βοηθάμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, έχει ένα πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα η Κομισιόν το COSME, ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2,3 δισεκατομμυρίων για την επόμενη εξαετία, εκ των οποίων σημαντικό ποσό αφιερώνεται στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Αν επιθυμείτε θα σας στείλω τις λεπτομέρειες. Το ίδιο και δεύτερη σας ερώτηση. Τι κάνουμε για να βοηθήσουμε αποτελεσματικά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων και την τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων ε, για φυτογενομικά μέτρα και ασφαλεία των τροφίμων. Ναι, τους βοηθάμε. Αποτελεί κομμάτι των ε, σε βάθος ολοκληρωμένων ε, συμφωνιών για τα προϊόντα. Έχουμε πολύ ουσιαστική τεχνική αρρωγή και χαίρομαι που λέω ότι στη Γεωργία και στη Μολδαβία έχουν σημειωθεί σημαντικές πρόοδοι και το βλέπουμε ήδη για τη νέα προϊόντα ζωικής προέλευσης εξάγονται πλέον που δεν εξάγονταν παλιότερα λόγω ακριβώς ε, των προτύπων αυτών από αυτές τις περιοχές. Ευχαριστώ να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Όσον αφορά το σχόλιο του κ. Λαντσμπέργκης για τη σχέση με τη Ρωσία, πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ δύο πολύ διαφορετικών πραγμάτων. Ένα πράγμα είναι οι συνομιλίες με τη Ρωσία, που δεν αρνηθήκαμε τις συνομιλίες με τη Ρωσία όπως γνωρίζετε. Από τις 12 Σεπτεμβρίου συμφωνήθηκε να γίνουν διμερείς ε, ε, συνομιλίε με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Εμεί πρόσφατα καλέσαμε τη Ρωσία γιατί η Ρωσία παρέμεινε σιωπηλή για να αντιμετωπίσουμε και τα δικά τους προβλήματα επανεκκίνησης των συνομιλιών και αναφέραμε ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τα διάφορα ζητήματα. Φυσικά κάτι εντελώς διαφορετικό ή θα ήταν να προβλέψουμε εμπορικές διαπραγματεύσεις και ειδικότερα διαπραγματεύσεις ελευθερών συναλλαγών. Και δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω γιατί Φυσικά η Επίτροπος Μάλμστρομ το εξήγησε λεπτομερώς πώς έχει η κατάσταση. Για να ολοκληρώσω λοιπόν καλωσορίζουμε τη δεσμευσή της Επιτροπής σας κύριε Πρόεδρε και είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε εφόσον το χρειαστείτε. Ευχαριστώ. And... Ευχαριστώ. Λοιπόν, για τον Νότο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να συμπληρώσω για τις χώρες της νότιας ευρωπαϊκής γειτονίας. Ε, Όσο είπε ο Λουκάς, ε, πολλά από αυτά ισχύουν και για τον Νότο, κυρίως όσον αφορά την ευρωπαϊκή αρρωγή προς τους μικρούς γεωργούς, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να τηρούνται τα πρότυπα μας SPS για τη γεωργία, όσον αφορά την υποστήριξη της υποδομής, την υποστήριξη προς μικρομεσές επιχειρήσεις. Μια μικρή διαφορά από αυτήν την άποψη είναι ότι εμείς ως Ευρώπη έχουμε εμπορικέ σχέσεις με τις χώρες της νότιας πλευράς της Μεσογείου και συμφωνείς πολλές φορές ήδη από τη δεκαετία του 70, οπότε δεν ξεκινάμε από το μηδέν, ούτε από πρόσφατες εξελίξεις. Ουσιαστικά έχουμε ήδη αμοιβέ, αλλά μερικές φορές ασύμετρες ε, συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών με τις περισσότερους εταίρους ε, της νότια γειτονία με εξαίρεση τη Συρία και τη Λιβύη. Εστιάζονται αυτές κυρίως στη συναλλαγή αγαθών και στη διάσταση πρόσβαση στην αγορά για αυτό το σκοπό. Και απομένουν να γίνουν πολλά και έχει γίνει ήδη πολλή δουλειά με τους εταίρους μας δεδομένων φυσικά και των ικανοτήτων τους και το πόσο τους ενδιαφέρει για ενίσχυση των συμφωνιών και για την εμβάθυνση ή τη διεύρυνση των διατάξεων για, σε μη δασμολογικούς και ρυθμιστικούς τομείς. Πιθανώς εισάγοντας στοιχεία που είτε δεν έχουν συζητηθεί είτε έχουν συζητηθεί μόνο επιφανειακά όπως οι υπηρεσίες, ε, οι δημόσιες συμβάσεις, τα πνευματικά δικαιώματα. έχει ξεκινήσει μια ε, προσέξη της CFTA για, με το Μαρόκο και κάτι τέτοιο έχει προσφερθεί στην Ιορδανία, την Ισία και την Αίγυπτο. Με τις άλλες χώρες δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ατζέντα. Εργαζόμαστε περισσότερο τομεακά σε αυτούς τους τομείς. Είμαι τον ενδιάμεσο στόχο υποστήριξη τη πρόσβαση των χωρών αυτών στον ΠΟΕ, χωρών που δεν συμμετέχουν ακόμα στον ΠΟΕ. Εμείς φυσικά ως Κομισιόν ε, επιθυμούμε να συζητήσουμε ε, μαζί σας για τις διαδικασίες αυτές και να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις. Θα ρούμε ότι γενικά οι εμπορικές συμφωνίες ήταν επωφελείς, προώθησαν τις εμπορικές δραστηριότητες και τις επενδυτικέ δραστηριότητες. Αλλά φυσικά τίποτα δεν είναι τέλειο και συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να υποστηρίξουμε τους εταίρους μας στις διαδικασίες ρυθμιστικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Τους υποστηρίζουμε στις διαδικασίες ρύθμισης των αγορών τους με τρόπο πιο ευθυγραμμισμένο με τη δική μας. Και μέρος αυτού, όπως ανέφερα, είναι η υποστήριξη των εξαγωγέων, των εταιρών χωρών, ώστε να ε, αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Αγορά. Να κάνω ένα σχόλιο τώρα σε πολλούς τομείς για τους οποίους δεσμευτήκαμε να ανοίξουμε τις ε, αγορές μας όπως για τις δεσμολογικές προσθέσεις για τη γεωργία δεν συμπληρωθούν στο 100%. Ακόμη λοιπόν και αν υπάρχει αγορά, κάτι άλλο υπάρχει που εμποδίζει όπως φαίνεται την προμήθεια από τους εταίρους. Φυσικά σε όλα αυτά όπως είπε και ο Λούκα για τον Νότο, το, την Ανατολή, τη τη Δύση ευχαριστώ να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις. Μαρία, έχετε να πείτε κάτι Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Κομισιόν για τη διαθεσιμότητά της. Έχω μια ερώτηση. Στις απαντήσεις δεν άκουσα ούτε μία φορά να αναφερόμαστε στα, δικαιώματα, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη δημοκρατία. Άκουσα μόνο τη λέξη αγορά, αγορά, αγορά. Ήθελα να μου πείτε κάτι παραπάνω για τα δημοκρατικά θέματα μιλάμε για πολιτικές γειτονίες και στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών το ζήτημα της δημοκρατίας είναι ουσιώδες. Θα ήθελα λοιπόν, ίσως να ήταν λάθος μετάφραση, θα ήθελα λοιπόν αφού η Κομισιόν είναι τόσο διαθέσιμη να μπορέσει να μας πει και κάτι για τα δημοκρατικά ζητήματα. Ευχαριστώ. Ήθελα απλά να απαντήσω στον εκπρόσωπο του ECR όσον αφορά τις ε, διαφορετικές ταχύτητες ε, των διαφορών χωρών, το επίπεδο ετοιμότητας, τα διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας των διαφορών χωρών στο πλαίσιο της γειτονίας. Αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τα διαφορετικά συμφέροντα. Από τη μία έχουμε την Αρμενία, η οποία κοιτάει προς άλλη κατεύθυνση και από την άλλη έχουμε τη Γεωργία ή την Ουκρανία ή τη Μολδαβία που ε, είχαν πρόσφατα εκλογές ε, και αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο θα σώσουμε την έννοια της ανατολικής γειτονίας. Αν δούμε την κάθε χώρα, τι έχει επιτύχει και τι θέλουμε και τι μπορεί να βελτιωθεί, με αυτόν τον τρόπο θα σώσουμε το όλο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα λοιπόν- πρέπει λοιπόν... να συνδυάσουμε τις απόψεις αυτές σε σχέση με την συζήτηση στην Επιτροπή μας ώστε μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής της Ρήγας τον Μάρτιο 2015 να τα καταφέρουμε να αποσαφηνίσουμε τη θέση μας για το εμπόριο και την πολιτική γειτονία, ποιες είναι οι θέσεις μας. Και φυσικά υποστηρίζουμε και τις τάσεις αυτές που αναφέρθηκαν. Εντάξει, Ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη και περνάμε στο 14 στην ημερήσια διάταξη. Όμως να θυμόσαστε, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και ένα μικρό ποτό που θα προσφερθεί εκτός αίθουσας αμέσως μετά την λήξη της συνεδρίασης για να γιορτάσουμε κάπως την καλή δουλειά μας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή μέχρι σήμερα, μέχρι απόψε. Σημείο 14. Παρακολούθηση δραστηριοτήτων ομάδων. Έχετε συνειδητοποιήσει τις ομάδες ε, που, ε, στις οποίες συμμετέχουμε για την παρακολούθηση δραστηριοτήτων. Ερωτώ, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω πληροφορίες, πληροφόρηση για Σιγκαπούρη, David Μάρτιν, παρακαλώ. Όχι, δεν έχουμε τίποτα καινούριο να πούμε είχαμε μια συνάντηση όπως την τελευταία συνάντηση για θέματα εμπορίου με τον κύριο, τους κύριους διαπραγματευτές και ακούσαμε από τα, αν θα, μας, θα ασκήσει προσφυγή Επίτροπος Μάμστρομ σε σχέση με το θέμα της Σιγκαπούρης ή όχι. Αυτό ήταν το πιο πρόσφατο. Για την Ταϊβάν τώρα εσείς έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Είχαμε την πρώτη επίσημη συνάντηση σε σχέση με την ομάδα για παρακολούθησης για την Κίνα. Έχουμε μια νέα δομή σε σχέση με τις σχέσεις ε, με την Κίνα και την Ταϊβάν πλέον. Είχαμε την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς έχουν εξελιχθεί αυτοί οι διάλογοι με την Κίνα και η υποεξέλιξη διαπραγματεύσεις για συμφωνία επενδύσεων σχετικά και είχαμε και μια παρουσίαση εξ ονόματος του επικεφαλής της αντιπροσωπείας εμπορίου από την Κίνα στις Βρυξέλλες των συναφών θεμάτων και είχαμε επίσης το εξής που διαπιστώθηκε και η γνώμη μου επ' αυτού είναι ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να είχαμε μεγαλύτερη ταχύτητα, με ταχύτερους ρυθμούς να μπορούσαμε να προχωρήσουμε, με μεγαλύτερο σθένος να προχωρούσαμε σε σχέση με τους εταίρους μας ε, αυτές τις διαπραγματεύσεις. Επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων για τις επενδύσεις θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο μετά από τον οποίο θα έχουμε μια συνάντηση της ομάδας παρακολούθησης δραστηριοτήτων και για μια συνάντηση για τη σχέση με την Ταϊβάν επίσης. Ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστούμε. Ο Χέλμουτ τώρα παρακαλώ. Ερώτηση εσείς. Μόνο μια ερώτηση, ναι. Δυστυχώς ε, δεν μπορούσα να παρακολουθήσω την ομάδα παρακολούθησης δραστηριοτήτων. Από πλευράς των Κινέζων υπήρξαν πρόσθετες παρατηρήσεις που να έγιναν σε σχέση με την άποψη τη δική τους των Κινέζων για την πρόσβαση στην αγορά και προϊόντων και τι γίνεται σε σχέση με τη Συμφωνία Επενδύσεων. Τη δεύτερη ερώτηση, Ζαχραντήλ, εσείς παρακαλώ. Να πω δύο λόγια για την ομάδα παρακολούθησης για το Βιετνάμ. Ο κύριος Βίνκλερ. Δεν είχα αρκετή πείρα ώστε να μπορέσω να μην πω τίποτα με πολλά λόγια. Δεν έχω εξασκηθεί σε αυτό το εγχείρημα προσπαθούσαμε να διαπιστώσουμε κάποια πράγματα, δόθηκαν διασφαλίσεις των επιθυμιών των Κινέζων εταίρων, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί πρόοδος σε αυτούς τους διαλόγους, σε αυτές τις επαφές. Έδωσαν, πώς να το διατυπώσω, διασφαλίσεις για την εξέλιξη, θετική εξέλιξη των πολιτικών μας σχέσεων και με την επίσκεψη του ε, Προέδρου του στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι τα ηχέγγια η ε, εγγύηση της δέσμευσης των Κινέζων αυτή η συνιστός, αυτή η τοποθέτηση. Και ο ε, Υπουργός Ζανγκ έδωσε την δική του άποψη για μια συμφωνία για τις διμερείς επενδύσεις, θέματα διμερών επενδύσεων, ώστε να μπορέσει αυτό να ευδοκιμήσει. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία έχουμε. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε τίποτα περισσότερο. Για το ISDS δεν έχουμε κάτι να πούμε. Πολύ καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά για την Νότια Ασία, Νοτιοανατολική Ασία έχετε εσείς τον λόγο. Ευχαριστώ. Ε, είμαι τόσο καιρό εδώ που μπορώ να σας πω ότι κινδυνεύω όταν στέκομαι ανάμεσα στα μέλη που κάθονται εδώ και τα ποτά τους που βρίσκονται απ' έξω. Όταν συναντηθήκαμε 19 Νοεμβρίου ήταν απολύτως επίκαιρο διότι είχε σημειωθεί σημαντική πρόοδος μετά την τελευταία ενημέρωση που είχε λάβει χώρα 20 Οκτωβρίου. Είχαμε μια πολύ ενημερωτική και ολοκληρωμένη συζήτηση για πολλά από τα επιτεύγματα που έχουν λάβει χώρα μέχρι στιγμής και συζητήσαμε επίσης και κάποιες από τις αναπομένουσες προκλήσεις. Συνοπτικά έχει σημειωθεί τεράστια ε, πρόοδος μετά από την τελευταία συνάντηση της ε, ομάδας παρακολούθησης από τον Απρίλιο φέτος στην Νοτιοανατολική Ασία ενισχύεται ε, διάφορα δικαιώματα, έχουν δημιουργηθεί νέα συνδικάτα, περισσότερες επιθεωρήσεις ασφαλείας κτηρίων και πυρκαγιάς έχουν λάβει χώρα, Έχουμε βάση δεδομένων τώρα για τις επιθεωρήσεις εργοστασίων και υπάρχουν online, αλλά ενημερωθήκαμε ότι χρειάζονται περισσότερα μέτρα, όπως διασφάλιση αποτελεσματικής ε, εφαρμογής ε, του νόμου περί εργαζομένων του Μπαγκλαντές, μεταφορά κάποιων ρυθμίσεων του ILO και συζητώνται τώρα αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο του Μπαγκλαντές να παρέχονται σε όλους τους εργαζομένους τα ίδια δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων όσων εργαζονται στις ζώνες επεξεργασίας εξαγωγών και να διασφαλίσετε ότι όλα τα θύματα λαμβάνουν όλη την υποστήριξη που χρειάζεται για την αποκαταστασή τους. Τέθηκε επίσης το ζήτημα του κατά πόσο καταβλήθηκαν πραγματικές αποζημιώσεις από όσους ε, υπέφεραν ή τις οικογένειές τους. Έχουμε σοβαρές ανησυχίες γι' αυτό. Εξακολουθούμε να το παρακολουθούμε. Ο πρέσβης του Μπαγκλαντές ε, θα βρίσκεται στην, ε, Επιτροπή τον Ιανουάριο στην Επιτροπή ΙΝΤΑ, συγγνώμη, τον Ιανουάριο ε, και θα συμφωνείτε μαζί μου ότι χρειαζόμαστε όλοι ένα ποτό μετά από αυτή την πολύ γρήγορη παρουσίαση Ελπιδοφόρο το ότι υπάρχουν τέτοιες εξέλιξει στο Μπαγκλαντές Το λοιπόν για το Βιετνάμ ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχει ναι, μια συνάντηση μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου. Αναμένουμε πιθανώς δύο ή τρεις ακόμη συναντήσεις αν όλα πάνε καλά. Όπως ανέφερε η Επίτροπος κ. Μάλμστρομ και αν ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις το πρώτο εξάμεινο 2015 αν και ελπίζουμε στο πρώτο τρίμηνο Προγραμματίζουμε να συναντηθούμε τέλη Ιανουαρίου, διότι ο 11ος γύρος προγραμματίζεται κάπου μεταξύ 19 και 23 Ιανουαρίου. Εκεί θα δούμε πώς ε, προχωράνε τα πράγματα. Αναμένουμε επίσης την αύξηση του νέου ε, πρέσβη του Βιετνάμ στις Βρυξέλλες αρχές του επόμενου έτους, οπότε σίγουρα θα τον καλέσουμε. Ίσως όχι για τον Ιανουάριο βέβαια, για τη συνάντηση του Ιανουαρίου, αλλά για την επόμενη συνάντηση, το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ωραία. Και ο κ. Λαμπεργη για την Ουκρανία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μόλις χτες είχαμε μια πρώτη συνεδρίαση παρακολούθησης. Είμαι ιδιαίτερος ευγνώμων στους συναδέλφους της Επιτροπής που συμμετείχαν. Ένας από τους ομιλητές ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Ουκρανία, όπως επίσης και ο Ουκρανός πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα θέματα που θύσαν αφορούσαν τις πρόσφατες εκλογές και τις προοπτικές μιας ε, ατζέντα μεταρρυθμιστικής. Όλοι σχεδόν οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στις μεταρρυθμίσεις. Είναι το βασικό θέμα μετά την κατάσταση του Νοεμβρίου είναι το θέμα το βασικό με την Ουκρανία. Μία από τις σκέψεις που διατυπώθηκε στη συνάντηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει από την Ουκρανία να δείξει ξεκάθαρη πολιτική θέληση υπέρ των ε, μεταρρυθμίσεων. Το υπογραμμίζω εδώ και το υπογράμμισα και τότε ότι υφίσταται, υπάρχει αυτή η πολιτική θέληση τη δείχνουν. Αυτό που δεν είναι βέβαιο είναι αν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησής της και είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξει και αυτή η δυνατότητα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν η αναφορά της ε, παρακολούθησης των διαφόρων ομάδων. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δραστηριότητα και τώρα έχω τη χαρά να προσκαλέσω όλους ε, όσοι είναι μέσα στην αίθουσα αλλά και πίσω από τα τζάμια να έρθουν να πιούν ένα ποτό για να γιορτάσουμε το έτος της πρώτης παραγωγικής χρονιάς της συνεργασίας μας.